Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζεται η ψηφοφορία, μια τελείωτη ψηφοφορία που είχαμε χθες, και σας ευχαριστώ όλους για την αντοχή σας και την υπομονή σας, ειδικά την Εύα που άρχισε να πατάει πάρα πολύ γρήγορα τα κουμπιά, είναι δύσκολος ο μηχανισμός. Πού είχαμε φτάσει χθε το βράδυ, είχαμε ψηφίσει όλα τα στοιχεία των ε, έξι εκθέσεων. Λοιπόν, ο Ζων Πολ θέλει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, στην αρχή της συνεδριάσεως θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου τους διερμηνείς που χτε έκαναν και τη δουλειά και κυρίω είχαν την καλοσύνη να μείνουν περίπου μία ώρα μετά την κανονική λήξη των εργασιών του, τις εργασίες του Θέλω να τα πω σε αυτούς που ήταν χθε εκεί και αυτού που δεν είναι σήμερα. Ίσως μπορούν να διαβιβάσουν ε, οι συνάδελφοι το μήνυμα ότι αυτή η χειρονομία εκτιμήθηκε πάρα πολύ από τους βουλευτές και κυρίως από εκείνου που είναι οι συνηθισμένοι τους πελάτες. Ευχαριστώ ξανά του διερμηνείς. Thank Σας ευχαριστώ. Πράγματι γιατί και αυτοί έμειναν μαζί μας. Λοιπόν, Είχαμε σφίσει όλα τα στοιχεία των ε, έξι εκθέσεων. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Μπούλμαν είχε εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις και είχε ζητήσει οι επιφυλάξεις ε, που αφορούσαν τις ε, διαπραγματεύσεις για συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση να καταγραφούν στα πρακτικά. Επεσήμανα πως ως Επιτροπή πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για το εάν ε, στοχεύουμε να μπούμε σε διαπραγματεύσεις ε, για συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Ε, βεβαίως ε, είπα πως αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να τελειώσουμε και στην πρώτη ανάγνωση. Ξαρτάται ως που θα φτάσουμε, ποια θα είναι τα αποτελέσματα και πρέπει άρα να δοθεί, να δοθεί μια εντολή στην διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου για να δούμε αν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις στην πρώτη ανάγνωση. Αυτό βεβαίω πρέπει να αφορά το συνολικό πακέτο, το οποίο αποφασίσαμε πως να μείνει πακέτο και άρα η πρότασή μου είναι με τη συνήθη διαπραγματευτική ομάδα, δηλαδή πρόεδρος, ε, εισηγητές και σκιώδης εισηγητές, να ξεκινήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όπως αναφέρθηκε από τον ε, κύριο Μπούλμαν, ήδη είχαμε κανονίσει πως το απόγευμα θα είχαμε έτσι μια κάποια ανταλλαγή απόψεων παρά τύπο τριμερή διάλογο με την Προεδρία γιατί είχαν ε, την ευγένεια να έρθουν να μας εξηγήσουν πού είχαν φτάσει εκείνοι και ποια είναι η γενική τους προσέγγιση και άρα και εμείς θα έπρεπε να ανταποδώσουμε και να περάσουμε στις ε, διαπραγματεύσεις. Σε λεπτομέρειες διαπραγματεύσεις μετά τις διακοπές του Πάσχα. Αυτό λοιπόν ζητώ από την Επιτροπή να μας δώσει ως εντολή. Ο Ζαν θέλει να πει κάτι σχετικά. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι για την ομάδα του ΕΛΚ πρέπει να πω ότι συμμεριζόμαστε το όραμά σας σχετικά με αυτά που πρέπει να γίνουν. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται περί παραδόσεως στην Επιτροπή αυτή όσο θυμάμαι, δηλαδή τα τελευταία έξι χρόνια πάντα να γίνονται διαπραγματεύσεις μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή όσον αφορά τα θέματα οικονομικά και χρηματοδοτιστικά τα οποία εξετάζουμε. Αυτό έχει το όφελος σε τομείς όπου χρειάζεται μία αντίδραση σημαντική να γνωρίζουμε καλύτερα τη θέση μας, τις θέσεις μας και καταδεικνύει εμπειρία ότι αυτό επιτρέπει αποτελεσματικότητα. Όπως κάναμε και για το πακέτο της εποπτείας, Πρέπει λοιπόν μετά από μια συζήτηση με το Συμβούλιο να διακόψουμε την ψηφοφορία ώστε να μπορούμε να επανέλθουμε πρώτου Κοινοβουλίου και εν συνεχεία να μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ε, νομίζω αυτή η διαδικασία που δεν είναι πλέον συνήθις που εξαπλώνεται απέδειξε ότι είναι αποτελεσματική για τα μεγάλα θέματα που εξετάσαμε το 2010 και γι' αυτό προφανώς είμαστε υπέρ ανεπισήμων συζητήσεων που να ξεκινήσουν από σήμερα, διευκρινίζοντας όπως είπατε και ίδια ότι στόχος δεν είναι να φτάσουμε πάση θυσία σε μια συμφωνία στη πρώτη ανάγνωση, αλλά να διεξαχθεί μια λογική συζήτηση με ένα στόχο την αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση η οποία επικρατεί για τους ε, συμπολίτε μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κέι, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω κάτι. Εμείς οι συντονιστές στην αρχή της διαδικασίας πέρασαν πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρόκειτο περί πακέτου με έξι σημεία και ότι θα εμπεριείχε διαφορετικού ηγητέ από διαφορετικέ ομάδε που θα εργάζονται από κοινού, ακολουθώντα παρόμοιε γραμμέ όπω και για το πακέτο τη εποπτεία. Δοθέντω ότι αυτή ήταν η απόφαση που ελήφθη, θα απογοητεύουν τα μάλα αν υπήρχε άλλη πρόταση το πακέτο των 6 ε, να μην προχωρήσει ε, σε αυτή τη φάση, να προχωρήσουν όλα μαζί. Καταλαβαίνω την απογοήτευση που πάντα, τη απογοήτευση των ομάδων πάντα δεν πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Σαν ομάδα εμεί είμαστε στην άλλη πλευρά του ζητήματο επανειλημμένα και σεβαστήκαμε τη θέση του Κοινοβουλίου όταν ε, διεξαγόταν διαφανής ε, ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή και ακολουθήσαμε τον τριμερή διάλογο καλή την πίστη μετά. Λοιπόν, είναι η αφετηρία μιας μακράς διαδικασίας, σας προειδοποιώ δεν είναι το τέλος. Εχθές ήταν πάρα πολύ σημαντικό το βήμα, πρώτο βήμα όμως, θα πρέπει καλή την πίστη να κρατήσουμε το πακέτο έτσι ενίο και αδιέρετο, θα το εκτιμούσα. Ευχαριστώ. Ζήσε το λόγο, Ούντο, αλλά έχει πάρει το λόγο χτες. Έχεις τίποτα να προσθέσεις. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παραμείνουμε στον ουσιαστικό τόνο που συνήθως έχουμε και να υπενθυμίσω μία διαφορά. Κοιτάξτε, χθες επικρατούσε μία κάποια διάθεση και κάποιοι είχαν ε, ναι, προετοιμάσει μία δήλωση η οποία θέλει να δώσει μία έντολη, δεν ξέρω για μια, συμβασμό στην πρώτη ανάγνωση. Αυτό έχει μία σαφή προϋπόθεση και η προϋπόθεση λέγεται συνένεση στα βασκότερα σημεία. Η σημαντική διαφορά βεβαίως με το πακέτο της επίβλεψης ε, του συναδέλφου βεβαίως είναι πως εκεί πέρα υπήρχε συνένεση ενώ εδώ πέρα δεν υπάρχει γιατί οι απόψεις ε, διαφέρουν σε πάρα πολλά σημαντικά σημεία και σας παρακαλώ να μην ε, το επιρρύψετε αυτό σε εμάς, γιατί εμείς ε, πάντα λέγαμε πως θα πρέπει να συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε μέχρι να επιτευχθεί η συνένεση. Το αρνηθήκατε εσείς και άλλοι, άρα δεν είναι δική μας η ευθύνη. Απλά τώρα πρέπει να διαπιστώσουμε πως οι προϋποθέσεις για την ε, εντολή συμβιβασμού σε πρώτη ανάγνωση δεν υφίστανται. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω να γραφτεί αυτό στα πρακτικά πως οι προϋποθέσεις δηλαδή δεν υπάρχουν για ένα συμβασμό στην πρώτη ανάγνωση και πλέον θα ήθελα να ζητήσω στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών στο Στρασβούργο να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και μπρο. Αυτό νομίζω είναι το σωστότερο που μπορούμε να κάνουμε με αυτό το πακέτο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να διορθώσω αυτά που είπατε χτες ακολουθούσα την ε, κανονική διαδικασία. Τώρα, αν θέλουμε να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, ε, πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με την Επιτροπή. Παρενεύεται πριν καταφέρω να το παρουσιάσω αυτό το θέμα και ένα από τα πράγματα που είχα υπόψη μου ήταν να το αναβάλουμε μέχρι σήμερα το πρωί. Αλλά τελικά με πρόλαβες. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω το άρθρο 70 που αφορά τις διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα και λέει πριν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η, συγγνώμη, η Επιτροπή Υπεύθυνη θα πρέπει καταρχήν να λάβει απόφαση με την πλειοψηφία των μελών και θετήσει εντολή προς ανατολισμούς ή προτεραιότητε. Ήδη το κάναμε αυτό ε, μέσω της ψηφοφορίας αλλά σαν επιτροπή μπορούμε να υιοθετήσουμε την εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα ήθελα να παραπέμψω και στο παράρτημα 21 του Δεντολογικού Κώδικα για τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας και την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων, από εκεί αναφέρει σε γενικό κανόνα σε γενικό κανόνα, το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί όλε τι δυνατότητε που προσφέρονται σε όλε τι φάσει τη κανονική νομοθετική διαδικασία. Η απόφαση να ζητηθεί να επιτευχθεί συμφωνία στην αρχή, στα πρώιμα στάδια τη νομοθετική διαδικασία, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση λαμβάνοντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ξεχωριστού χαρτοφυλακίου και θα πρέπει να δικαιολογείται πολιτικό, παραδείγματο χάρη λόγω πολιτικών προτεραιοτήτων και για την μη επίμαχη ή τεχνική φύση της, ε, του θέματος κατεπίγουσα κατάσταση ή τη στάση δεδομένης προεδρίας σε συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει να πω ότι στην παρούσα κατάσταση πιστεύω ότι πρόκειται περί πολιτικής προτεραιότητας είναι κατεπήγον το θέμα, δηλαδή αν μπορούμε να καταφέρουμε συμφωνία θα βοηθήσει να εξομαλυνθούν οι δύσκολες καταστάσεις που κρατούν στην αγορά και δοθήσει στις νοτροπίες της Προεδρίας για αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι δεδειγμένο να προχωρήσουμε. Άρα δεν είναι θέμα συνένεσης όπως λέτε, αλλά είναι ένα θέμα ψηφοφορίας της πλειοψηφίας και αυτό έτσι προτίθεμε προτίθεμαι να το παρουσιάσω σε μερικά λεπτά. Σβέν, έχει συζητήσει εσύ το λόγο. Ε, είναι ατυχές διότι τώρα συζητούμε κάτι, όχι με 40 να περιμένουν, θα έπρεπε να γίνει, είναι συνεδρία που φορά τους συντονιστές κανονικά. Εκεί πάντα επιδιώκαμε την πλέον δημοκρατική λύση. Και πρέπει να πω ότι μετά από διαβουλεύσεις με την Προεδρία μας, ο συνηθισμένος κανόνας ακολουθείται Δηλαδή η συμφωνία της πρώτης ανάγνωσης είναι αυτό που επιδιώκεται αν υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή. Γιατί και υπάρχει ένα σωστό ε, δημοκρατικός λόγος, διότι οι συνάδελφοί μας στις άλλες επιτροπές δεν μπορούν να εκφραστούν επί των διαφόρων σημείων. Αυτό σημαίνει ότι τους στερούμε από το να ψηφίσουν στην Ολομέλεια των βασικών θεμάτων. Αυτό είναι ένα θέμα για την ομάδα μας όπου ακούστηκαν πολλές ανησυχίες από διάφορες ομάδες και από διάφορα μέλη που δεν είναι σε αυτή την Επιτροπή. Χτες εκφάστηκαν, μάλλον υπήρξαν πολλές ε, θέσεις που καταψηφίστηκαν, όχι με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, αλλά 60-40 και οι συνάδελφοι ε, των άλλων επιτροπών δεν μπορούν να, στη ΣΥΜΚΟ δεν μπόρεσαν να τοποθετηθούν και δεν θα μπορέσουν να εκφραστούν στην Ολομέλεια για να υπερασπιστούν τη θέση του Κοινοβουλίου ενώ του Συμβουλίου. Είναι δημοκρατικό πρόβλημα αυτό. Και θέλω αυτό να το τονίσω. Υπάρχει πίεση από τις αγορές. Συνέστημα κατεπήγοντος. Είναι πράγματι κατεπήγον, συμφωνώ το θέμα. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Για βασικό θέμα όπως αυτό, το να στερούμε τους συναδέλφους από το δικαίωμα να συγκαθορίζουν τη θέση του Κοινοβουλίου ενάντια του Συμβουλίου. Εάν περάσει αυτό μέσω της ψηφοφορίας, αναλαμβάνεται σοβαρή ευθύνη να ε, παραβείτε τις παραδόσεις του Κοινοβουλίου ότι η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση επί πολύ σημαντικών θεμάτων ε, μπορεί να είναι κάτι που αποφασίζεται μόνο με μεγάλη διαφορά, μεγάλη πλειοψηφία. Πρόεδρο, αυτό δεν ταιριάζει με τι διατάξει που διάβασα προηγουμένω. Ε, δεν ξεκινάμε μια γενική συζήτηση. Περβάνος, ε, λυπούμε, δεν σου δίνω το λόγο. Αν υπάρχει άλλος συντονιστή ο οποίο επιθυμεί να λάβει το λόγο, εφόσον μίλησαν όλοι οι υπόλοιποι. Θα ψηφίσουμε, θα έχετε τη δημοκρατική δυνατότητα. Σιλβί. Ε, απλά ήθελα να πω πως βεβαίως θα αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες ε, του ΣΒΕΝ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία. Αυτό το οποίο κάνουμε όμως τώρα είναι να ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις. Θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν είμαστε ε, έτοιμοι να τελειώσουμε γρήγορα και μπορώ να σας πω πως ε, η θέση μας δεν είναι να πούμε σήμερα πως είμαστε έτοιμοι να πάμε σε πρώτη ανάγνωση. Ξεκινήσουμε τη συζήτηση και θα δούμε και θα το ξανασυζητήσουμε Σβέν στους συντονιστές. Θα δούμε που είμαστε και αν δεν υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία θα ε, συνεχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, όπως διευκρίνησα. Επίσης, θα πρέπει βεβαίως να ενημερώνονται όχι μόνο οι συντονιστές, αλλά και η Επιτροπή μας για το πώς πηγαίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις από καιρούς καιρών. Έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε, προτείνω τώρα να ψηφίσουμε. Περβάνς, γιατί? Όχι, όχι, δεν νομίζω. Μα γιατί δεν ήσουν καν εδώ στην ψηφοφορία. Ε, Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξέρω επί βάση ποιου άρθρου του κανονισμού μα αρνείστε το λόγο. Δεν πρόκειται περί συνεδρία των συντονιστών, πρόκειται περί ολομελίας της Επιτροπής, της Οικονομικής Νομισματική Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να δίνετε το λόγο σε όλα τα μέλη. Αν θέλετε μόνο οι συντονιστέ να εκφραστούν, θα έπρεπε να συγκληθεί με συνεδρίαση των συντονιστών. Όμω δεν είναι αυτή αυτό το σχήμα εντό του οποίου συνεδριάσεω ε, και θέλω να λάβω το λόγο για αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. Θα έδινα προτεραιότητα στους συντονιστές και στους συγητές. Αλλά, περβάνς, ορίστε, μίλα πριν τον συγητή. If you're ready to open the floor and... Εάν μπορείτε να δώσετε το λόγο και στους συγητές, με τα χαράς να μιλήσω μετά από αυτούς. Αν θέλετε γενική συζήτηση. Είπατε ότι θέλετε να δώσετε το λόγο μόνο στους συντονιστές. Αυτό ήταν το θέμα που ήθελα να θέσω. Καλώς. Αφού μου δίνετε το λόγο, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ελπίζω να μην προδώσω τη σκέψη του συντονιστού των σοσιαλιστών και δημοκρατών, δεν νομίζω. Είπατε ότι εδώ υπάρχει σημείο που είναι κατεπήγον πολιτικό πώ και ότι οι αγορές περίμεναν τοποθέτησή μα. Νομίζω ότι στην οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια τώρα, η προσδοκία των αγορών είναι ο, καλύτερος, ε, ο χειρότερος δείκτης μιας καλής διακυβέρνησης. Και στο θέμα αυτό δικηβεύονται δύο πράγματα. Προφανώς το πολι... η πολιτική συζήτηση που διεξάγεται μεταξύ μα και το είδαμε στην ψηφοφορία που έλαβε η χώρα χθε το βράδυ. Δεν υπάρχει συνένεση. Και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινά διαπραγματεύσει με μια πίεση εξαιρετικά μεγάλη, όχι μόνο του Συμβουλίου, αλλά και των αγορών για μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, είναι η καλύτερη λύση για να πετύχουμε κακή συμφωνία. Και σας καλώ να εξετάσετε όπως, ε, πώς βλέπουν τις διαπραγματεύσεις τους απ' έξω. Το λέμε επί σειρά ετών ο καθένας καλείται να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει τη θέση του, την ισχύ του και στο τέλος γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση ε, που στις ε, 10 Μαρτίου όσον αφορά το θέμα των αποφάσεων στην πρώτη ανάγνωση. Διότι στις διαπραγματεύσεις υποπίεση του Συμβουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγει πάντα χάρη στις διαιρέσεις μας να υποστηρίζει πλήρως το Συμβούλιο. Εδώ έχουμε πολιτικό διακυβευόμενο και δημοκρατικό διακυβευόμενο. Εάν δεν σεβαστούμε, αν δεν γίνουν σεβαστά δικαιώματα του Κοινοβουλίου σε αυτή την κατάσταση, οι απόψει του Συμβουλίου πολιτικά και δημοκρατικά ε, που είναι αντίθετα και οι θέσει του που είναι αντίθετε με τι δικέ μα τελικά θα είναι αυτέ που θα περάσουν. Θέσει του Συμβουλίου. Πρόεδρο. Έχουμε στεναρότατε θέσει, ισχυρέ θέσει σε πολλά θέματα και έχουμε όλες τις ψήφους, έχουμε, ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η θέση σε κάθε θέμα. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα επί των οποίων διαπραγματευόμεθα που δεν είμαστε τόσο διαιρεμένοι όπως θα ήθελα να το παρουσιάσουν μερικοί. Και νομίζω ότι έχουμε δείξει όπου είμαστε διαιρεμένοι ακόμα και εκεί να έχουμε αρκετά καλό αποτέλεσμα. Ελίσα, ήθελε το λόγο. Madam Chair, I think... Κυρία Πρόεδρε, σε μια τέτοια στιγμή η βαρύτητα του ζητήματος απαιτεί σωστές αποφάσεις και το μήνυμά μου είναι σαφές. Το κοινοβούλιο είναι διχασμένο σε πολύ κέρια ζητήματα, όχι οριακά. Και νομίζω πως αυτό το οποίο επήγει είναι να έχουμε λίγη σοφροσύνη στη διαδικασία. Οπότε, παρακαλώ τους συναδέλφους να μην μας εξαναγκάσουν σε μια θέση η οποία δεν ακολουθεί τις συνήθεις διαδικασίες του Κοινοβουλίου και την αλληλεγγύη που είναι μία από τις πιο σημαντικές πηγές δύναμης ισχύως του Κοινοβουλίου. Δεν είμαστε υπό την πίεση των αγορών, είμαστε υπό μία πίεση που μπορεί να διασπάσει την Ευρωζώνη και για πολύ καιρό τις πολιτικές διαδικασίες και το μέλλον της Ένωσής μας. Δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Και πιο σημαντικό από την πιθανή πίεση των αγορών είναι το ότι έχουμε την πίεση των πολιτών μας. Και πρέπει να δούμε το τι συμβαίνει σε όλες τις χώρες με πολύ επιφυλακτικές και επικριτικές πολιτικές δυνάμεις για το, την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Πλέον αρκετά απαιτείται από εμάς τους εκπροσώπους των πολιτών να είμαστε σόφρονες. Μην σας παρακαλώ εκβιάστε τα πράγματα τώρα. Και αυτή είναι η έκκλησή μου στους συναδέλφους. Δεν κερδίζουμε τίποτα και μπορεί να χάσουμε πολλά εάν εξαναγκαστούμε σε μια διαπραγμάτευση χωρίς να έχουμε μια κοινή αντίληψη του πού θέλουμε να πάμε. Αυτά ήθελα να πω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρκους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αναρωτιέμαι πραγματικά σε ποιο σινεμά μπήκα. Νόμιζα ότι ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υπάρχει ένας κανονισμός και αποφασίζουμε με πλειοψηφία. Χτες, 4,5 ώρες, αποφασίσαμε με πλειοψηφίε. Δεν είναι δυνατόν τώρα για ένα διαδικαστικό ζήτημα να προσπαθούμε να κάνουμε τη θέση της μειοψηφία θέση της πλειοψηφίας. Είναι απαράδεκτο. Και ζητάω από τους ε, συναδέλφους ε, των ε, υπολείπων ομάδων. Θέλετε να πάμε στην Ολομέλεια. Ούτε εκεί πέρα δεν θα κερδίσετε. Αν δείτε τις πλειοψηφίες ποιες ήταν χτες, ούτε στην Ολομέλεια θα κερδίσετε. Οπότε ούτε και μέσω αυτής της διαδικασίας δεν θα έχετε πλειοψηφία. Ε, έτσι είναι η δημοκρατική διαδικασία. Καμιά φορά κανείς χάνει, καμιά φορά κανείς κερδίζει. Αν χάνει πρέπει να το αποδεχτεί το ίδιο και όταν κερδίζει. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να αποδεχτούν πώς τα πράγματα πήγαν όπως πήγαν και δεν θα αλλάξει τίποτα με το να προσπαθούμε μέσω διαδικαστικών ζητημάτων να αλλάξουμε τα πράγματα. Απομονώνεστε και έτσι και σε άλλα σημεία δεν θα υπάρχει αλληλεγγύη. Thank you. Ευχαριστώ. Ρόμπερτ, ζήτησες ε, το λόγο και αν δεν υπάρχει άλλος ε, σκιώδης συγητής ή συγητής που θέλει να μιλήσει θα κλείσει εδώ ο κατάλογος. Ε, Ρόμπερτ, μην μη συγχύζεστε, συνάδελφοι, θα είμαι, θα είμαι σύντομος. Ξέρετε πως πολιτικοί είμαστε, έχουμε χάσει και κερδίσει ψηφοφορίε ψηφοφορίες και βεβαίως σέβομαι τις αποφάσεις της ε, πλειοψηφίας και τις χτεσινές. Αλλά η μόνη καθαρή λύση θα ήταν το συντομότερο δυνατόν να πάμε με αυτό το πακέτο στην Ολομέλεια. Έτσι ώστε όλοι οι βουλευτές να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν για αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα. Και μπορεί κάλλιστα η χτεσινή πλειοψηφία να επαναληφθεί. Αλλά τότε θα είναι σαφής η δημοκρατική απόφαση ενός ερετού κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα, δυστυχώς, κάπου χωρίς διαφάνεια Κάποιοι άνθρωποι μαζεύτηκαν σε μια κλειστή αίθουσα με το Συμβούλιο, με την Κομισιόν και θα μαζευτούν και βεβαίως θα προκύψουν ζητήματα τα οποία, ε, θα προκύψουν συγχωρείτε αποτελέσματα τα οποία μπορεί να είναι αμφισβητήσιμα. Οπότε το μόνο ξεκάθαρο, το συντομότερο δυνατόν να πάμε στην Ολομέλεια και αν είστε το σίγουρος πράγματι θα περάσετε και εκεί πέρα την άποψή σας και τότε θα έχουμε και οι διαπραγματευτές μας θα έχουν από πίσω τους την ολομέλεια ολόκληρη. Ούτω, ε, αν, αν θες να διακόψεις τους δικούς σου, μίλα, ναι. Άστο. Ένα διαδικαστικό, πρόεδρε. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εδώ, τότε μέσω της έκθεσης Σβάτς να το κάνουμε να αφήσουμε η Ολομέλεια να καθορίσει την εντολή όταν θα φτάσει εκεί η έκθεση αυτή. Αυτό είναι το πιο καθαρό διαδικαστικά επί του οποίου θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Ίσως και οι συνάδελφοι των άλλων ομάδων θα μπορούσαν αυτή τη δημοκρατική πρόταση να την δεχτούν. Είδα είχε ήδη έτοιμα του Ζαν και είχαμε αυτό το θέμα για την ψηφοφορία. Ζαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα κράτησε αυτή τη συζήτηση όπω και ο Μάρκο Φέμπερ. Υπήρχε μια πλειοψηφία που εκφράστηκε στο Κοινοβούλιο. Από ό,τι γνωρίζει, στο Κοινοβούλιο δεν υπάρχει καμία υποχρέωση συνένεση. Καμιά φορά και εκλογέ μα επί όλων των ψηφοφοριών μα κατηγορούν για συνενέσει. Σήμερα υπάρχουν σαφεί ε, τοποθετήσει οι οποίε διαμορφώθηκαν μετά από πολλού μήνε διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, αν εκείνοι που ήταν εισηγητέ δεν καταλάβαιναν τι έκαναν, αυτό γίνεται ανησυχητικό και δεν πιστεύω ότι το να πάμε στην Ολομέλεια με τους ήλιους βουλευτές που μιλούν τώρα, διότι ήλοι θα μιλήσουν ότι θα αλλάξει κάτι ε, όσον αφορά τα όσα συζητήθηκαν. Μία πλειοψηφία λοιπόν καθορίστηκε χτες επί κάποιων ζητημάτων όπως είπατε κυρία Πρόεδρε αυτή η πλειοψηφία είναι πολύ μεγάλη υπάρχουν θέματα τα οποία ήδη ε, είναι αντικείμενο συνένεσης και συζητήσεις με το Συμβούλιο θα επιτρέψουν σε καλύτερο καθορισμό των περιθωρίων ελιγμών και των δυνατοτήτων που θα έχει το Κοινοβούλιο να επιβάλλει τις θέσεις του. Νομίζω ότι να καθυστερούμε τις διαδικασίες δεν θα έχει καμία συνέπεια στον αφορά την εικόνα του Κοινοβουλίου αρνητική. Ξέρετε, μιλάμε, μιλάνε πολύ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν το μόνο που λένε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι δεν μπαίνει σε διαπραγματεύσεις και δεν θα καταλήγει σε γρήγορες ε, αποφάσεις, δεν επηρεάζει την εικόνα μας. Λοιπόν, λέω να ψηφίσουμε την εντολή για τις διαπραγματεύσεις, που εν πρώτη θα είναι ανεπίσημες και μετά μπορούμε να δούμε πού θα καταλήξουν. Αλλά δεν είναι καλό να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση κι άλλο. Ζαν Πολ ζήτησε να ψηφίσουμε και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε. Βάλτε τις κάρτες σας στο μηχάνημα για την ψηφοφορία και να επενθυμίσω σε όλους σας, εάν έχετε κάτι δεν καταλάβετε, η πλειοψηφία που πέρασαμε χθε ήταν Βόρτμαν Κόλ 27 υπέρ 10 κατά, αυτή ήταν η ισορροπία των ψήφων, Φεγιό 28 υπέρ 7 κατά, Γκουλάρτ 36 υπέρ 11 κατά, Φερέρα 41 υπέρ 4 ψήφοι κατά, Χάγκλαν 38 υπέρ 5 κατά, Φόρντ 25 υπέρ 13 ψήφοι κατά, δεν θεωρώ οδήποτε αποτέλεσμα να είναι αποτέλεσμα με μικρή διαφορά, μικρή πλειοψηφία. Αυτό, πρόεδρε, το έτοιμά μου η ψηφοφορία να διεξαγόταν με, την, με τον καθορισμό από την Ολομέλεια στη, της εντολής πάει πιο πέρα από το αίτημα Γκοζές. Πρώτα λοιπόν να ψηφίσουμε το δικό μου. Καλώς. Θέλουμε να ψηφίσουμε για το κατά πόσο θα αναβληθεί το θέμα για μη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ψηφίζουμε, ξεκινάμε. Καλώς. Ένα σας εντύπωνα βγάλει την κάρτα και τρεις του ΕΛΚ επίσης να αποσυνδεθούν. Καλώς. Είναι δύο που είναι στενδεμένοι και δεν ψήφισαν. Κάντε το τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Οπότε τώρα θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία επί της διαπραγματευτικής εντολής για την έναρξη συζητήσεων με την Προεδρία. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 14 ψήφοι κατά. Οπότε θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την υπομονή σας και την ανοχή σας. Θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη όταν ανακαλύψω ποια είναι. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όσοι φεύγουν παρακαλώ με ησυχία για να συνεχίσει η συζήτηση για τα παράγωγα. Never mind, such is life. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, χάσαμε και λίγο χρόνο με τη συζήτηση, οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Βέρνερ Λάγγεν. Να σας υπενθυμίσω. Σας παρακαλώ, ε, οι συζητήσεις εκτός σας. Συνεχίζουν οι συζητήσεις, ε, συζήτηση που είχε ξεκινήσει στο Στρασβούργο. Εξακολουθώ να έχω έναν κατάλογο μιλητών. Πρώτα απ' όλα θα παρέμβει ο Βέρνερ, μετά η Swinburne. Ε, πράσινη δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει, αν θα είναι ο Σβέν ή κάποιος άλλος, αν είναι κάποιος εδώ. Αντολίν και εγώ. Εάν θέλει για κάποιος άλλος ε, τον λόγο να μου κάνει νόημα. Βέρνερ. Ε, ευχαριστώ. Η συζήτηση έπρεπε να γίνει από τις 9 μέχρι τις 9.40. Έχουν ήδη περάσει και τρία λεπτά παραπάνω. Να κάνω μια σύντομη εισαγωγή γιατί συνεχίζεται η συζήτηση όπως είπατε. Πρώτα απ' όλα, χτες μάθαμε μεταξύ άλλων από τον Γιάνσλερ που ήταν εδώ πέρα στην Επιτροπή πως ε, το Κογκρέσο θέλει να αναβάλει κατά 18 μήνες ε, την έγκριση του νόμου Ντόντ Frank, οπότε βλέπετε πως κινδυνεύει όλη η διαδικασία. Οπωσδήποτε συμφωνούμε πως δεν είναι δυνατόν όπως στην ε, Βασιλεία 2 εμείς να αποφασίσουμε τη ρύθμιση και να κοιτάνε οι Αμερικάνοι από μακριά ποια πλεονεκτήματα από αυτά θα δεχτούν και να μην ε, ακολουθήσουν ολόκληρη τη ρύθμιση. Δεύτερον, Ξέρετε πως ε, τα παράγωγα ήδη χαίρεται, ήδη από τη Γερμανία μιλάμε για πάνω από 600.000 παράγωγα μόνο τον ε, μήνα Μάρτιο, ε, πολλά από τα οποία είναι υψηλού κινδύνου, τα λεγόμενα παράγωγα knockout, τα οποία οδηγούν σε απώλεια της Τιμή τη ε, μετοχής, οπότε δεν ξέρω εάν θα έπρεπε να επιτρέπονται καν. Και τρίτη παρατήρηση, θέλω να ευχαριστήσω την γραμματεία. Η γραμματεία προσπάθησε να συμμαζέψει τις 975 τροπολογίες. Ε, την ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Έχουμε την πρώτη ε, επεξεργασία και μετά την συζήτηση θα ήθελα αμέσως μετά τις ε, διακοπές ε, του Πάσχα να συγκινούν οι συζητήσεις στο επίπεδο σκιωδών εισηγητών και μετά να περάσουμε στις συμβαστικές τροπολογίες για να μπορέσουμε να σεβαστούμε την ε, προθεσμία. Αυτές είναι οι εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή για άλλη τη δουλειά έκανε και αυτός και η ομάδα του μέχρι τώρα και ελπίζω κάπως να καταφέρει να κάνει διακοπές το Πάσχα και να συντάξει και τους συμβιβασμού συμβιβασμούς που αποτελέσουν νέο κομμάτι της δουλειάς μας. Χαίρομαι διότι παρόλο που έχουμε 977 τροπολογίες υπάρχει σημαντικός βαθμός συνένεσης μεταξύ των περισσότερων μας επί πολλών ζητημάτων και θεωρώ ότι όλοι προς την ίδια κατεύθυνση κοιτάμε αλλά έχουμε ακολουθήσει διαφορετικές προσεγγίσεις ε, θα εστιαστώ επί δύο σημείων που εξακολουθούν να φαίνονται πιο ανοιχτά από άλλα. Όσον αφορά τις μη οικονομικές εξαιρέσεις που είναι αποτέλεσμα κοινή συμφωνία στο Κοινοβούλιο ότι οι επιχειρήσει οι τελικοί χρήστες των παραγωγών θα πρέπει να, ε, να είναι στην εξαίρεση από το Central Clearing, την κεντρική καθάριση και θα πρέπει οι ζητούν ε, τι αποτελεί συνένεση αφορά τι αποτελεί προστασία hedging των βασικών επιχειρηματικών κινδύνων. Αυτό αφορά την οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων που καθορίζονται τελικά από την ΕΣΜΑ. Νομίζω ότι στου κανονισμού επίπεδου 1 ίσω θα ήταν συνετό να δώσουμε κάποιου προσανατολισμού σχετικά με το θέμα, εν μέρη, ούτω όμως, να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει καθορισμό σαφή εξαίρεση που δημιουργεί κενά και τρύπε, Άλλο ούτως ώστε οι επιχειρήσει να έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με το κόστο του και ποια είναι η νομική κατάσταση. Ποια θα είναι πιθανόν η νομική κατάσταση. θα ζητούσα τα μέλη να εξετάσουν εκ του και στην τροπολογία μου 488 για να αξιολογήσουν κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προσανατολισμό, κατάλληλο προσανατολισμών που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα η ΕΣΜΑ σαν βάση για επίσημα κριτήρια. Ε, θα ήθελα να προχωρήσω και στο θέμα της, ε, του διαχωρισμού ε, που αφορά πολλές τεχνικές λεπτομέρειες με τις οποίες ασχολήθηκαν οι βοηθοί μας. Είναι τεχνικό θέμα το segregation, ο διαχωρισμός που έχει ξεφύγει κάπως από τις τροπολογίες και χαίρομαι που πολλές τροπολογίες πολλών πολιτικών ομάδων εστιάζονται από αυτού του σημείου διότι τελικά θέλουμε οι επενδυτές να έχουν ένα επίπεδο προστασίας που απαιτείται και απαιτούν και μια ασφάλεια δικαίου και ηρεμία που συνεπάγεται κατά τέτοιο. Κατά τη διάρκεια κατάρρευσης της Lehman Brothers, οι επενδυτές που ε, μέσω λογαριασμού Lehman μπήκαν στην καθεστή δικασία δεν ήξεραν με βεβαιότητα τι συμβαίνει με τα χρήματά τους. Δεν έχασαν τα χρήματά τους, αλλά συνεχώς ήξεραν ότι κάπου βρίσκεται σε κάποιο συλλογικό καλάθι. Αλλά όχι πότε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση. Και γι' αυτό και εγώ και άλλοι υποβάλαμε μια δυνατότητα που θα έχουν οι πελάτες ε, να έχουν εντελώς ξεχωριστούς λογαριασμούς είτε με πλήρη διαχωρισμό των πελατών ή γενικών ε, λογαριασμών omnibus. Ε, δυνητική ευχέρεια θα υπάρχει διότι ίσως να συνεπάγεται μεγάλο κόστος για πολλούς εκαθαριστικούς φορείς. Ένας φορέας ήρθε και μου είπε ότι θα πρέπει περίπου να έχουν 6.000 λογαριασμού πελατών ξεχωριστού αν τελικά δοθεί εντολή για τέτοιο σύστημα. Θα πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό του μοντέλο και χρειάζεται νέα τεχνολογία και νέα συστήματα για να μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτέ οι υπηρεσίε ε, που πρέ... υπηρεσίες πρέπει να παρέχουν βεβαιότητα και ασφάλεια στους πιο προσεκτικούς επενδυτές και θα είναι έτοιμοι να πληρώσουν το κόστος αν είναι λογικό. Όμως όχι όλοι οι επενδυτές θα επιλέξουν αυτή τη ε, διαδικασία διαχωρισμού. Αν είναι υποχρεωτική διαδικασία, το συμπληρωματικό κόστο ίσως να είναι αποτρεπτικό ε, για να μπορούν οι επενδυτές να ακολουθήσουν τη διαδικασία. Οπότε θέλω να είναι δυνητικό το μέτρο και να μην είναι υποχρεωτικό το μέτρο για του πελάτες. Και τέλος, κάτι που ανέφερα σε κάποιες συζητήσεις, είναι η αγορά του ξένου συναλλάγματος. Και θα θέλαμε αυτός ο κανονισμός να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Όμως θα έλεγα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη συγκεκριμένη αυτή κατηγορία στοιχείων ενεργητικού. Προσπαθούμε καμιά φορά να διορθώσουμε προβλήματα που ήδη ίσω έχουν επιληθεί. Σίγουρα με το ξένο συνάλλαγμα ε, δεν νομίζω ότι συμπληρωθεί στο πακέτο θα μειώσουμε τον κίνδυνο του συστήματο. Οι αγορέ ξένου συναλλάγματο είναι θεμελιωδώ διαφορετικά από άλλα παράγωγα προϊόντα. Η πλειοψηφία των συμβάσεων αναφέρουν πρόσωπο με πρόσωπο ε, και υπάρχει μια δυνατότητα να χρεοκοπήσει κατά διάρκεια μια συμβάση σε μια πλευρά τη σύμβαση. Στην περίπτωση όμω των ε, ξένων αυτών συναλλαγμάτων είναι να μην υπάρχει το συνάλλαγμα από τη μια πλευρά να πληρώσει μια συγκεκριμένη ημέρα. Και εκεί είναι το πρόβλημα και ο κίνδυνο τη διευθετήσεω. Ο τομέα αναγνώρισε τον κίνδυνο αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δημιούργησε την τράπεζα CLS για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό το θέμα, θα ήθελα να ζητήσω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στι τροπολογίε 149, 247 και 347 που ζητούν οι ιδιαιτερότητε τη αγορά του ξένου συναλλάγματο να ληφθούν πλήρω υπόψη πριν προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε μια υποχρέωση εκαθάριση. Και ελπίζω ότι στο πνεύμα των εργασιών μα μέχρι τώρα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε καλά ω σκιώδη, ώστε να καταλήξουμε σε σωστή πρακτική και ανάλογη ε, ρύθμιση μέσω του κανονισμού. Ε, σε συνεννόηση με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω κάποιον εδώ από του Πρασίνου. Θέλει να πάρει το λόγο. Εν τη αυτή περιπτώσει, αν τον είναι επόμενο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Έχω υποβάλει κάποιε λίγε τροπολογίε. Ο κύριο στόχος ήταν να είμαστε συνεκτικοί με την απάντηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Είναι τέσσερι πτυχές εδώ κυρίω. Πρώτη, αναφέρεται στο να συμπεριλαμβάνονται τα μέλη των κεντρικών συμβαλωμένων μερών σε αυτή τη ρύθμιση. Είναι ένα σημαντικό θέμα πιστεύω αυτό, διότι στο τέλος τέλος θα αποτελούν μέρος της διακυβέρνησης και αυτό είναι σημαντικό στο μέλλον να μπορούν έτσι να αναλύουν τα συγκεκριμένα θέματα συμφερόντων. Δεύτερον, οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης ε, που θα είναι σταθερό και δυνατό και με επαρκής, ε, με επαρκή συστήματα διαχείρισης που θα έχει περιθώρια και ε, κεφαλαιακά δικαιώματα αλλά και περιθώρια εδώ πρόκειται για μια υποδομή, για τις υποδομές σας στην αγορά και φυσικά εδώ πρόκειται για ελάχιστο κόστος, μηδενικό κόστος αν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό είναι αναγκαίο να έχουμε μια ρύθμιση σχετικά όσον αφορά την πρόσβαση. Όχι μόνο να μην είναι αρνητική η, δια... η αντιμετώπιση, αλλά να υπάρχει διαφάνεια και επιπλέον να υπάρχει και δικαιοσύνη, να είναι δίκαιο το σύστημα. Αυτά πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα ως στοιχεία για να αποφύγουμε υπερβολικό κατακαιρματισμό όσον αφορά την ιεράρχηση των αναγκών της αγοράς υπάρχουν και, υπάρχει και μια άλλη πτυχή που είναι σημαντική. Όχι μόνο υποχρέωση να υποβάλλονται εκθέσεις, αλλά να διατηρούνται τα αναγκαία έγγραφα για να μπορούν για πέντε χρόνια να υπάρχουν τεκμήρια για το τι γίνεται. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για αυτό το θέμα, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να ελέγχουμε την λειτουργία της αγοράς. Και εν τέλει όσον αφορά την δράση της ΕΣΜΑ, θα πρέπει η ΕΣΜΑ ως υπηρεσία να διασφαλίζει ότι όλες οι αρμόδιες αρχές θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. αυτές τις πληροφορίες. Αυτό είναι αναγκαίο για τη διαφάνεια σε σχέση με αυτή τη ρύθμιση. Okay, uh, ευχαριστώ. Ο Γιούργεν παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις υπό το δικό μας πρίσμα. Το λάβαμε υπόψη εγκρίνοντας το ότι ο εισηγητής τον αριθμό των εξαιρέσεων καταρχήν τον περιόρισε σημαντικά και προσπάθησε να αποκλείσει εξαιρέσεις. Αν δει κανεί τώρα όμως τις τροπολογίες πως έχουν, που πάλι ξαναζητούν μια ολόκληρη σειρά εξαιρέσεων να υπάρξουν, για δύο αιτήματα για αυτές τις εξαιρέσεις θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα είναι το θέμα αν τα παράγωγα όσον αφορά τις ε, ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες θα πρέπει να εξαιρούνται. Αναφέρεται ότι ο κίνδυνος λέει, είναι λέει, περιορισμένος. Μπορεί ίσως αυτό να συμβαίνει, αλλά εμείς θεωρούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα των δύσκολων να υπολογιστούν κινδύνων για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή και για τα επιτόκια. Και αν δούμε τι έγινε για παράδειγμα το 1998 είχαμε ένα ρόλο που έπαιξαν αυτά τα παράγωγα όσον αφορά τα συναλλαγματικά και τις ισοτιμίες και αποτελούν και ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς. Γι' αυτό υπό το δικό μας πρίσμα δεν θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει τέτοια εξαίρεση. Θέλω να το αναφέρω αυτό, να εξαιρεθεί αυτός ο τομέας ε, δραστηριοτήτων ή να θεωρηθεί εξαίρεση από πλευρά ορισμού. Δεύτερο τομέα είναι τα συνταξιδοτικά ταμεία που θέλουν εδώ ε, κάποιοι να εξαιρεθούν και γίνεται επιχείρημα αναφέρεται για το κόστος των ταμείων. Από την άλλη πλευρά αυτά θα μείωναν κάπως ε, τα, τις συντάξεις. Αυτό μπορεί να ισχύει, όμως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπό το πρίσμα μας αυτοί οι εμπλεκόμενοι με τα συνταξιοδοτικά ταμεία ανήκουν στους μεγαλύτερους εμπλεκόμενους της αγοράς και γι' αυτό δεν είναι σκόπιμο, δεν φαίνεται να είναι λογικό να εξαιρεθούν από το clearing, την υποχρέωση συμψηφισμού και εμείς θεωρούμε ότι εδώ θα έπρεπε να αποφύγουμε μια τέτοια εξαίρεση. Μια παρατήρηση για τις ε, υπηρεσίες συμψηφισμών, clearing. Αν έτσι ρυθμιστούν όπως προτείνεται θα είναι αρκετά μεγάλες και θα είναι τουλάχιστον κάποιος κίνδυνος ε, συστημικός κίνδυνος όσον αφορά την αγορά και γι' αυτό πιστεύω στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πρέπει να είναι διαφανές το πλαίσιο αυτών. Και για μας ανήκει ότι όλες οι πράξεις στην αγορά θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες για τους ελεγκτές, να υπάρχει ένα διαφανές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνονται όλα αυτά και που θα είναι ελέγξιμο. Γι' αυτούς τους λόγους είμαστε υπέρ να είναι ή σε δημόσιο φορέα και όχι σε ιδιωτικό φορέα μια τέτοια αρχή συμψήφισμού. Μια τελευταία παρατήρηση εν τέλει. Με τον εισηγητή εντωμεταξύ έχω συζητήσει αυτό το θέμα. Ξέρω ότι δεν είναι ε, χωρίς προβλήματα και τριβές. Εμείς όμως θα επιθυμούσαμε αν το εμπόριο με τρόφιμα και ζωοτροφές να εξ, μπορούσε να εξαιρεθεί από τα παράγωγα. Δηλαδή εδώ να είχαμε μια ε, τέτοια απαγόρευση. Ο εισηγητής μου είπε ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπάρχουν σκέψεις να υπάρξει μια τέτοια πρόταση. Ίσως θα μπορούσαμε και γι' αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε ότι δεν θα είχε εδώ κάποιο νόημα στην ε, οδηγία αυτό να συμπεριληφθεί. Αυτό με, όμως ε, με κάποιο τρόπο ίσως θα μπορούσαμε αλλού να το εντάξουμε. Αυτό είναι σκόπιμο και σημαντικό ως ε, παρατήρηση, ως σημείωση. Είναι ένα σημαντικό σημείο αυτό το θέμα της κερδοσκοπίας όσον αφορά τα τρόφιμα επισητιστικά προϊόντα. Και αν παρακολουθούμε τα δημοσιεύματα του τύπου, όχι μόνο τα, του αριστερού τύπου αλλά και του αστικού τύπου, βλέπω μια ολόκληρη σειρά παρατηρητών που απαιτούν να γίνει αυτό. Αυτό θα ήθελα να πω εν κατακλείδη. Ευχαριστώ. Sven, were... Ευχαριστώ πολύ. Σβέν, ήσουν στον κατάλογο μιλητών. Τώρα που είσαι εδώ, θέλω να μιλήσει, ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να έρθω πιο νωρί, να παρέμβω πιο νωρί. Θα διαβάσω, διότι ο Πασκάλ δεν είναι εδώ και είναι σκιώδης της ομάδας μας και διαβάσω συντομία τη δήλωσή του σχετικά με το θέμα όσον αφορά την κάλυψη των παραγόγων. Μέγιστο ποσό των παραγόγων ό,τι η θα πρέπει να καλύπτεται μέσω τυποποιημένων συμβάσεων και νομίζουμε ότι τουλάχιστον 80% είναι εφικτό κατά την άποψή μας. Η υποχρέωση συμψηφισμού clearing θα πρέπει να επεκτείνεται στους δυνατόν τα, τα περισσότερα είδη συμβάσεων τύπων συμβάσεων για συμβάσεις αποτέλεσμα συναλλαγών. Αυτό ισχύει de facto. Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις ψηφισμού μόνο για αντικειμενικά εντοπισμένος προστασία hedges εμπορικών κινδύνων από μη χρηματοστικούς φορείς και όχι κατά τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει το επίπεδο προστασία το hedge, όπως το IRS 39. Περαιτέρω, θα πρέπει να υποχρεώσει κοινοποίηση όλων των συμβάσεων και των φορέων, ακόμα και σε συμβάσει που δεν υπόκεινται στο συμπληθισμό και, και τα παράγωγα ε, για μη οικονομικά. Δεν πρέπει να εφαρμόσετε κάποιο κατόφλιο και δεν χρειάζεται κοινοποίηση. Η ΕΣΜΑ λοιπόν θα πρέπει να συνδέεται μέσω των φορέων ελέγχου της ενεργειακής αγοράς, μέσω της ΕΣΑ, για να υπάρχει ε, συμμόρφωση με την εντολή, τη συγκεκριμένη. Τα OTC παράγωγα CCP και ε, ο τίτλος οδήγησε σε σύγχυση. Καταρχήν εφαρμόζεται μόνο σε παράγωγα OTC ή αν τα άρθρα CCP επίσης εφαρμόζονται όσον αφορά ε, τα παράγωγα που αποτελούν δικείμενο συναλλαγών ε, πρέπει να καλύπτονται τα πάντα όχι μόνο στα, στα κλή Αυτή είναι η, η πρόθεση στο επεξηγηματικό σημείωμα. Και δεύτερον, πληροφορίες για όλα τα παράγωγα πηγαίνουν στα καταπαιτευτευτήρια ε, παραγόγων εμπορίου και μπορούμε να συμφωνήσουμε. Οπότε ο, για τα swaps και τα forwards ο τομέας του συναλλάγματος, συναλλαγματικών δεν μπορώ, να σταματάω γιατί είναι δύσκολο να διαβάσω αυτή τη δήλωση. Δεν έχω συνηθίσει. Λοιπόν, για τα αντισυμβαλόμενα μέλη Τα CCP όλων των ειδών θα πρέπει να ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό φαίνεται να συμφωνεί λίγο πολύ με το αρχικό κείμενο. Δεύτερον, προτιμούμε να πρέπει να εφαρμόζονται για περιορισμένο αριθμό αδειών τραπεζών ε, και παρόμοιες σε κάθε κράτος Περιορισμένα τι σημαίνει, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να παράσχουν υπηρεσίες υψηφισμού. Τρίτον, ε, καμία διαλειτουργικότητα των CCPs μέχρι ότου να έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά ε, επί πενταετία. Η ΕΣΜΑ έχει αρνηθεί οι CCPs Και εκεί σε αυτό το χώρο, σε αυτό το βήμα θα πρέπει να εκφράζεται η ευρωπαϊκή άποψη. Τα CCP των χωρών θα πρέπει να πληρούν τι προδιαγραφές όπως και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να χρησιμεύσουν σαν φορείς τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η ΕΣΜΑ μετά θα πρέπει να καθορίζει ελάχιστε προδιαγραφές για απαιτήσει αποθεματικού ή εγγυήσεων και κατεπηγόντω θα πρέπει να αυξάνονται οι οι όροι αυτοί και να περιορίζονται το εμπόριο. Και τέλο, τα CCPs οι επιτροπές για το αξιολόγηση κινδύνου CCP θα πρέπει να μπορούν να έρχονται σε επαφή με εξωτερικούς συμβούλους ή επόπτες, ούτως ώστε να, εξετάζ, να αντικατοπτήσουν σωστά ο αντίκτυπος που έχουν αυτά τα παράγωγα στους εξωτερικούς φορείς. Διμερείς διευθετήσεις. Δεχόμαστε ότι όχι όλα τα νόμιμα παράγωγα μπορεί να υποστούν την αναγκαία τυποποίηση για να περάσουν CCP. Οι απαιτήσει για εγγυήσει μεταξύ μερών και, αναγκέ και απαιτήσει κεφαλαίου θα πρέπει καταρχάς να εξασφαλίζουν ότι το κόστος αντιμετώπισης του κινδύνου θα είναι υψηλότερο από ό,τι αν χρησιμοποιούσαν CCP και δεύτερον θα πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση με την αναβάθμιση της οδηγίας που καλύπτει τις κεφαλουχικές απαιτήσει τραπεζών για τον κίνδυνο των συμβαλωμένων μέρων. Όσον αφορά λοιπόν τα trade repositories θα πρέπει να καταγράφουν τα πάντα, ακόμα και περίπλοκα μη τυποποιημένα παράγωγα θα πρέπει να καταχωρούνται αρκετά λεπτομερώς, ώστε οι υποπτικές αρχές να μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με το στόχο τους και το κίνδυνο. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να είναι επιλεκτική δυνατότητα υποβολής αναφορών στου υποπτικούς φορείς, αντί στα trade repositories. Και τρίτον, θα πρέπει να είναι προσβάσιμα αν ευκαθυστερήσουν από όλου του αρμόδιου φορεί. Και τρίτον, για τρίτε χώρε, πρώτα απ' όλα Αυστηρή, δύσκολο να διαβάσω στα αγγλικά, αυστηρή αμοιβαιότης της διευθέτησης των CCP και στα γερμανικά διατύπωση είναι παράξενη, της ρύθμισης των CCP και των trade repositories φαίνεται κάτι ανέφικτο νομικά. Δεύτερον, συνένεση όσον αφορά την ισοδυναμία ενεργής συνεργασίας ε, εποπτικών αρχών τρίτων χωρών με την ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Πασκάλ προσβλέπει στην καλή συνεργασία που ήδη ξεκίνησε και συνεχίζεται με τους ε, σκιώδεις και με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίος ομιλητής είμαι εγώ. Και μετά θα δώσω το λόγο ξανά στον Βέρνερ. Ε, δεν θα διατρέξω όλα όσα είπα και πριν. Δεν θα τα επαναλάβω, τα έχετε ξανακούσει και δεν έχω αλλάξει άποψη. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι να συζητήσουμε κάποιους τομείς όπου μάλλον έχει προχωρήσει κάπως συζήτηση. Είναι ενδιαφέρον, όλοι έχουμε λογικές ιδέες, αλλά δυστυχώς ε, δεν μπορούν να είναι όλοι, όλες στο ίδιο πακέτο. Ίσως κάτι ακραίο να είναι να κάνουμε αυτό το οποίο είπε ο Γιώργεν, τα CCP να είναι υπηρεσία κοινή ωφέλεια. Αλλά φαίνεται πως έχουμε ένα μοντέλο στο οποίο δεν είναι τα κεντρικά αυτά μητρώα συναλλαγών. Οπότε θα έχουμε μια ευρυδική κατάσταση, δηλαδή θα έχουν όλο τον ηθικό κίνδυνο τον ε, ΔΕΚΟ, αλλά σε ιδιωτικά χέρια. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην καταλήξουμε εκεί τελικά. Όσον αφορά το τι θα πρέπει να πάει στον συμψηφισμό αυτόν και το θέμα της διαφάνειας Συζητήσαμε και πριν πως ε, εάν ε, αυτό το οποίο αναμένουμε τα OTC τυποποιηθούν και καταλήξουν σε χρηματιστήρια, δεν θα μείνουν και πολλά πράγματα για να καλύπτει η οδηγία. Και αυτό δεν είναι σωστό. Ε, το μισό πρόβλημα νομίζω λύνεται και εδώ πέρα νομίζω συμφωνούμε λέγοντας πως τα πάντα θα πρέπει να αναφέρονται γιατί πρέπει να ξέρουμε ενώ να, να αναφέρονται σε κάποια αποθετήρια ε, γιατί μετά φτάνουμε στη συζήτηση που λέμε το οριζόντιο ή το κάθετο. Εγώ δεν θέλω να είναι ή το ένα ή το άλλο τα πράγματα, εγώ θέλω να είναι τρισδιάστατα. Πρέπει να μπορούμε να πάμε πάνω κάτω, αριστερά και δεξιά και διαγωνίως. Δηλαδή να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως απαγορεύουμε το να έχουμε διασυνδεδεμένα αποθετήρια και χρηματιστήρια, αρκεί να μην γίνεται αυτό με τρόπο αντιανταγωνιστικό και επηρεάζονται έτσι οι τιμές και οι ευρωπαϊκές αγορές. Αυτή είναι η άποψή μου για το που πρέπει να καταλήξουμε και νομίζω πως είναι ένα όραμα στο οποίο θα ήθελαν να καταλήξουν τελικά και οι ΙΠΑ σύμφωνα με την ομοθεσία Ντόντ Φρανκ αλλά όπως ε, είπε και ο συνάδελφος, πράγματι δεν ε, έχουν ακόμα καταλήξει για τα συμβόλαια μελλοντική ε, εκπλήρωση. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε ένα τρισδιάστατο τελικά, όπως το χαρακτήρισα, μέλλον, να δούμε το τι θα γίνει. μπορούμε να έχουμε τελικά κάποια χρηματιστήρια. Τώρα, για το θέμα αυτών των συλλογικών σωμάτων. Εγώ θέλω να υπάρχει μια σαφής διαδικασία λήψης αποφάσεων, οπότε θα συμφωνούσαμε την πρόταση του εισηγητή να δούμε και άλλες ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες, αλλά φοβάμαι πως δεν μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο θα δυσκολέψει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πάλι για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, όταν ε, είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον Γκάρι Γκένσλερ, Φαίνεται πως αυτό το οποίο ζητούσαμε ήταν ένα είδος εγγύησης ε, που ήμασταν διατεθειμένοι να αποδεχτούμε στην Ευρώπη και ήταν ζήτημα για εμάς αλλά όχι ε, για το νομοθεσία Dodd Franks ε, στις ΗΠΑ γιατί δέχονταν πολύ περισσότερα πράγματα για εγγύησης και κάποιες από αυτές ίσως να μην ήταν τόσο στίβαρες. Οπότε είπαμε πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να το εξετάζουμε το θέμα γιατί είναι σοβαρό. Δεν μπορεί να έχουμε ε, κάτι τόσο ακριβό να επιβαρύνει τα συνταξιοδοτικά ταμεία όταν πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να χρηματοδοτήσουμε αυτό το, το μέλλον. Τέλος, για τα χρηματιστήρια συμφωνώ με αυτό το οποίο υπόθηκε ήδη, δηλαδή το να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε συμψηφισμό αντί να περάσουν όλοι στο CLS, νομίζω πως θα είναι λάθος. θα πρέπει να περάσουμε ε, τα πάντα νομίζω στην πλευρά του, του συμψηφισμού και να λύσουμε εκεί πέρα το, το ζήτημα για τις συναλλαγές Intergroup. Εγώ αρχικά είχα πει και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πως θα πρέπει να εξαιρούνται. Οπότε Μετά είδα και τις δικές μου τροπολογίες και είπα πως θα πρέπει να είναι κάπως ανοιχτό και να είναι κάπως πολύ ανοιχτό και θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διμερείς ε, ρυθμίσεις. Αλλά δεν ξέρω αν και αυτό μας εξασφαλίζει πλήρως. Πρέπει να γίνουν ακόμα κάποια πράγματα για να δούμε το τι πρέπει. θα γίνει εκεί πέρα. Το άλλο ζήτημα το οποίο δεν έχουμε οπωσδήποτε αντιμετωπίσει είναι το θέμα των ομίλων. Ομίλων εταιριών. Για να μην ε, υπάρχει δηλαδή χρήση της εξαίρεσης του τελικού χρήστη εντός ομίλων εταιριών. Δηλαδή ίσως μπορούμε να δανειστούμε κάτι από αυτά τα οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή για τους ομίλους εταιριών που ξαφνικά συνειδητοποιώ πως μπορεί να γίνεται ίσως οπότε ίσως κάνω κάποιες περιττέρω προτάσεις οπότε συμφωνώ πλήρως τέλος πως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ και να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την κατάσταση. Οπότε επανέρχομαι εδώ πέρα στο σημείο από το οποίο άρχισα που πάλι στις, στην ανταλλαγή απόψεων με τον Κάρι Γκένσλερ είπαμε πως εάν έχουμε κάτι το οποίο είναι πολύ καθορισμένο στα λεγόμενα κάθετα σύλλο και δεν ταιριάζει με τον Ντόντ Φρανκ μπορεί αυτό να εμποδίσει κάποιες από τις ρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά βεβαίως την ισοδυναμία με αυτά τα οποία ισχύουν στη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα βεβαίως πολλά. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά ζητήματα. Και πρέπει να τα σκεφτούμε λίγο ακόμα. Βέρνερ, έχει το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις που και με τις τροπολογίες μπορούμε να δούμε τι θέλουν να πούνε. Και με τον συνάδελφο Σουίνμπορ να αρχίσω. 488. Δίνει λεπτομέρειες για τους ισολογισμούς ε, γενικά. Τι θα καθορίσουμε στο επίπεδο 1, level 1 και τι θα αφήσουμε στο επίπεδο 2, level 2. Πιστεύω ότι μια ολόκληρη σειρά θεμάτων στο πρώτο επίπεδο νομοθετικά μπορούν να ρυθμιστούν χωρίς να καθαρίζονται λεπτομέρειες για τους εθνικούς νομοθέτες. Είναι σημαντικό το Financial Stability Board, λαμβάνοντας υπόψη και τη Βασιλεία στις 15 Απριλίου, μια έκθεση προόδου για τις ε, αγορές παραγόγων OTC ε, έχει ε, προταθεί και αναφέρεται ότι στην επόμενη έκθεση προόδου Οκτωβρίου 2011 θα έχουμε κυρίως λεπτομέρειες για την υλοποίηση των διαφορετικών κατηγοριών παραγόγων που θα προταθούν επιτόκια όσον αφορά τα παράγωγα, ε, τις, ε, τα αγαθά και τα συναλλαγματικά. Αρκετά θέματα τα οποία αναφέρθηκαν πιο πριν σε σχέση με παράγωγα από τους συναδέλφους. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα αυτά τα θέματα, μέχρι σήμερα, στην πρόταση κανονισμού για την ΕΣΜΑ θα πρέπει να ενταχθούν και από την Επιτροπή θα πρέπει να εγκριθούν μέχρι μέσα 2012, ώστε αν είναι δυνατόν αυτή η συγκεκριμένη πρόταση σε μια ιστερότερη φάση των διαπραγματεύσεων να μπορέσει να ενταχθεί. Μέχρι τότε δεν θα έχουμε καθοριστική γνωμοδότηση από πλευράς μας που θα έχουμε δώσει. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι έκανε. Εχθές περαιτέρω προτάσεις ε, υπέβαλε που δεν αντανακλώνται ακριβώς έτσι στις τροπολογίες των συναδέλφων. Θέλει με τις αρμοδιότητες ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην αγορά για το ένα ή άλλο θέμα να διαβουλεύεται. Το θεωρώ λογικό και σκόπιμο αυτό το αίτημα και στις ε, προτινόμενες τροπολογίες πρέπει να λάβουμε αυτή την πτυχή υπόψη, χωρίς όμως αρνητικά να έχει αυτό επίπτωση στις χώρες μη ζώνης ευρώ. Και όσον αφορά την τρισδιάστατη ε, προσέγγιση, συνάδελφε πρόεδρε Sharon Bowles, με βάση τις τροπολογίες πρέπει ακριβώς να εξετάσουμε να δούμε τι γίνεται. Νομίζω συμφωνούμε αν ακούω τις παρατηρήσεις σωστά ότι λίγες εξαιρέσεις πρέπει να υπάρξουν όσον αφορά την, το γενικό πεδίο εφαρμογής. Εξαιρέσεις όσον αφορά και τις υποχρεώσεις συμψηφισμού, clearing. Για τις υποχρεώσεις καταχώρησης καταγραφής συμφωνώ απόλυτα. Όλα πρέπει να καταγράφονται και να καταχωρούνται. Για τις υποχρεώσεις όμως ε, όσον αφορά το συμψηφισμό με τους τελικούς χρήστες, ε, end users και κάποια άλλα ξεχωριστά πρέπει να δούμε. Και ε, υπάρχει ανάγκη να συζητηθούν ακόμα και τα θέματα των συνταξιοδοτικών ταμείων που έχουμε σε κάποιες χώρες, ε, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία κυρίως, μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία που κατά κανόνα δεν κερδοσκοπούν αλλά σκοπεύουν στο να κατοχυρώσουν, να διασφαλίσουν τις ε, μακροπρόθεσμες, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα. Και το hedging εδώ είναι το ερώτημα σε ποιο βαθμό διμερές clearing, διμερής ε, συμψηφισμός θα μπορεί να επιτρέπεται. Δεν έχω τελεσίδικη απάντηση. Με τις διαβουλεύσεις όσον αφορά τους συγητές και τους σκιώδεις συγητές πρέπει να υπάρξουν. Θα υπάρξουν προτάσεις τι θα γίνει με αυτά τα συνταξιδοτικά ταμεία. Είναι ένα από τα επίμαχα δύσκολα θέματα αυτό. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι δεν παρεκκλίνουν τόσο πολύ οι απόψει μα, δεν διαφωνούμε τόσο πολύ. Και από πλευρά συναδέλφου ούτε προαναφέρθηκε ότι το εμπόριο με τα επισητιστικά προϊόντα, τρόφιμα, ζωοτροφέ κτλ. Έχει ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει ξεχωριστό κανονισμό που θα υποβληθεί από πλευρά τη μία αναφορά στι αιτιολογικές σκέψεις θα μπορούσε να θεωρηθεί πιθανή, αλλά η πλήρης ένταξη σε αυτή την πρόταση δεν είναι σκόπιμο να γίνει, μια και η ξεχωριστή ρύθμιση έχει προαναγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ θερμά και από τις 2 Μαΐου θα υπάρξουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις για να υπάρξει ή δυνατόν στενός ε, ε, συντονισμός και να μην έχουμε κάποια ε, πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν σε μειοψηφίες και πλειοψηφίες με διαφορετικές έντονες απόψεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Λέει εδώ ότι αν είναι δυνατόν στην Επιτροπή μέχρι τις 24 Μαΐου και λέει 20 ενδεκάτου στην Ολομέλεια. Έχουμε λοιπόν χρόνο κάποτε εφέτος θα γίνει αυτό. Ευχαριστούμε όλους λοιπόν και τώρα περνάμε στη συνέχεια στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, σημείο 10. Ποιο είναι αυτό, είναι τα σχέδια κατοχύρωσης ε, καταθέσεων, εγγύσεων καταθέσεων. Και έχουμε και το θέμα της εξέτασης των τροπολογιών. Θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής ε, Πέτας Δήμων. Πιέζει ο χρόνος επειδή είχαμε τα προηγούμενα θέματα που έπρεπε να ρυθμίσουμε για το six pack. Αν κάποιοι μπορούν να είναι συντομότεροι θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Παρακαλώ. Ο κύριος Σίμων, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα έλεγα σήμερα νομίζω μέσα σε ένα ε, λογικό πλαίσιο χρονικό μπορούμε να τήρησουμε τα πράγματα όπως και με τις τροπολογίες 215 τροπολογίες που ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που τις κατέθεσαν ιδιαίτερα επειδή πολλές από αυτές τις τροπολογίες τις τοποθετήσεις της δικής μου έκθεσης και τις απόψεις τις υποστηρίζουν και σκόπιμα τις συμπληρώνουν εν μέρη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά καταρχήν και πρώτα να επισημάνω ότι υπάρχει πολλές, σε πολλές πλευρές συνένεση για την βάση όσον αφορά τον εξοπλισμό αυτών των ταμείων και όχι όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε την βάση για τις ε, ε, προϋποθέσεις επιστροφής. Επίσης, ε, συνένεση βρέθηκε για το θέμα ποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σχέση με καταθέσεις ε, θα πρέπει να ισχύουν για την προστασία αυτών των καταθέσεων. Εδώ ιδιαίτερα και όσον αφορά τις μικρές ε, αρχές δήμων κοινοτήτων που εδώ ε, θεωρείται ότι πρέπει να μπορούν να προστατεύονται και λόγω του ορισμού των ε, ε, προϋποθέσεων στις περαιτέρω συζητήσεις ε, σίγουρα πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε ένα σωστό συμβιβασμό. Επίσης και προς την κατεύθυνση της έκθεσης μου κάποιες τροπολογίες για την προστασία υπηρεσιών, ασφαλιστικών υπηρεσιών, επίσης και όσον αφορά και τις πωλήσει ακινήτων. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για πιο χρονικό διάστημα αυτά πάνω από το όριο των 100.000 ευρώ που αναγνωρίζεται ως όριο προστασίας κατά πόσο μπορούμε να υπερβούμε αυτό το όριο. Αλλά και εδώ πιστεύω στη συζήτηση μπορούμε να καταλήξουμε σε μια σωστή ρύθμιση και συμφωνία. Εξίσου παρομοίως και προς την κατεύθυνση των δικών μου θέσεων στην έκθεση υπάρχουν κάποιες τροπολογίες όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου της εποπτείας. Εδώ ιδιαίτερα κάποιες προτάσεις όσον αφορά την επανεξέταση του προτύπου λειτουργίας των, των πιστο, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να υπάρχει η βάση των ε, αξιόπιστων ε, πράξεων. Και εδώ πρέπει να μπορέσουμε να συζητήσουμε, αλλά και εδώ πιστεύω πάλι ότι μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία. Επίσης εξίσου στη συνέχεια θετικά ενισχύονται κάποιες, ενισχύουν κάποιες τροπολογίες τις προτάσεις που έχουμε στην έκθεσή μου, στο σχέδιο έκθεσής μου, αιτήματα για μια ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού μηχανισμού, ιδιαίτερα μια ενισχυμένη δε ένταξη της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και της ε, ΕΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για την νέα, το νέο αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων <clears throat> άσχετα από τις προτάσεις που εμείς θα, διατυπώσουμε για αυτά τα θέματα εδώ και την έκθεση Φερέρα και όσον αφορά το 2010. Νομίζω υπάρχει σωστή συμπλήρωση που εδώ θα μπορούσαμε να ε, υιοθετήσουμε. Σίγουρα υπάρχουν στι τροπολογίε κάποιε πολύ ενδιαφέρουσε αποσαφηνήσει. Για παράδειγμα, στον ορισμό, στην έννοια των καταθέσεων και των όρων και προποθέσεων, Τι εμείς θεωρούμε ότι εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο και τι όχι. Και εξίσου μια διαπίστωση του συναδέλφου Jean-Paul Gauzès που μπορεί ως διευκρίνηση να βοηθήσει. Δηλαδή ότι μια υποχρέωση καταβολής ποσών υπάρχει μόνο τότε όταν βρίσκονται τα ποσά αυτά κάτω από το όριο των ε, οριακών αυτών στόχων. Αυτό ήδη στην, ε, το, στο σχέδιο έκθεσης ε, εμπεριείχε Αυτή η αποσαφήνιση όμως οδηγεί στο να αποφύγουμε κάθε παρανόηση και κάθε παρερμηνία και νομίζω ότι είναι συμβατή απόλυτα με τη στοιχεία της δικής μου, του δικού μου σχεδίου έκθεσης. Το ίδιο ισχύει για το ποιο νόμισμα, σε ποιο νόμισμα θα πρέπει ο καταθέτης να αποζημιώνεται, σε ευρώ ή στα νομίσματα κράτους μέλους, στο νόμισμα κράτους μέλους ε, που ε, χρησιμοποιείται το νόμισμα αυτό για τις ε, δοσοληψίες των τραπεζών εκεί. Υπάρχει και κάποια όμως παρέκκληση ε, απόψεων και που πρέπει εδώ με κριτικό πνεύμα να συζητήσουμε. Το ένα είναι το θέμα του ύψους ε, του τελικού ποσού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1,5% έχει προτείνει σε σχέση με τα, τις καταθέσεις, ε, το συνολικό όριο των καταθέσεων. Εδώ είναι το μεταξύ, και το είπα αυτό πιο πριν, στην κάλυψη αυτών των καταθέσεων στην, στην, στην εγγύηση καταλήξαμε, το ύψος δηλαδή αυτό αυτόματα ε, μπορώ να πω ότι έτσι μειώνεται. Όμως τώρα έχουμε κάποιες τροπολογίες που στοχεύουν σε μια κατεύθυνση να πάμε στο 1,0% να μειωθεί ακόμα περισσότερο δηλαδή αυτό το επίπεδο. Σημαντικό εδώ είναι αφενός να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα ε, λογικό, εύλογο επίπεδο προστασίας των καταθετών να μπορεί να βασίζεται και να είναι αξιόπιστο αυτό και μάλιστα προς ε, όφελος ε, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να μην χρειάζεται ένα κράτος να παρεμβαίνει παρά μόνο σε περίοδο, περίπτωση απόλυτης ανάγκης. Από την άλλη πλευρά, σαφώς τα συμφέροντα όσον αφορά τις τράπεζες σε δεν τα έχουμε σε σχέση με τις, ε, τα τέλη των τραπεζών όσον αφορά τη Συμφωνία Βασιλείας. Δεν τα έχουμε αφήσει να φτάσουν σε υψηλό υπερβολικό επίπεδο. Εδώ όμως αξίζει αυτό το θέμα να το συνεχίσουμε να το εξετάζουμε. Ας πάρουμε το 1,5% ως στόχο. Ας δώσουμε περισσότερο χρόνο στις τράπεζες όμως να πετύχουν αυτή την κατεύθυνση, αυτό το όριο, ώστε η επιβάρηση των τραπεζών ετήσια γραμμικά να παραμείνει η ίδια τελικά σε σχέση με αυτή την πρόταση. Δηλαδή, σε εξειδικευμένα το 1,5% σε 15 χρόνια να, το, να μπορέσουμε να το συλλέξουμε και όχι σε 10 χρόνια. Η μεγαλύτερη περίοδος θα έχει επίπεδο ασφάλειας που θα διασφαλίζεται χωρίς να είναι υπερβολική επιβάρηση των τραπεζών όσον αφορά την επιβάρηση με 1% επί 10 χρόνια των τραπεζών να καταλήγαμε σε ένα 15 ε, διάστημα. Σημαντικό είναι το θέμα αρχής. Θέλουμε τώρα μια εξάντε χρηματοδότηση εκ προημίου, εκ των προτέρων ή εξ πόστο, εκ των υστέρων χρηματοδότηση. Εδώ από τους συναδέλφους ε, του Ηνωμένου Βασιλείου είχαμε κάποιες τροπολογίες που στοχεύουν στο να έχουμε εξ πόστο, εκ των υστέρων συστήματα κάλυψης. Όπως ε, καθορίζεται από την έκθεσή μου, μια τέτοια πρόταση με ιδιαίτερα κριτικό πνεύμα την αντιμετωπίζω. Εδώ θα είχαμε κυκλική επίπτωση ε, που θα ευνοούσαμε στις κρίσεις σε κρίση θα πρέπει κονδύλια από τις τράπεζες να ε, Νομίζω σκόπιμο είναι στις ε, καλές περιόδους αντικυκλικά από τις τράπεζες ε, να αντλείται ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα ε, εκραίει σε αυτό το ταμείο και αν χρειαστεί σε περίοδο κρίσης να αντλούνται από αυτό το ταμείο τα ποσά και όχι οι τράπεζες να επιβαρύνονται επιπλέον με επιπλέον επιβαρύνσεις. Επιπλέον για τις τράπεζες είναι σκόπιμο όσον αφορά την προβλεψιμότητα σχεδιασμού να καταλήξουμε σε ένα ε, πλαίσιο ασφάλειας, να γνωρίζουν οι τράπεζες τι πρόκειται να γίνει και να μην εκπλήσονται μετά όταν έχουν μπροστά τους κάποιους κανονισμούς ε, για κρίσεις που δεν θα εμπεριέχουν το στοιχείο του σχεδιασμού ή του προγραμματισμού προηγούμενα. Εξίσου επίμαχο όσον αφορά τη δική μου πρόταση αλλά και την πρόταση της Επιτροπής είναι η ιδέα να έχουμε ένα καθαρό pay box, ένα καθαρό ταμείο θα έλεγα για ε, καταβολή αυτών των ποσών. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα πρακτική σε πολλές χώρες ήδη όπου έχουμε πρόληψης μέτρα, προληπτικά μέτρα και μέτρα διάσωσης που ε, έχουν προγραμματιστεί για τη διάσωση τραπεζών και μέσω των συστημάτων κατοχήρωσης καταθέσεων, διασφάλισης καταθέσεων, ούτε λαμβάνει υπόψη επίσης το ότι αυτά τα ταμεία θα μπορούσαν πολύ πιο αποτελεσματικά να χρησιμοποιούνται το σκέλος της πρόληψης με κάτι τέτοιο στο τέλος θα παρακολιόταν και τίθεται το ε, θέμα του να δούμε αν θα ήταν ευνοϊκότερο με τέτοιο τρόπο να διασφαλίζουμε καταθέσεις. Εδώ δεν ε, θα μπορούσαμε καθόλου να καταλήξουμε σε μια τέτοια περίπτωση ε, καταβολής ποσών. Πόσο επίμαχο είναι αυτό το θέμα το βλέπει κανείς με τις τροπολογίες που στοχεύουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Όχι μόνο λένε ότι θέλουμε ένα καθαρό ταμείο box, αλλά θέλουμε σε σχέση με τη χρηματοδότηση ε, μέτρων που θα ε, γίνονται, αλλά στο ύψος ε, των συνολικών ποσών χωρίς οποιουσδήποτε παράλληλους όρους ή προϋποθέσεις. Το αντίστοιχο δηλαδή ακραίο για την καθαρή πρόταση Paybox. Αυτά είναι ακραίες θέσεις όμως. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αφενός η ελαστικότητα θα διασφαλίζεται, μέτρα πρόληψης να μπορούν να υιοθετηθούν και να λειτουργήσουν, μέτρα διάσωσης να είναι εφικτό να υιοθετηθούν, αλλά στο τέλος τέλος θα πρέπει αν έχουμε μια τέτοια περίπτωση, αν καταλήξουμε στην κατάθεση, στην καταβολή αυτών των ποσών, να μην αδειάσει αυτό το ταμείο και δεν μείνει πια τίποτα σε αυτό. Γι' αυτό στους προσδιορισμούς που κάνουμε καθορίζουμε τα πράγματα ότι τα κονδύλια των ταμείων θα πρέπει και να προβλέπετε στο ε, ολικό ύψος των δύο τρίτων των ολικών κονδυλίων να μπορούν να λειτουργήσουν για τέτοιου είδους μέτρα παρεμβατικά. Χωρίς ε, να υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνο ότι στο τέλο τέλο θα αδειάσει ένα τέτοιο ταμείο και δεν θα υπάρχουν πλέον κονδύλια ώστε σε περίπτωση κρίση ε, να ε, γίνονται οι πληρωμέ. Υπενθυμίζω την, πρώτη, την ρύθμιση ότι θα πρέπει μέχρι τα δύο τρίτα να μπορούν να λειτουργήσουν τέτοια μέτρα και να παραμείνει ένα περιθώριο ασφάλειας. Πρέπει να μείνουμε σε ένα συμβιβασμό μεταξύ του καθαρού paybox και της πλήρους χρήσης των κονδυλίων χωρίς να είναι δυνατό να αδειάσει το Ταμείο. Αυτό χρειάζεται να συζητηθεί παράλληλα με κάποια άλλα σημεία όπως για το θέμα του πώς θα διαμορφωθούν τα κονδύλια εκείνα που θα πρέπει να καταβάλλονται στο Ταμείο. Εδώ υποβάλλεται η πρόταση όχι μόνο ε, μετρητά να γίνονται δεκτά, αλλά και μια συνδρομή μέσω ενεχειριασμού ε, ενεργών ε, ποσών, δηλαδή κεφαλαίων. Και εδώ θα πρέπει και αυτό να συζητηθεί, όπως επίσης και το θέμα του προσδιορισμού των περιόδων ή των διοριών για την καταβολή. Εδώ έχουμε και σχετικά αιτήματα. Υπό το δικό μου πρίσμα δεν θα ήθελα να έχουμε μια υπερβολικά μεγάλη προθεσμία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έναν πολίτη, απλό πολίτη να ε, κυκλοφορεί 20 ολόκληρες ε, μέρες χωρίς να έχει ε, μετρητά στη διάθεσή του. Από την άλλη πλευρά κατανοώ απόλυτα ότι τα σημερινά συστήματα δεν είναι σε θέση μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες ή σε μια εβδομάδα, σε 7 ημέρες με άλλα λόγια να καταλήγουν σε τέτοιες πληρωμές. Μια και εδώ μια κέρια προϋπόθεση, θεμελιώδης προϋπόθεση θα ήταν ε, σε σχέση με τις ε, ε, εγγυημένες καταθέσεις θα ήταν μια ρύθμιση που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στα κράτη-μέλη. Εδώ πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό πιστεύω. Στο δικό μου σχέδιο έχω υποβάλει μια αντίστοιχη πρόταση. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω ποια είναι αυτή η πρόταση. Ας επανέλθουμε, ας αφήσουμε τις πέντε μέρες να λειτουργήσουν ως διορία. Αλλά συστήματα που δεν είναι σε θέση σήμερα να το κάνουν αυτό, να έχουν μια μεταβατική περίοδο στη διάθεσή τους, μόνο σε περίοδο σε διορία 20 ημερών να καταβάλουν αυτά τα ποσά. Υπό την προϋπόθεση ότι στις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες ένα ανώτατο ποσό 5.000 ευρώ, ευρώ θα καταβάλουν χωρίς ε, περαιτέρω εξέταση ad hoc ε, προς τους πελάτες τους αυτό με πολύ μικρή επιβάρηση, ας το πω έτσι, γραφειοκρατική ε, μπορεί να διασφαλιστεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και έτσι διασφαλίζει ότι οι καταθέτες αφενός ταχύτερα μπορούν να έχουν χρήματα ρευστά μετρητά στην τσέπη τους, από την άλλη πλευρά όμως οδηγεί στο να αποφύγουμε εδώ οι τράπεζες ε, να υποστούν υπερβολικές επιβαρύνσεις ε, και μάλιστα σε μια διορία που σε αυτή τη χρονική περίοδο δεν θα ήταν ε, εφικτή, δεν θα ήταν λειτουργική. Ένα επιπλέον σημείο για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι και πρέπει ανοιχτά να το συζητήσουμε είναι το θέμα του υπολογισμού, υπολογισμού των εισφορών, των τελών. Εδώ πολλές τροπολογίε καταδεικνύουν το ότι δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πρότυπό τη όσον αφορά το ε, spread των κινδύνων ε, την διασπορά κινδύνων και τον υπολογισμό των επιμέρους ε, συνεισφορών προς το Ταμείο. Εδώ εν μέρη προτείνεται είτε ενεργά ο υπολογισμός ε, των σπρέτ ε, των κινδύνων ε, είτε απάλληψη και σε σχέση με την πρόταση αυτή πρέπει να βρούμε μια μέση οδό και πάλι. Ας αφήσουμε εδώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουμε ένα πρότυπο που μπορεί να υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη αν σε σχέση με την αγορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ταιριάζει αυτό. Όμως ταυτόχρονα αφήσουμε στα κράτη-μέλη την ελαστικότητα στη διάθεσή τους να κάνουν δικούς τους ξεχωριστούς υπολογισμούς τα κράτη-μέλη που από τις ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, θα πρέπει να μπορούν να συντεριάζουν με αυτές, όχι αυθαίρετες ε, καταστάσεις δηλαδή, αλλά να υπάρχει μια ομοιομορφία των απαιτήσεων για τα πρότυπα και τις μεθόδους υπολογισμών που θα γίνονται. Αυτά ω επισκόπηση για τι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί και μια αξιολόγηση από πλευρά μου αυτές, για αυτέ τι τροπολογίε. Χαίρομαι για τι συζητήσεις με τους γεώδεις συζητητέ και του άλλου συναδέλφους που έχουν καταθέσει τροπολογίε που όπω είπα και εγώ είμαι πραγματικά ευελπιστό ότι σε πολλά σημεία μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. That was a... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ εκτενής η παρουσίασή τώρα πιέζει ο χρόνος. Θα δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στη Βίκη Φόρντ γιατί ξέρω πως πρέπει να φύγει και τον Μπέρκχαρτ. Οπότε ελπίζω να είστε σύντομοι. Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει εδώ πέρα και ευχαριστώ όλους τους εμπλεκομένους. Συμφωνώ πράγματι για το ζήτημα της εγγύησης ε, καταθέσεων και πρέπει να σκεφτούμε λίγο το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα, όχι μόνο για να βοηθήσουμε μόνο τους ε, καταθέτες, αλλά για να οδηγηθούμε σε μια λύση. Εάν ε, τα χρήματα π.χ. αφορούν κατάθεση σε, άλλο, σε κάποιο άλλο book, εντάξει, αλλά εάν πηγαίνουν κάπου αλλού, σε, π.χ. για την κεφαλαιοποίηση ενός ε, τραπεζικού ιδρύματος, τότε πλέον δεν έχουμε ίσως ανταγωνισμού, οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα σχέδια εγγύησης καταθέσεων. Επίσης συμφωνούμε για, τις, για τα παραρτήματα, δηλαδή τις προτάσεις που μπορεί να κάνει η Επιτροπή και μπορούν μετά να εφαρμοστούν. Βεβαίω, ο αναλόγω με τι ώρε που ισχύουν σε κάθε χώρα, γιατί συμφωνώ πω πρέπει να είναι ίσε οι συνθήκε ανταγωνισμού, υπάρχουν και διαφορετικέ τοπικές παραλλαγές στις αγορές και πρέπει βέβαια να λειτουργήσει το σύστημα. Δεδομένου του ότι ανησυχώ λίγο για, τον αποκλεισμό, για την εξαίρεση στο άρθρο 11 παράγραφος 1 που πηγαίνει κάπως παραπέρα από τοπικές ε, παραλλαγές. Ε, ναι, πράγματι πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το εξάντε, την εξάντε χρηματοδότηση σε σχέση με την εξπόστ κατά βάση πρέπει να φροντίσουμε να μπορούν ε, να λαμβάνουν ε, γρήγορα τα χρήματά τους σε περίπτωση κατάρρευσης της ε, τράπεζες μέχρι το εγγυημένο ποσό η καταθέτηση, αλλά πρέπει να δούμε γενικότερα τη συζήτηση και τα στοιχεία ρευστότητα και το ότι όσα γίνονται μέσω της βασιλείας, της περίοδους παρατηρήσεις που κάνουν όλοι παγκοσμίω για να έχουν επαρκή ρευστότητα και να μην καταρρεύσουν εξ αρχή οι τράπεζες. Πρέπει να φροντίσουμε πώ θα υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στην περίπτωση που θα έχουμε μια κατάρρευση, αλλά στη Βασιλεία μιλάμε για μια περίοδο παρατηρήσεις ε, υπό παγκόσμιε κατευθυντήριες γραμμές για να δούμε τα... της Αλλά ίσως ε, δεν ξέρω, πρέπει ίσως να αποσαφινιστεί πώς μπορούν και τα κράτη-μέλη να κάνουν μια τέτοια περίοδο παρατήρησης σε σχέση με το εξάντε και εξπόστ για να δούμε το ζήτημα τη ρευστότητα μετά από την περίοδο αυτή η παρατήρηση όπως σα είπα για να μην καταραίουν ούτω ή άλλως οι τράπεζε να φροντίσουμε να προστατεύονται οι καταθέτες και να υπάρχει ρευστότητα για τις ε, τράπεζες και πως είναι σε θέση να δανείζουν και την ευρύτερη οικονομία. Θεωρώ πως υπάρχει ένα σύστημα πιθανούς ε, προχρηματοδότησης που μπορεί να μην οδηγήσει στην, ε, στην κύκλική συμπεριφορά που ανέφερε, πράγματι Πίτερ, και βασικότερο δεν χρειάζεται να πληρώσει και ο φορολογούμενος. Αλλά είναι μετά ευρύτερο ζήτημα το εάν θα μείνει σε ένα χωριστό λογαριασμό, θα μείνει σε ένα χωριστό λογαριασμό αυτά τα χρήματα ή εάν θα παραμείνουν εντός των ιδίων των ε, πιστοτικών ιδρυμάτων. Οπότε συμφωνώ με τις ε, τροπολογίες. Τώρα προσωρινά υψηλά υπόλοιπα λογαριασμού είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε με την ε, Σάρον ε, για το την περίπτωση αυτή, στην οποία παραδείγματος χάρη είναι παγωμένο το ποσό, στην περίπτωση που κάποιος έχει πεθάνει, ε, να μην μπορούν να περάσουν σε διαφορετικούς λογαριασμούς τα, τα χρήματά τους. Τέλος, για την εκταμίευση, είπαμε για την διαφορά δύο με πέντε ημερών, μία εβδομάδα, υπάρχουν και αργίες ενδιάμεσα. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση λοιπόν, καθώς ε, πάρα πολύ συχνά μπορεί να γίνει και στην αλλαγή του έτους ε, η κατάρρευση μιας τράπεζας. Ο Σβέν επίσης μίλησε για οργανισμούς χαμηλού ρίσκου, μπορούμε να το δούμε, αλλά ίσως θα μπορούσαμε απλά στα παραρτήματα να πούμε πως αυτό ισχύει για την κάθε χώρα, για τη συγκεκριμένη χώρα που εξετάζουμε. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν μπορούσα να επιταχύνουμε, διότι φορετικά θα πρέπει να βγάλουμε σε μια την σε διάταξη. Ο Μπέρκαρτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι μπορώ να είμαι πραγματικά σύντομο υπό το πρίσμα το δικό μου τα ουσιαδέστερα σημεία για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκθεση τα συζητήσαμε ήδη την προηγούμενη συνεδρίασή μας και εγώ φυσικά θέλω στους συναδέλφους να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες αυτές. Πιστεύω ότι πολλές τροπολογίες θα μπορέσουν να συγχωνευτούν, θα πρέπει να συγχωνευτούν σε συμβιβαστικές τροπολογίες, ώστε στο τέλος τέλος δεν θα πρέπει όλες τις 215 αυτές τροπολογίες να ψηφίσουμε, αλλά λιγότερες. Κυρίως με ευχαριστεί το γεγονός ότι η κυριότερη σκέψη της έκθεσης βρίσκει ευρεία συνένεση από τα μέλη. Υπό το δικό μου πρίσμα το άνοιγμα της αρχής Paybox της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν κάτι κατεπηγόντως αναγκαίο ώστε οι de facto διαφορές των τραπεζικών συστημάτων στα κράτη-μέλη με σωστό τρόπο να μπορέσουν να ενταχθούν. Γι' αυτό στο σχέδιο έκθεσης προσπαθήσαμε την συγκεκριμένη διαμόρφωση των συστημάτων διασφάλισης να το αφήσουμε στους ίδιους τους εμπλεκόμενους ως υπεύθυνους να το διαμορφώσουν. Ταυτόχρονα όμως στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τίθενται τα πράγματα σε μια δυνητική εθελοντική βάση και είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε και πάλι. Ένα σύστημα διασφάλισης καταθέσεων μπορεί τα κονδύλια για προληπτικά μέτρα να τα χρησιμοποιεί, δεν πρέπει όμως υποχρεωτικά να το κάνει αυτό. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που πάνε προς την κατεύθυνση χρηματοδότησης εξάντε και και για τη δυνατότητα της χρήσης κονδυλίων κάτι τροποποιούν, κάτι αλλάζουν. Παρ' όλα αυτά η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων υποστηρίζει αυτή την αρχή που προανέφερα. Υπό το δικό μου πρίσμα λοιπόν δεν θα πρέπει να συζητήσουμε θέματα αρχής στη συζήτηση αλλά κυρίως θα πρέπει οι προθεσμίες καταβολής των ποσών, το ύψος των ποσών, ο υπολογισμός των κινδύνων, οι εισφορές, συνεισφορές και τα διαθέσιμα κονδύλια να τεθούν στο τραπέζι και να ε, ξαναεξεταστούν. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία καταβολής αυτών των ποσών και υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη με το, το Συμβούλιο θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να γίνει στο τέλος ε, ως τελική πρόταση. Το ίδιο ισχύει και για τα τελικά ποσά και για τον υπολογισμό των εισφορών. Θα πρέπει πάλι νομίζω να ξανασυζητήσουμε τα θέματα των spreads Παρ' όλα αυτά όμως ε, τις γνωμοδοτήσεις ε, της ε, Γιούρι και Ίνκο θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και όχι ένα άνοιγμα μόνο προς τα πάνω να δούμε αλλά και μια ειδική ρύθμιση για τους κινδύνους που ενδεχόμενα θα πρέπει να εξεταστούν για ένα άνοιγμα προς τα κάτω θέμα των διαπραγματεύσεων, συμβαστικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι ποια κονδύλια για τις πληρωμές αυτές στα ταμεία ασφάλισης θα πρέπει να γίνουν δεκτά. Εγώ θεωρώ ότι η τροπολογία του φίλου και συναδέφου Ζαν Πολ Γκοζές είναι πολύ καλή πιστεύω ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια συμβιβαστική γραμμή για όλους. Ευελπιστώ ουσιαστικά ότι σε αυτή την τελική ρύθμιση των πραγμάτων και τελικό συντονισμό θα τα καταφέρουμε και θα καταλήξουμε σε αποδεκτούς συμβιβασμούς. Ευχαριστώ πολύ. Wolf. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Βούλφ. Ουσιαστικά όλα αναφέρθηκαν, αλλά όχι από όλους. Και γι' αυτό και από μένα κάποια σύντομα σχόλια, αν Έχουμε συντονιστεί πολύ καλά σε σχέση με τον εισηγητή για αυτό το θέμα και κατά τούτο βρισκόμαστε πολύ κοντά στις θέσεις μας ο ένας με τον άλλο. Χαιρετίζω αυτή την προσέγγιση του Paybox ως ξεχωριστού στοιχείου που θα ενταχθεί. Το βρίσκω όμως και καλό ότι παρόλη τη συμφωνία για την θεσμική διασφάλιση όπως την έχουμε στη Γερμανία για παράδειγμα και τέτοιου είδους ιδρύματα για να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις και να υποχρεούνται τα 100.000 ευρώ ξεχωριστά να τα διασφαλίζουν αυτή τη ρύθμιση έτσι. Αυτό δεν αντιμετώπισε πάντα μεγάλη ικανοποίηση, αλλά νομίζω ότι επιβάλλεται μια τέτοια ρύθμιση. Χρειαζόμαστε μια πολύ σαφή τοποθέτηση όσον αφορά την ε, πρικοδότηση με κονδύλια και για τον υπολογισμό όσον αφορά τις εισφορές. Πιστεύω ότι οι εγγυημένε καταθέσεις οι εγγυήσει για τις καταθέσεις θα μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουν όταν θα έχουμε ένα αναβαθμισμένο τέτοιο επίπεδο για την ποιότητα. Δεύτερον, είμαι απόλυτα υπέρμαχος της χρηματοδότησης ex ante. Και έτσι λοιπόν ε, δεν θα έπρεπε να έχουμε ξεχωριστέ ρυθμίσει σαν κράτο μέλο. Αυτό θα οδηγούσε σε στρεβλώσει. Τουλάχιστον μετά από μια μεταβατική περίοδο, μετά από κάποια χρόνια, πρέπει να έχουμε μια εξ άντε εκ προημίου, εκ των προτέρων χρηματοδότηση. Και αυτό θα έπρεπε να ε, λειτουργήσει δεν θα έπρεπε αυτό να θεωρηθεί πρόβλημα. Όσον αφορά την πρικοδότηση με τα κονδύλια, πραγματιστική πρόταση για την καταβολή ε, αυτών των ποσών θα έπρεπε να είναι οι πέντε μέρες ή μια εβδομάδα για να μπορέσουμε αρχικά έτσι να λειτουργήσουμε. Σημαντικό είναι και αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κατάχρηση με αυτό το pay box ώστε κάποιες αδυναμίες όσον αφορά την πρικοδότηση με κονδύλια με αυτόν τον τρόπο να αντισταθμίζονται. Μόνο το πολύ πολύ μια γεφυροποίηση, μια μεταβατική περίοδο θα μπορούσε έτσι να ε, καλυφθεί με αυτή τη ρύθμιση. Επαρκούμε σε αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Ευχαριστώ. Γιώργεν, θα μιλήσεις στο λόγο. Α, συγγνώμη Σβέν. Τάχασα, χασα, μπερδεύτηκα. Δεν κανένα πρόβλημα. Θέλω... Θα ήθελα πρακτικά να πω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα σημεία τα οποία προανέφερε η εισηγητής. Δεν θέλω να επαναλάβω εδώ διάφορα πράγματα. Οι διαφορές σε σχέση με αυτά τα οποία ανέφεραν οι προλαλήσαντες δεν είναι πολύ μεγάλες. Λοιπόν, θα ήθελα σε δύο πράγματα να αναφερθώ όσον αφορά τον Λάγκαν. Το πρώτο είναι το ερώτημα, το ζήτημα, τι γίνεται σε σχέση με τους κινδύνους και τη διαφορά των διαφορετικούς κινδύνους όσον αφορά τις διάφορες συνεισφορές ε, για τα ασφαλιστικά συστήματα, όσον αφορά διάφορα ιδρύματα. Στην αρχική προσέγγιση άρθρο 11.1 τι λέγεται. Ένα πρότυπο αναφέρεται και στο 11.3 σε αυτό το άρθρο ανοίγει η προοπτική προς την κατεύθυνση εθνικά τα κράτη-μέλη να μπορούν να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα πρότυπα όμως ανταποκρίνονται και περιγράφουν σε σχέση με την διαφορά όσον αφορά την συνεισφορά. Και αναφέρεται εδώ διαφορά μεταξύ 75% και 200%. Και αν αυτά τα συγκρίνουμε με το πραγματικό κίνδυνο στον πραγματικό κόσμο, αυτή η διαφορά είναι πιο μικρή γίνεται δεκτό τις εξαιρέσεις και 37,5% θα μπορεί να είναι αυτό το ποσοστό. Αυτή η διαφοροποίηση δεν επαρκεί όμως ώστε η διαφορά μεταξύ μιας ε, πολύ στεναρής ε, τράπεζας, στεγαστικής τράπεζας ή στεγαστικού ταμιευτηρίου να αντισταθμίσει τα πράγματα με μια τράπεζα που κάνει, ας το πω έτσι, ε, επενδύσεις κεφαλαίου και εκτίθεται σε μεγαλύτερους κινδύνους. Αυτό όμως είναι άδικο, διότι μόνο αν οι συνεισφορές ανταποκρίνονται στον πραγματικό κίνδυνο κάτι τέτοιο θα ήταν δίκαιο. Και γι' αυτό θα πρέπει για αυτό το θέμα να ξανασυζητήσουμε. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι σε αυτό το σημείο φυσικά θα πρέπει και για τους τύπους ε, που χρησιμοποιούνται στο παράτημα ή τους προσδιορισμούς του παρατήματος να συζητήσουμε. Και έτσι σε σχέση με τις προτάσεις ακριβώς ε, που οι προτάσεις που υποβάλλονται δεν πρέπει οι σταθερές ε, τράπεζες, οι αξιόπιζες τράπεζες να επιβαρυνθούν ε, υπέρμετρα και αυτό πρέπει να είναι ένα μάθημα το οποίο θα συναγάγουμε από αυτή την κρίση. Δεύτερο σημείο που σύντομα θέλω να αναφέρω, πόσο συγκρίσιμα και παρόμοια πρέπει να είναι αυτά τα ε, θεσμικά όργανα μέσα στο πλαίσιο αυτών των εγγύσεων. Έχουμε κάποιες τροπολογίες που στοχεύουν να δημιουργήσουν μεγάλους περιορισμούς, ιδιαίτερα όσον αφορά το σύστημα των ιδρυμάτων και της κατοχυρωσής τους, τροπολογία 108 και 139 έχω υπόψη μου για παράδειγμα. Αυτά όμως για τα μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπου σε σχέση με τις κεντρικές δομές ε, με τις οποίες συγκρίνονται ή θα τους επιβαλόντουσαν, αυτό θα δημιουργούσε ιδιαίτερε επιβαρύνσεις ε, για αυτά τα μικρά ιδρύματα. Συμφωνώ εν τέλει με την παρατήρηση ότι είναι ακριβώς αντιπαραγωγικό με τέτοια συστήματα να τα χρηματοδοτούμε εξ post, εκ των υστέρων διότι ακριβώς εκείνη στη συνέχεια όσον αφορά ε, την καταβολή αυτών των κονδυλίων θα εξαιρούνται εκείνοι οι οποίοι θα έχουν συνεισφέρει περισσότερο στη δημιουργία αυτού του προβλήματος. Δεν είναι αυτό η σωστή εφαρμογή των κανόνων για τον ανταγωνισμό. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τους εισηγητές και πιστεύω ότι κάτι στο λογικό και το καλό θα καταλήξουμε να εγκρίνουμε. Και τα προβλήματα τα οποία η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δημιουργούσε για προληπτικές δράσεις ε, που είναι προς στο συμφέρον ενός σταθερού χρηματοοικονομικού συστήματος αν μπορούμε να τα αντισταθμίσουμε σε συνεργασία και με το Συμβούλιο να μεριμνήσουμε ε, περισσότερα πρότυπα διασφάλισης αυτών των ιδρυμάτων να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτό θα ήταν θετικό για τις χρηματοοικονομικές αγορές στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα, Γιώργεν. Ευχαριστώ. Πράγματι θα είμαι σύντομος γιατί έχουν υποθεί όλα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ λοιπόν για την συνεργασία με τον εισηγητή. Να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε ο προλαλής σας προς των δύο μοντέλων ασφάλισης για εμάς πρέπει να υποστηριχθεί και βεβαίως ε, χαιρετίζουμε ότι καταλήξαμε σε ένα λογικό συμβιβασμό χρηματοδότηση εξάντε ή εξπόστ για εμάς είναι σαφές. Εξάντε δεν θέλω τώρα να το ιδεολογήσω, έχουν ακουστεί για τους ε, στόχους επάρκειας ε, στο ύψος ε, που ακούστηκε, το υποστηρίζουμε και θεωρούμε απαραίτητο αυτό το οποίο έθεσε ο Σβέν για τον κίνδυνο. Εκεί πέρα επί της είμαστε διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε την πρόταση του Σβέν Α, θεωρώ βεβαίως πως θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια λογική λύση. Αν είναι δυνατή αυτή βεβαίως και στα παραρτήματα, οι τύποι που υπάρχουν εκεί πέρα είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Αυτά από μένα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαν οι σκιώδεις όσον αφορά το, τους αγορητές. Είμαι εγώ, η Αρλίν, ο Αντελίν και έχουμε πολλούς. Θα περιοριστώ εγώ σε τομείς που είναι διαφορετικοί. Όσον αφορά τις τοπικές αρχές ή κατά πόσο θα πρέπει να έχουν ε, τη δικαιοδοσία είτε όχι, κάνω διάκριση με το μέγεθος, ανάλογα αν έχουν επαγγελματικό ταμεία, επαγγελματία ταμεία που υποτίθεται ότι τα επιβλέπει όλα αυτά είτε όχι. Πρέπει να παραδεχτώ ότι βασίστηκα στην δική μου εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το θέμα αυτό με την τοπική αυτοδιοίκηση όπου κάποια πολύ μικρά τοπικά συμβούλια, μικρές ενορίες, ε, κάποιοι φορείς έχουν κάποιον που ξέρει τα πράγματα υποτίθεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθούν τα χρήματά τους πάρα πολύ ε, προσεκτικά. Κάποιοι έχασαν τα χρήματά τους στην όλη ιστορία της Ισλανδίας και προειδοποιήθηκαν να βγάλουν τα χρήματά τους από την άλλη και δεν τα πέσυραν. Δεν νομίζω ότι τις μεγάλες τοπικές αρχές θα πρέπει να τις θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο. Όσον αφορά εκ των υστέρων, εκ των προτέρων. Θυμάμαι στην προηγούμενη θητεία είχαμε το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων και των μηχανισμών και ο τότε ηγητή ήταν πολύ σκεπτική όσον αφορά τα διάφορα σχήματα ελέγχου των υστέρων, διότι θεώρησε ότι θα μαζευτούν πολλά τα χρήματα, αλλά είχε επίση δισταγμού και για τα σχήματα εκ των προτέρων, διότι θεωρούσε ότι τα χρήματα δεν θα μαζευόταν ούτε σε αυτή την περίπτωση. Ε, νομίζω ότι αν διαβάσετε λοιπόν την ομιλία του στην Ολομέλεια του ηγητού είναι ενδιαφέροντα τα πράγματα. Προσπάθησα να τα εξορροπήσω όλα αυτά λέγοντα ότι ίσως μπορεί να δείξει κανείς την κεφαλοχική βάση, την μέση κεφαλοχική βάση. Αν υπάρχει πολύ ψηλά κεφαλοποιημένο τραπεζικό σύστημα, ίσως θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερη χρηματοδότηση των ε, ενώ αντίθετα από μια τράπεζα που δεν είναι τόσο υψηλά κεφαλοποιημένη, διότι θα είναι διαφορετικοί παράγοντε κινδύνου. Ανησυχώ όσον αφορά το, τους σκοπούς χρήσεως του Ταμείου, Μ' αρέσει η ιδέα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνέχεια παροχής υπηρεσιών προς το κοινό το σημαντικότερο είναι ο κόσμος να έχει πρόσβαση στα χρήματά του. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη όσον αφορά διευθετήσεις που επιτρέπουν μεταφορές και συνέχεια πρόσβασης. Αλλά ε, ανησυχώ για χρήση αυτού για επίλυση εκτός από αυτή την διατήρηση της συνέχειας για άλλους σκοπούς. Εάν προσπαθεί το Ταμείο αυτό να διασώσει διάφορα τραπεζών και το καθεξής ε, και σε άλλες χώρες, τότε αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό όσον αφορά τον καταναλωτή. Εγώ είμαι εκείνη που μπήκα στο παράρτημα και όχι για πρώτη φορά και προσπαθούσα να αλλάξω τα πράγματα και κατέληξα στο συμπέρασμα και όχι για πρώτη φορά ότι η βαθμολόγηση, οι δείκτες, αναλογίες κλπ, ποσοστά, όλα αυτά θα έπρεπε να εξεταστούν. Νομίζω ότι υπάρχει συνωμοσία εναντίον μας, διότι στο πρόγραμμα στις 4 το πρωί δεν μπορείς να μπει ανθρωποποίηση στο παράρτημα. Αυτό που έκανα ήταν ότι θεωρούσα ότι θα πρέπει να είναι στις κατανάθεσιν πράξεις Ε, κατ' ουσίαν πηγαίνουν στο Συμβούλιο. Ήθελα να κρατήσω όμως το πλαίσιο. Να αλλάξουν οι αριθμοί μέσω τεχνικών προδιαγραφών. Έχω συγκεκριμένο πρόβλημα όσον αφορά το κέρδος ε, σαν δίκτυ κινδύνου. Αν έχουμε μια ε, ε, επιχείρηση που βγάζει πολλά κέρδη, αυτό είναι, έχει πηγαίνει τους κινδύνους. Δεν είναι αυτό ένα κινητήρα για υπερβολικό κέρδο από κάποιε τομεί. Ε, το μπόνους, σαν κίνητρο δηλαδή. Και δεν ταιριάζει και το θέμα της αντασφάλισης που δεν έχει μέγιστο κέρδος για λόγο ύπαρξης. Κατέληξε συμβιβασμό. Άφησα το πλαίσιο. Τι θεωρείται δείκτης κινδύνου αφαίρεσα το στοιχείο του κέρδους για να μην παρισφρήσει εκ νέου μέσω των εξουσιοδότηση πράξεων. Γι' αυτό ακολούθησα αυτή την προσέγγιση. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Δεν ξέρω αν το σύστημα επέτρεψε να τα εκφράσω σωστά. Ίσως δεν είναι βέλτιστη λύση. Ίσως πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Κάποιες πτυχές κέρδους επηρεάζουν την κατάσταση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο. Απλώ ήθελα να πω ότι έχω πραγματικό πρόβλημα όσον αφορά το στοιχείο του κέρδου. Διότι ίσω είναι κάπω αντίστροφο κίνητρο. Στρεβλό κίνητρο. Δεν ήθελα να πειράξω άλλα πράγματα. Δεν ήθελα να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Τελείωσα. Έχω άλλες ε, τροπολογίε που νομίζω ότι είναι εύκολο να εξηγηθούν. Δίνω το λόγο στην Αρλίν. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, λέει η Αρλίν. Τρία έχω να πω πράγματα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή καταρχά. Πολύ ισχυρή έκθεση, σαφέστατη. Το θέμα του νομίσματος, το συνάλλαγμα, το νόμισμα στο οποίο πιστεύω τα χρήματα. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, το άρθρο 5 λέει ότι πληρώνουμε ε, τον καταναλωτή στα χρήματα του λογαριασμού πρέπει να πληρώνεται ο καταναλωτή ακριβώ το νόμισμα που κατέθεσε. Στο νόμισμα του λογαριασμού. Α το σκεφτεί η Επιτροπή πολύ προσεκτικά. Εάν θα αλλάξουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικά με αυτό. Εάν υπάρχουν λόγοι για να αλλάξουμε την πρόταση, πρέπει να το δικαιολογήσουμε. Διαφορετικά, ο καταναλωτή πρέπει να επιλέγει για να μην χάσει από αλλαγή συναλλάγματο, αλλαγή νομίσματο. Εκτιμώ κάποιε τροπολογίε τη Προέδρου και τη κυρία Φόρντ για προσωρινά υψηλές αποταμιεύσεις. Η δωδεκάμενη περίοδος για προσωρινέ τέτοιε καταθέσει, ή καταθέσει θα μπορούσαν να γίνουν δεκτέ, γιατί να μειώσουμε την προστασία του καταναλωτού. Δεν θέλω να μειωθεί. Αν υπάρχει λόγο, σα το κάνουμε, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό που να δικαιολογεί την τροπολογία. Ο κ. Μπάρα, ο σκιώδη του εισηγητή, σωστά είπε ότι πρέπει να εξετάσουμε τι τροπολογίε που υποβάλλονται από τις επιτροπές που συντάσσουν γνωμοδοτήσεις, κυρίως από τις τροπολογίες ΙΜΚΟ 33 και 36 για το άρθρο 14, στην περίπτωση συγχωνεύσεως χρηματοστικών οργανισμών η αλλαγή κάλυψη από τα συστήματα εγγύσεως καταθέσεων ο καταναλωτής πράγματι θα πρέπει να δικαιούται μέρη να αποσύρει τις καταθέσεις του χωρίς να, χάνει, να του επιβάλλονται κυρώσεις και να χάσει τόκους. Ελπίζω να λάβει υπόψη η Επιτροπή τις στοιχείες του καταναλωτού που είναι σημαντικά θέματα για μας να εγγυόμεθα αυτές τις πτυχές στο σύστημα εγγύσεως καταθέσεων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δίνω την Προεδρία στην Αρλίν. Επόμενος αγορητής είναι ο Αντολίν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου στα συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια, διότι έκανε εξαιρετική δουλειά στα συστήματα εγγυήσεων καταθέσεων που έχουν πολύ μεγάλη σημασία στον αφορά τον ανταγωνισμό, ώστε να υπάρχει ένα ισοδίκαιο πεδίο δραστηριότητας στον ανταγωνισμό και η σταθερότητα και το κόστος σε σχέση με τις εγγυήσεις για τα κράτη-μέλη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ότι η ε, εγγύησης αυτές θα είναι επιβάρυνση και να είναι προς όφελος των καταθετών. Είναι ένα σύστημα σε σχέση με την χρηματοδότηση εξάντε που είναι θεμελιώδες και αυτό μπορεί να συνεισφέρει για την σταθερότητα και αυτό είναι ένα κεκτημένο και έχει και ένα προληπτικό χαρακτήρα αυτό το σύστημα που είναι ιδιαίτερη σημασία. Αυτή στην πρώτη γραμμή πρέπει να είναι η κατεύθυνση και να είναι πιο φθηνό και σε σχέση με τη διασφάλιση των καταθέσεων για τις τροπολογίες μου που τις ε, κατέθεσα θέλοντας να προσφέρω κάποια στοιχεία ώστε η συγγήτρια να μπορεί να καταλήξει σε συμβιβασμούς και να μπορούν να υπάρξουν κάποια σημεία αναφοράς ε, για τεχνικά ε, θέματα. Προσπάθησα να υπογραμμίσω ότι είναι ένα σύστημα εθελοντικό και ευρωπαϊκό ταυτόχρονα, ευρωπαϊκό, όχι μόνο στο πλαίσιο του για τις καταθέσεις, αλλά αφορά όλα τα ιδρύματα και τους φορείς που έχουν καταθέσεις. Και όλα αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν σε συστήματα εγγύησης καταθέσεων, με ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας ώστε να υπάρχει ένα συντονισμός για το υποπτικό έργο. Και από το 2013 όπου θα υπάρξει και η αναθεώρηση, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σε βάθος μεταρρύθμιση και να έχουμε και τη δυνατότητα ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου, όπου θα εντάσσονται τα εθνικά ταμεία και οι διάφορες πηγές που θα μπορούν να συνεισφέρουν, να μπορούν να αντληθούν μετά από αυτό σε υπερεθνικό επίπεδο. Ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε επιλύσει ακόμα και που πρέπει και πολύ με θετικό τρόπο που αναφέρεται στην έκθεση και που πρέπει έτσι να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να εκφράσω ε, κάποια θέματα σε σχέση με αυτό. Θέλω να προσθέσω τη φωνή μου στα θετικά σχόλια για το έργο της εισηγήτριας. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα τα οποία συζητώνται εδώ, θα μπορούσαμε να διαρωτηθούμε αν η πενθήμερη ή επταήμερη προθεσμία είναι μια βιώσιμη πρόταση. Πολλές φορές ε, τρεις μέρες χρειάζεται ένα έμβασμα να φτάσει από μια χώρα στην άλλη. Καλή ιδέα θα φαίνεται να είναι, παρότι όμως μπορεί να μην είναι λειτουργική, ακόμα λαμβάνοντας υπόψη τη μετεξέλιξη του συστήματος. Δεν θα επέτρεπε μια τέτοια λειτουργία το σύστημα όταν κάποιος αποφασίζει, ένα σύστημα που αποφασίζει ποιο διάστημα θα πρέπει να, χρησι, να ε, χρειάζεται χωρίς ε, οποιαδήποτε διασφάλιση ε, καταθέσεων καταθετών σήμερα. Θα έπρεπε να καθορίσουμε μια προθεσμία που θα είναι ευέλικτη. Η πρόταση η, λαμβάνει υπόψη την πρόταση του, των down payments, των προκαταβολών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του συστήματος και να συσχετίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων αλληλοεμπιστοσύνη. Δημιουργούμε ένα σύστημα που πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο της εμπιστοσύνης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης ως βάση. Και σε σχέση με την πρόταση, μία πρόταση ότι τα ιδρύματα αυτά θα πρέπει να συνεισφέρουν σε περίπτωση πτώχευσης ε, χρεοκοπίας ε, μιας ε, τράπεζας. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση ότι ένα ίδρυμα θα εμβάζει, θα δίνει τέτοια κονδύλια θα πρέπει να προηγείται από μία προκαταβολή ή εισφορά όσον αφορά τις ε, εγγυήσεις ε, πρέπει η βάση εμπιστοσύνης να θεμελιώνεται σε τεκμήρια και γεγονότα και όχι σε μία πληρωμή χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση για επιστροφή. Ένα άλλο θέμα για τα συγκεκριμένα έγγραφα. Κάτι που είναι σημαντικό είναι το θέμα του ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός ε, αρρύθμιστος ή ε, στρεβλός. Θα πρέπει να ρυθμίζονται τα, οι σχέσεις μεταξύ των Ιδρυμάτων. Θα πρέπει ίσως εδώ να εισαχθεί ένας μηχανισμός που να μπορεί να ενημερώνει εκ προημίου για τις ε, εγγυήσεις αυτές με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγουμε το να αποφύγει μία τράπεζα αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ε, να μην είναι δυνατόν δηλαδή να εξαιρεθεί να πρέπει να πληρώνει τα, τους τόκους ε, για αυτά τα ποσά εφόσον εκκρεμούν για παράδειγμα μια εξάμηνη διάρκεια για την ε, τελική καταβολή των ποσών. Επίσης θα έπρεπε να δούμε αν είναι δυνατόν να συνμηθεί να επιβραχυνθεί αυτή η περίοδος, αυτή η διορία. Υπάρχουν διάφορες ε, προτάσεις ε, για το ε, τελικό ποσό όσον αφορά τα, τις τελικές αυτές πληρωμές. Μία πολύμηνη περίοδος είναι υπερβολικά μεγάλη και θα πρέπει να μπορέσουμε να την επιβραχύνουμε και μία περίοδος που θα είναι πιο σύντομη θα ήταν ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ. Έχουμε μείνει 30 λεπτά πίσω. Με 320 τροπολογίες έχεις πολλή δουλειά να κάνεις, προσπαθώντας να πετύχει συμβιβασμού και να μιλήσει στου διάφορους που υποβάλλουν τροπολογίε, τροπολογίες. Οπότε, εν συντομία, αν μπορεί να ανακεφαλαιώσει χωρί να ανταποκριθεί σε διάφορα σχόλια. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση. Ευχαριστώ για τι ε, πρώτε 115 τροπολογίε. Ε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Για τις υπόλοιπες ήδη προηγούμενα τοποθετήθηκα και είπα ότι σε πολλές ε, πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε καλή πορεία να καταλήξουμε σε κοινέ ε, προτάσεις, κοινέ ρυθμίσεις. Η συζήτηση αντανακλά μόνο μια εισαγωγή στα ουσιοδέστερα σημεία και έτσι δεν χρειάζεται εδώ να επαναληφθούν αυτά τα πράγματα. Τρία σημεία θέλω να αναφέρω που δεν κάλυψα πιο πριν και που τώρα ανεφύησαν στη συζήτηση. Καταρχήν από πλευρά ε, του συναδέλφου αν θα πρέπει έξι μήνες σε σχέση με αλλαγή ενός συστήματος πιο πριν να προαναγγείλω αυτή την αλλαγή. Είναι ένα σύστημα που για τους πιο διαφορετικούς λόγους πρέπει να συζητήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και προσβλέπω στις συζητήσεις που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον και για τον ε, προγραμματισμό και σχεδιασμό ασφάλειας σε σχέση με την κατάρτιση αυτών των συστημάτων ώστε να ε, μην ε, μας βρει απροετοίμαστους ε, μια τέτοια περίπτωση, ένα σενάριο αλλαγής σε σχέση με μια κρίση. Και για το νόμισμα στο οποίο θα πληρώνονται αυτά τα ποσά στο τέλος, εδώ έχουμε περιορισμό σε ευρώ και νόμισμα κράτους μέλους. Και ιδιαίτερα δεδομένων αυτών των μικρών περιόδων παράδειγμα πενθήμερη περίοδο, αν ε, περιοριστούμε σε αυτά τα δύο νομίσματα, τότε θα ε, μπορεί να ε, λειτουργήσει η πρόταση αυτή. Αν όμως έχουμε και τις πιο απίθανες ρυθμίσεις για τρίτα νομίσματα, επί πλέον νομίσματα, τότε δεν θα είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα εύθετο χρονικό διάστημα στην καταβολή αυτών των ποσών. Τρίτο σημείο το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε είναι η ανάπτυξη των περαιτέρω εθνικών συστημάτων προ ένα ευρωπαϊκό ε, δίκτυο ασφάλεια. Πράγμα που είχαμε ζητήσει ω Κοινοβούλιο στο παρελθόν να δημιουργηθεί, να γίνει. Θέμα είναι κατά πόσον θα προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό ταμείο και πόσον είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Και από πλευρά του συναδέλφου Σάντσε ε, Πρεσέντο, όπω ε, προαναφέρθηκε, αν θα γίνει αυτό ή αν θα αφήσουμε εθνικά συστήματα να λειτουργούν που σε κεντρικό, από κεντρική υπηρεσία θα συντονίζονται περαιτέρω. Για όλα αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να συζητήσουμε. Κατά τα άλλα ευχαριστώ πρέπει να πω τους συναδέλφους ε, για τις προτάσεις τους και κυρίως ε, για την ευρεία υποστήριξη στις προτάσεις ε, της έκθεσής μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε λοιπόν στις 9 Μαΐου για να πάει στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Περνάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα. Συστήματα εγγύηση των ασφαλίσεων. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης και 77 τροπολογίες και ε, εισηγητής είναι ο κύριος Σκίνερ. το λόγο. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε... Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους Όπω συνήθω ε, ήθιστε σε αυτέ τι περιστάσει, όσου υπέβαναν τροπολογίε και ιδιαίτερα ευχαριστώ του Σκιώδη. Δυστυχώ ο κύριο Καρά δεν μπορεί να παρίσταται και ο Ζων Πολ θα μιλήσει εκ μέρου του και άλλοι στην αίθουσα. Τα καλά μαντάτα είναι ότι έχοντα μιλήσει με του Σκιώδη εισηγητέ ε, και του εκπροσώπου χθε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε συμβιβασμού αρκετά γρήγορα όσον αφορά αρκετά από τα σημαντικά κρίσιμα θέματα και αν δεν έχει ήδη υποθεί Πολλά από αυτά που πρότειναν διάφοροι σαν ανεξάρτητες τροπολογίες φαίνονται ότι είναι πάρα πολύ καλές συμβουλές. Οπότε θεωρώ ότι τολμώ να πω ότι μπορούμε να βρούμε περιθώριο, να συμφωνήσουμε και αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή τίμια έκθεση, ειλικρινή έκθεση που θα μπορούσε να είναι η βάση συζητήσεων και επιχειρηματολογίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη λευκή βίβλο της. Είναι έκθεση ιδέα πρωτοβουλία, αλλά το Κοινοβούλιο τοποθετείται από το το θεμάτων, οπότε είναι σαφές ποια είναι η θέση μας και ελπίζω να μας ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να πω όσον αφορά τα μεγάλα ζητήματα και υπάρχουν και μεγάλα θέματα, θα μπορούσαμε να τα καθορίσουμε καταρχάς εκ των προτέρων έναντι εκ των υστέρων, όπως ακούσατε σε πρώτερη συζήτηση. Ο ορισμός ενός φυσικού προσώπου είναι κάτι που ήδη το αναφέραμε σε κάποιο βαθμό. Το πεδίο εφαρμογή όπως ισχύει για ζωή και μη ζωή ε, είναι δύο τμήματα το τομέα είδαμε στροπολογίες και τι γίνεται σε περίπτωση όπου μια ασφαλιστική εταιρεία δεν χρεοκοπήσει, αλλά γίνεται, ε, μπαίνει σε θέμα, σε ρευστοποίηση. Και τα χρέη μένουν επί μακρά περίοδο. Όταν με ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει στο run-off, δηλαδή δεν υπάρχει ρευστοποίηση, τα τα διοικητικές δαπάνες μειώνονται πολύ ε, σημαντικά, άρα έχουμε σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου. Η, η ασφάλεια δεν χρεοκοπεί. Συνήθως πληρώνονται οι άνθρωποι. Είναι το θέμα της μορφής που έχει ο τομέας. Δεν θα πρέπει να υπαρηφανεύονται γι' αυτό ότι μέχρι τώρα τα κατάφεραν να αποφύγουν κάποια από τα χειρότερα που πέρασε ο τραπεζικός τομέας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά να καλωσορίσουμε ότι αυτό συνέβη. Παρομοίω, θα πρέπει να εντοπίσουμε ότι υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ τη τραπεζική βιομηχανία και τη ασφαλιστική. Οπότε η αντιμετώπιση δεν πρέπει να είναι απαραίτητα ίδια και θα πρέπει να τα αποφύγουμε αυτό. Πάση θυσία. Με υψηλό κόστο αν υπάρχει. Λοιπόν, το θέμα ε, ποιο είναι ο φιλοξενούμενο. Όπω είμαι στη Φερεγκιότητα 2, Solvency 2, που είναι τεράστιο σχήμα εγγύσεω ασφαλίσεων. Ε, ακολουθήσαμε την εξή προσέγγιση, να υπάρχει επαρκέ κεφάλαιο και παραπάνω κεφάλαιο στο τέλος και επίσης επιμείναμε ότι θα πρέπει οι διάφοροι φορεί να κάνουν ό,τι πρέπει στις διασυνοριακέ. συναλλαγές. Λοιπόν, ελπίζω ότι το θέμα ε, χώρας έδρας και φιλοξενούμενου, home host, δηλαδή ο επόπτης της χώρας έδρας ε, θα είναι εκείνος που θα μπορεί να ε, συμβουλεύσει τους φιλοξενούμενους επόπτες όσον αφορά τι δραστηριότητε και τις ευθύνε ε, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τομήλου. Άρα είναι σημαντικό για να γίνονται αντιληπτοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Αυτό αφορά την προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να εστιαστούμε απόλυτα ούτω ώστε οι καταναλωτές θα μπορούν στο τέλος ε, να έχουν ένα, τους όρους να συμπεριλαμβάνουν σε νομικά δεσμευτικό έγγραφο, ε, μια σύμβαση. Εδώ διαφέρουμε από άλλου τομεί των χρηματοστικών υπηρεσιών. Έχουμε ένα νόμιμο συμβόλαιο και μπορεί να επιβληθεί μέσω ε, νομικής προσφυγής. Δηλαδή, σε μια χρονική περίοδο, όπως την Equitable Life στο Ηνωμένο Βασίλειο, που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τοποθετήθηκε υπέρ πολλών που προσέφηγαν στο Κοινοβούλιο και διαμαρτυρήθηκαν για τη χρεοκοπία αυτής της εταιρεία. Είδαμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, παραδείγματο χάρη, νομοθετική διαδικασία, δικαστική διαδικασία που κατέληξε στο διαμεσολαβητή, ο οποίος τοποθετήθηκε αποφάσει υπέρ όλων όσων προσέφηγαν ότι τα συμβόλαια τους είχαν παραπλανήσει οπότε η κυβέρνηση που ήταν υπεύθυνη για το εποπτικό σύστημα έπρεπε να παρέμβει. Άρα υπάρχουν κάποια συστήματα όπου πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σφαιρικά, ολιστικά και όχι να πηγαίνουμε σε κατά περίπτωση συνεπίληση όπως κάποιοι το έκαναν. Ε, εκτιμώ ότι ο τομέας ανησυχεί τα μάλα για το θέμα αυτό, αλλά το ίδιο και οι καταναλωτέ θα πρέπει να πετύχουμε ισορροπημένη προσέγγιση και θα πρέπει να είμαστε σωστοί και να μην υποθέτουμε ότι παρακολουθήσουμε αντιδράσει παρόμοιε όπω με άλλου τομεί και μέσω αυτού του τρόπου ότι θα ε, προστατεύσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους καταναλωτές. Ε, έχω να προτείνω πράγματα σε εκείνους που έβαλαν τροπολογίες όσον αφορά το θέμα ασφαλιών ζωής και μη ζωής. Ε, τους καταλαβαίνω, τους σέβομαι, αλλά πρέπει να τους πω ότι οι καταναλωτές οι οποίοι είναι στον τομέα μη ζωής ίσως να μην εμπλέκονται μόνο σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα, αλλά να ασφαλίζουν και τα σπίτια τους. Ε, επίσης εισιτήρια αεροπορικά. Και συμφωνούμε όλοι ότι ως καταναλωτές θα πρέπει να καλύπτονται το πεδίο αυτό, αν θέλουμε να μιλήσουμε για λογικότητα, το ύψος του κινδύνου ε, βλέπω βέβαια αυτή την προσέγγιση με τα χαρά να συνομιλήσω με άλλου που υπέβαλαν κάποιε τροπολογίε και να λάβω υπόψη κάποιε πτυχέ του θέματο αναλογικότητα του κινδύνου. Αλλά δεν θα πρέπει να δηλιάσουμε όσον αφορά το γενικό πεδίο που θα πρέπει να έχει αυτή η πρόταση. Θα σταματήσω εδώ κυρία Πρόεδρε αν επιτρέπετε και θα επανέλθω αργότερα σε αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν να μην ακούσουμε του κοιόδης ή... Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τους... Ε, να μην ακούσουμε του ήττε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τις ομάδες και μετά τους υπολείπους ναι. συναδέλφους. Από το ΕΛΚΟ, κύριος Γκοζές. Ευχαριστώ κυρία ε, Προέδρε. Ο κύριος Μάτμαν Καρά ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρίσταται και με ανέθεσε το καθήκον το αξιέπαινο να εκφράσω τη θέση του. Ε, και εκείνο θέλει να συγχαρεί και να ευχαριστήσει τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Ε, εκτιμεί τη διαφοροποίηση των διαφόρων τύπων ασφάλισης και θέλει να θετηθούν διατάξεις που αντικατοπτρίζουν αυτή τη διαφοροποίηση κατά την εφαρμογή των αποζημιώσεων. Εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το κείμενο αυτό επιτρέπει έναν ορισμό των διαφόρων σημείων των λεπτομεριών που παρέμεναν κάπω αόριστα στην αφαιρεγκαιότητα 2, Solvency 2. Υπογραμμίζει και ο Σόπτον Καρά στη σημασία τη εξαίρεση των, των ε, μεσαζόντων, ε, των ασφαλίσεων, των σύστημα εγγυήσεων, ε, βασμένοντα τη λευκή βίβλο ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά τη φερικαιότητα των διαφόρων ασφαλιστικών εταιριών δεν θα πρέπει να διευρυνθεί σε αυτό το στάδιο των συζητήσεων το πεδίο εφαρμογή. Λοιπόν, προθεσμία πληρωμών αποζημιώσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τι ασφαλιστικέ εταιρείε, καθώ και η εξολόγηση των αποζημιώσεων είναι πιο δύσκολο από ό,τι για μια τράπεζα και ίσω να χρειάζεται εφαρμογή ε, τεχνογνωσίας τεχνικών συμβουλών μπορεί η προθεσμία να αναβληθεί για τις αποζημιώσεις χωρίς εξαιρέσεις ε, ο Ότμαν Καράς θέλει να συζητήσει το θέμα των φυσικών προσώπων που έχουν άμεση σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία που είναι αφαιρέγγια, του διευθυντές, έχει χειριστές, ε, διοικητικά στελέχη και θα πρέπει να συζητήσουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ ασφαλιών ζωής και μη ζωής. Πριν από όλα το θέμα των διαφόρων μοντέλων ασφάλισης ζωής και μη ζωής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη επίσης τους διαφόρους κινδύνους ε, κάθε μοντέλου. Θα ήθελα να προσθέσω προσωπικά ότι το Ταμείο εγγύσεων των Ασφαλίσεων θα πρέπει προφανώ να παρεμβαίνει σαν τελευταία προσφυγή και αν δεχόμαστε το πεδίο εφαρμογή της ασφάλεια μη ζωή, θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε από τις ασφαλίσεως διασυνοριακού χαρακτήρα όπως των αυτοκινήτων. Αυτές παρατηρήσεις είχα για τον Ότμαρ και τις δύο τελευταίες που έκανα ήταν προσωπικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ ο κύριος Σμιτ για την άλλη της Φιλελεύθερης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ σέβομαι τον Πίτερ και τη δουλειά του ξέρει τι κάνει, αλλά ίσως μπορούσαμε ούτως ή άλλως να έχουμε κάποια επικοδομητική συζήτηση. Ε, κοιτάξτε, το θέμα είναι η προστασία των καταναλωτών, αλλά όπως υπόθηκε από τον Πίτερ και τον κύριο Γκοζές υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στην Ευρώπη και δεν καλύπτονται όλες οι χώρες. Ε, νομίζω είναι 20 από τα 27 που καλύπτονται και είναι πολύ διαφορετικά. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και είπατε πως ο κλάδος ενδιαφέρεται. Ναι, ενδιαφέρεται και έχουν έρθει και μαζί μου σε επαφή από την πατρίδα μου και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες πως παραπάει στη ρύθμιση. Εγώ είμαι υπέρ των εναρμονισμένων κανόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά νομίζω πως πρέπει να προσέξουμε αυτά τα ζητήματα. Όπως είπατε δηλώνουν πως ε, η φερεγγιότητα 2 υπάρχει ήδη και πρέπει να εφαρμοστεί. Ε, υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα εκεί πέρα για την προστασία των καταναλωτών. Και είπατε κι εσείς τις αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες δεν είναι οι ίδιες όπως ξέρετε στις ασφάλειες ε, σε σχέση με τις τράπεζες. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε αυτές τις ανησυχίες και ε, να βρούμε ένα σύστημα αποφελές και για τους καταναλωτές και για τον κλάδο και έχω πει πολλές φορές στην Επιτροπή μας κάποιο άσκησε κριτική βεβαίω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, πως δεν πρέπει να δημιουργούμε κανονισμούς και διαφορετικά συστήματα που εμποδίζουν τη λειτουργία της αγοράς. Και πρέπει επίσης να έχουμε κατά και το κόστος. Γιατί το κόστος για τον κλάδο, όπως ξέρουμε, τελικά θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Ξέρετε, ο Τζάμπα πέθανε. Οπότε πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Εσείς αναφέρατε πως ε, έχω κάποιες επιφυλάξεις για το πεδίο εφαρμογής οδηγίας και είπατε πως η ασφάλεια ζωής είναι ίδιες με την ε, ασφάλεια του σπιτιού. Δεν, δεν εννοώ αυτό. Αυτό το οποίο εννοώ είναι πως αν χρεοκοπήσει η εταιρεία, μια ασφαλιστική εταιρεία ε, και ελάχιστε το έχουν πάθει αυτό, αυτό το αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν τότε μπορεί κανείς να ασφαλιστεί σε άλλη εταιρεία μια μέρα στην άλλη. Αλλά βεβαίω αν καίγεται το σπίτι σας ταυτόχρονα τη στιγμή που χρεοκοπεί αυτή η εταιρεία τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Τέσσερα δεν ξέρω αν θα πρέπει να δημιουργούμε τέτοια συστήματα για να καλύψουμε αυτό το θέμα. Για την ασφάλιση αυτοκινήτου υπάρχει η ίδια συζήτηση. Ενώ να υπάρχουν κάποια σωστά επιχειρήματα. Γιατί να καλύπτεται κάτι τέτοιο. Και ίσως κάποια καλύτερα επιχειρήματα από αυτά τα οποία ανέφερα. Η αρχή της χρηματοδότησης, ναι αυτή είναι μια συζήτηση για τα συστήματα επίσης αποζημίωσης των επενδυτών. Εγώ είμαι διατεθειμένος να κάνουμε μια συζήτηση για το εξάντα και το εξπόστ. Πρέπει να δούμε το, το καλύτερο σύστημα ποιο είναι, αλλά συμφωνώ πως χρειάζεται χρηματοδότηση. Αρχές χρηματοδότησης έτσι, στιβαρές. δεν ξέρω αν θα πρέπει να δημιουργούμε ένα σενάριο με τα χειρότερα δυνατά συμβάντα για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κάτι τέτοιο κοστίζει πολύ. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το οποίο λέει η Επιτροπή μας και αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν. Αυτό το οποίο απαντάει. Θεωρώ πως υπάρχουν πολλά ζητήματα και ερωτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη για αυτές τις προτάσεις. Και αυτά νομίζω από μένα. Έχουμε και κάποιες τροπολογίες και πολύ ευγενικά απαντήσατε. στο παρελθόν ε, διμερός, ε, νομίζω πως θα, συνεχίσουμε και με τους άλλους σκιώδεις συζήτητες Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα για την συνένεση ε, όσον αφορά αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίγολτ ε, για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια θέματα που θα ήθελα να αναφέρω. Αν μια ασφαλιστική εταιρεία χρεοκοπήσει, για μένα δεν είναι λογικό, εάν δημιουργήσουμε ένα σύστημα αποζημίωσης, μέρος ε, της απώλειας να το καλύψει ο καταναλωτής. Αντιλαμβάνομαι τα ζητήματα ηθικού ρίσκου, αλλά ε, αυτή τη στιγμή ε, ε, συνάπτει κανείς μια σύμβαση, δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει στη σύμβαση αυτή το εάν θα χρεοκοπήσει σε 20 χρόνια αυτή η εταιρεία και θα είναι άδικο να αφήσουμε τον καταναλωτή να πληρώσει άμεσα το, το κόστος. Πράγματι τα συστήματα αυτά τελικά θα τα υπομειστεί ούτως ή άλλως ο καταναλωτής, αλλά είναι μια δίκαιη νομίζω κατανομή της ευθύνη να μην ε, υπάρχει επιπλέον κόστος για τον πελάτη μιας εταιρεία η οποία χρεοκόπησε. Αυτό δεν είναι δίκαιη κατανομή του κόστους. Και είμαι επιφυλακτικό για τις ε, τροπολογίες που προτείνονται στην έκθεσή σου, Πίτερ, που ζητούν κάτι τέτοιο. Το δεύτερο σύντημα. Αυτή η χρηματοδότηση εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, σας ευχαριστώ όλοι που είσαι διατεθειμένος να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα και διμερώς το συζητήσαμε Πίτερ. Υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα του γιατί επιλέξαμε ένα ισχυρό στοιχείο ex ante στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων των τραπεζών και γιατί έγινε το ίδιο στην έκθεσή σου για τους επενδυτές και τα ίδια επιχειρήματα στοιχείων και εδώ πέρα. Πράγματι πρέπει να ρυθμίσουμε τις ασφαλιστικές εταιρείε και η Οδηγία Περιφερειακότητας 2 αυτό φροντίζει, αλλά οι εποπτικές αρχές μας λένε πως δεν έχουμε τους πόρους να αξιολογήσουμε τα μοντέλα κινδύνου των ασφαλιστικών εταιριών. Εγώ ανησυχώ λίγο όταν βλέπω τις ε, ικανότητες ε, των ανθρώπων στις ασφαλιστικές εταιρείες σε σύγκριση με των εποπτικών αρχών. Αν αυτό συμβαίνει λοιπόν, ξέρετε, μάλλον δεν μιλάμε στα ίδια, με τα ίδια άτομα. Εγώ όταν βλέπω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, πρέπει να πω πως ε, δεν θα είναι ποτέ τόσο καλές οι εποπτικές αρχές για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Οπότε αν θα συνεχίσουν να εμφανίζονται τέτοιες περιπτώσεις, τότε το ερώτημα είναι τι είναι δικαιότερο, εξάντε ή εξπόστ. Και νομίζω πως είναι σαφέ. Εάν έχουμε μία προσέγγιση εξάντε, τότε και η ασφαλιστική εταιρεία ε, η οποία δημιούργησε το πρόβλημα έχει συνεισφέρει. Πρώτο επιχείρημα. Δεύτερον, εάν έχουμε εξωτερικούς παράγοντες που φέρνουν σε δύσκολη θέση ασφαλιστικέ εταιρείε που δεν μπορούμε να τι αναμένουμε τόσο γρήγορα. Υπήρχε όπω η τωρινή κατάσταση ας υποθέσουμε πως μεγάλες οικονομίες στην Ευρωζώνη θα έχουν προβλήματα με τα ομόλογα τους. Τότε θα βλαπτούν πάρα πολλές ε, ασφαλιστικές εταιρείε και ας είχαν σωστή διαχείριση. Οπότε τότε η συνεισφορά εξπόστ θα είναι κάτι το οποίο θα ενισχύσει τον κύκλο ο οποίο υπάρχει. Θα βλάψει ξανά τι ασθενέστερε ασφαλιστικέ εταιρείε. Αν έχουμε δηλαδή συμμετρικά σοκ σε μια οικονομία, τότε Υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα υπέρ του να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα χρηματοδοτείται εξ άντε. Και δεν βλέπω γιατί να μην ισχύσει κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Ίσχυε το επιχείρημα αυτό στι τράπεζε, μόλι τώρα έγινε η συζήτηση στην Επιτροπή μα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο διαφορετικέ οι ασφαλιστικέ. Και τέλο, για το ζήτημα τη εποπτική αρχή στην ε, οικία χώρα. Κοιτάξτε, σε μία κοινή αγορά και αν θέλουμε να έχουμε περισσότερες ε, διασυνοριακές συμβάσεις, το οποίο το θέμε για την επιλογή των καταναλωτών, τότε θα πρέπει να έχουμε παρόμοιες προδιαγραφές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε, εάν θέλετε για επιχειρήματα, για λόγους επικουρικότητας να λέτε πως θα έχουμε λίγα και πολύ, λίγες και πολύ χαμηλές ε, κοινέ προδιαγραφές, τότε δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την αρχή του οικείου κράτου. είτε έχουμε υψηλέ προδιαγραφές και τότε μπορείτε να έχετε αυτή την αρχή του οικείου κράτου. ή έχουμε χαμηλές προδιαγραφές και πρέπει να έχουμε μία εναρμόνιση. Και η, η, την αρχή αυτή της ε, επιτήρησης στο οικείο κράτος. Αυτά δεν κολλάνε μεταξύ τους. Έχουμε υπέρ του να έχουμε μια στιβαρή προσέγγιση κοινών προδιαγραφών που βεβαίως μπορεί να είναι υψηλότερε σε εθνικό επίπεδο αλλά να υπάρχει μια κοινή αγορά, κοινέ ψηλέ προδιαγραφές και μετά να συζητήσουμε την αρχή της χώρας υποδοχής αλλά το να συνδυάσουμε την οικία χώρα με χαμηλές προδιαγραφές αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα. Και τελευταία παρατήρηση και περισσότερο είναι ζήτημα ρητορίε εδώ πέρα. Πράγματι, οι ασφαλιστικές εταιρείε δεν είναι σαν τις τράπεζε, αλλά στην κρίση έκανα παρόμοια λάθη. Πολλοί ε, χρήστες, ε, τελικοί χρήστε, πελάτες ε, ασφαλιστικών εταιριών θα έχουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις γιατί ε, έγιναν επενδύσεις σε προϊόντα τα οποία δεν απέδωσαν ε, όσο αναμένονταν. Οπότε κάποια προφίλ κινδύνου επίσης είχαν ε, επεξεργαστεί με λανθασμένο τρόπο και θα το συζητήσουμε αυτό ε, και πιο πολύ στο πλαίσιο της κρίσης ε, του ευρώ. Και πολλές ασφαλιστικές εταιρείε επίσης υποφελήθηκαν από τις διασώσεις των τραπεζών, οπότε δεν μπορούμε να πούμε πως οι ασφαλιστικές εταιρείε δεν επηρεάστηκαν από την κρίση και τα λάθη που έγιναν στον χρηματοοικονομικό τομέα. Νομίζω στη διατύπωση, Πίτερ, θα βρούμε κάτι το οποίο είναι δίκαιο για τη... Ε, τις αλλά μην παριθάνουμε πως δεν έγινε κανένα λάθος κατά τη διάρκεια της κρίσης. Κυρία Λούλινγκ. Euh, ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω εν συντομία όσον αφορά τις τροπολογίες που κατέθεσα Κάποιε τι συνυπέγραψα με τον κύριο Καράς, που είναι ο εισηγητής μας, σκιώδης εισηγητής, και ο κύριος Γκοζέ ήδη αναφέρθηκε στις ε, προτάσεις. Δεν θέλω να επανέλθω στι λεπτομέρειες, αλλά θέλω να πω ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής στο καθεστώ εγγύσεω των ασφαλίσεων στα φυσικά πρόσωπα διότι η συμπερίληψη των νομικών προσώπων θα ήταν μια πηγή πάρα πολλών ε, περιπλοκών. Επίσης πρότεινα ένα όριο όσον αφορά τις αποζημιώσεις των απολειών που δέχονται. Ξέρω ότι αυτή η ιδέα δεν είναι κάτι που στηρίζουν όλοι, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει αντί αυτή η περιπτώση να θεωρήσουμε την ασφάλεια ζωής σαν μια τοποθέτηση οικονομική. Είναι μια οικονομική τοποθέτηση όπως οποιαδήποτε άλλη και, και ισχύει σε πάρα πολλά κράτη-μέλη και ξεκινώντας από αυτό Μία ανώτατο όριο, παραδείγματο χάρη στα 10.000 ευρώ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κανονικό. Και να, το να μην προβλέπουμε ένα ανώτατο όριο είναι ότι αναλαμβάνουμε συστημικό κίνδυνο για όλο το σύστημα των ασφαλιών και γι' αυτό εγώ παρακαλώ τον εισηγητή να έχει την καλοσύνη να λάβει υπόψη τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Κύριος Κίντς. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα, όλη αυτή η έκθεση καλύπτει ένα σημαντικό κενό, γιατί όλοι είπαν ότι έχουμε 20 διαφορετικά καθεστώτα σήμερα στην Ευρώπη. Η δική μου εξέταση 12 διαπίστωσε, μαζί και με τον οικονομικό, χώρο ελεύθερων οικονομικών συναλλαγών. Χρειαζόμαστε, πιστεύω, όταν προσπαθούμε να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, ένα σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένο πεδίο ε, και γι' αυτό δεν συμφωνώ όπως ε, προτάθηκε η εξάντε χρηματοδότηση ως πρόσθετη δυνατότητα να λειτουργεί. Πρέπει ένα ενιαίο πλαίσιο να διασφαλιστεί. Δεν είμαι τόσο θετικός ε, όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείε ε, όπως ο φιλελεύθερο συνάδελφο ε, Όλε Σμιτ. Έχω βιώματα και εμπειρίες ε, από την πρόσφατη εμπειρία μου έγινε μια διάρρηξη στο διαμέρισμά μου στις Βρυξέλλες και επειδή ευτυχώ δεν είχα τι μαλφή ή μετρητά δεν πήραν τίποτα ακόμα και τα ποσά ήταν εκεί απλά την πόρτα εισόδου κατέστρεψαν σε παρέμβαση χωρί μικρόφωνο σίγουρα ναι έπρεπε να αντικαταστήσω την είσοδο και παρόλα αυτά πίστεψε η ασφαλιστική εταιρεία να μην, ότι δεν χρειαζόταν να παραναπληρώσει ε, κάτι ε, όσο, όσο το ίμιση, το μισό του ποσού ως φορφετέ, ως ε, καταποκοπήν ποσό. Βλέπετε ότι αυτή είναι η κατεύθυνση των ασφαλιστικών εταιριών από πλευράς ε, νοοτροπίας. Δεν πρέπει εδώ να λαμβάνουμε λανθασμένα υπόψη τα συμφέροντα εταιριών και αυτά τα οποία επιβάλλονται για την προστασία καταναλωτών να λειτουργήσουν σωστά. Το ότι δεν μπορεί να πτωχεύσει τόσο ξαφνικά μια ασφαλιστική εταιρεία στην Μανχάιμερ είχαμε μια υπερβολική δράση σε συγκεκριμένο είδος ε, συναλλαγών, όμως για την ε, ε, equity, life equity βλέπουμε ότι έγινε η αντίστοιχη αυτή περίπτωση, πτώχευσε και δεν έχουν πάρει τα, τις αποζημιώσεις οι πελάτες ε, μέχρι σήμερα. Θα έλεγα ως συμπέρασμα, ας προσπαθήσουμε το δυνατόν να καταλήξουμε σε εναρμονισμένες δομές για το σύνολο της Ευρώπης και να μην έχουμε πάλι αυτές τις εναλλακτικέ δυνατότητες απελευθέρωσης ή εξαίρεσης κάθε χώρα να έχει κάτι ξεχωριστό για το επίπεδό της. Δεν θα έχουμε έτσι ένα ισοδίκαιο πεδίο δράσης και η διαφοροποίηση μεταξύ ασφαλίσεων ζωής ή διαφορετικών ασφαλίσεων είναι κάτι το οποίο επανειλημμένα προ προαναφέρθηκε δεν θα πρέπει εδώ να έχουμε ε, στεγανά. Μεταξύ τώρα ε, κράτους υποδοχής και ε, κράτους θηγατρικού υποκαταστήματος. Συμφωνώ με αυτά, όμως Life έδειξε ότι αυτά δεν λειτουργήσαν σωστά στο παρελθόν. Δεν υπήρξε συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας. Δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι αυτόματα όλα αυτά επιλύονται ως διαμαγείας. Χρειάζονται χρόνο για να επιληθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα λάβει τον λόγο εισηγητής μας τώρα για να κάνει κάποια σύντομα σχόλια από πλευράς του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Και βλέπω πως υπάρχει έντονη συζήτηση, αλλά νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ανεξαρτήτως βέβαια στο ότι κάθεστε εσείς οι δύο δίπλα και δεν μπορείτε να συμφωνήσετε, θα συμφωνήσουμε. Κοιτάξτε, αυτή είναι η έκθεση ίδιας πρωτοβουλία, αλλά είναι μια δήλωση. Το τι κάνουμε, ποια επιχειρήματα αναπτύσσουμε για το ότι η Κομισιόν θέλει να ε, κάνει κάτι σε ολόκληρη την Ένωση χωρίς να μας ρωτήσει. Οπότε συμφωνώ πως ε, ελπίζω να μας ακούσουν όσον αφορά την στιβαρή μας ε, προσέγγιση. Τώρα για αυτό το οποίο είπε ο Ζανπολ. Κοίταξε, ο Ότμαρ μάλλον κάπου απαντάει το τηλέφωνο του όπου και αν είναι, οπότε θα είμαστε σε επαφή γιατί είναι σημαντικό και, το, και η διασυνοριακή πτυχή, πράγματι για τα αυτοκίνητα, ασφάλιση αυτοκινήτων, υγεία ζωής κτλ. Όπου και αν πάει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, η ασφάλεια θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής. Οπότε κάπου πρέπει να έχουμε ε, κάτι το οποίο θα υπάρχει μια εγγύηση για, για το ότι οι συμβάσεις αυτές, γιατί είναι συμβάσεις σε αντίθεση με τις τραπεζικές συναλλαγές, πως ε, οι συμβάσεις αυτές θα τηρηθούν. Όλα η διαφορά μεταξύ ζωής και μη ζωής, λες πως εσύ θέλεις συγκεκριμένους λόγους για το γιατί θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογή, να το δούμε αυτό. Δεν νομίζω πως ε, θα είναι βλακώδες, απλά θα είναι λάθος να αποκλείσουμε τον κλάδο, τους κάλους κλάδους πλήν ζωής. Ας δούμε το πώς βλέπουν οι ρυθμιστικές αρχές αυτά τα ζητήματα. Ξέρουν πως υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα για αντιμετώπιση του κινδύνου στον κλάδο ζωής και στους υπόλοιπους. Υπάρχουν υπολογισμοί, το χρησιμοποιούσαμε στην ε, φερεγγιότητα 2. Καλύτερα αυτό να κάνουμε αντί να το αποκλείσουμε για να υπάρχει ένα συμβασμός με αναλογικότητα. Αλλά δεν, δεν, θα... δεν είμαι υπέρ του να αποκλείσουμε στοιχεία του κλάδου αυτή τη στιγμή. Τόσο θα πρέπει να το συζητήσουμε. Επίση. Ε, για τα εμπόδια. βεβαίω ε, δεν θέλουμε να εμποδίσουμε κανένα να αγοράσει ασφάλιση και βεβαίω ε, όσο πιο ακριβή γίνεται και κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει την ασφάλεια, τότε μεταβάζονται στην κοινωνία το κόστος. Γιατί αν καίγεται το σπίτι σου και εσύ δεν έχεις ασφάλεια και καίγεται και το σπίτι του γείτονά σου, πλέον έχουμε ένα, μια καταστροφή και δεν ξέρω, ίσως και συστημικό κίνδυνο τέλος πάντων. Ναι, ναι, μπορεί. Λοιπόν, κατα... μπορεί να πληρώσουν οι καταναλωτές σε τελική ανάλυση, δεκτό αυτό που λέτε, πράγματι, αλλά δεν θα πρέπει να μην προστατεύουμε τους, τους καταναλωτές, να υπάρχει μια αναλογικότητα για να μπορούν και οι εταιρείε να λειτουργήσουν και να είναι εξασφαλισμένοι και οι καταναλωτές. Σβέν, για το θέμα της χώρας προέλευση. Σημαντικό, αλλά όπως είπε και ο Βόλφ, που λέει πως στην Equitable Life δεν υπήρχε επιτηρήση, πράγματι απέτυχε εκεί πέρα το σύστημα και πρέπει να πούμε πως το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ε, και η χώρα προέλευσης ε, και ε, χώρα υποδοχής ε, και εκεί πέρα υπήρχε μια δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς ρύθμιση με τρόπο που στη Γερμανία δεν ε, ε μπορούσε. Βεβαίως τώρα αυτά τα έχει λύσει η οδηγία Φερικιότητα 2. Οπότε εγώ θα θεωρώ πως αυτό θα είχε αντιμετωπιστεί τότε. Δεν επαρκούσε αυτό το οποίο προϋπήρχε και άρα η Equitable Life έχει σημειωθεί νομίζω, έχουμε σημειώσει την πρόοδο που έχει γίνει τώρα. Έχουμε τους συλλογικού φορείς, ε, έχουμε την δυνατότητα επιβολής, οπότε δεν εφευρίσκουμε ξανά τα ίδια πράγματα. Ας το δούμε λοιπόν πριν προσθέσουμε τίποτα άλλο και να γίνει μια συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ να ξεκινήσω μια συζήτηση, αλλά νομίζω πως πρέπει να δούμε τα έγγραφα εδώ πέρα ε, του επίπεδου 1 δεν χρειάζεται νομίζω να κάνουμε τίποτα άλλο. Τέλος, κανείς νομίζω δεν είπε χαμηλές προδιαγραφές, ε, είπαμε ελάχιστες προδιαγραφές. Αυτό λέω εγώ, αυτό σημαίνει πως μπορεί κάποιος να προσθέσει. Και μπορεί να έχει βεβαίω και τα ελάχιστα, αλλά πραγματικά και αυτό επιτρέπεται και πρέπει να σκεφτούμε ε, εάν είναι να επιτρέψουμε την ανάπτυξη κάποιων συστημάτων προστασίας σε κάποια και σκεφτείτε παραδείγματο χάρη τι γίνεται με τις ε, ε, αμοιβέ ε, ασφαλής π.χ. στη Γερμανία εάν πάμε για μάξιμου εναρμόνιση σκεφτείτε τι συνέπειες θα έχει αυτό θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες να σας δώσω ένα παράδειγμα Κοιτάξτε, στις ε, τράπεζες κεφάλαιο επίπεδου 1 είναι κεφάλαιο, αλλά στις ασφάλειες ε, δεν είναι, ε, μετρητά, με αλλά στις ασφάλειες δεν είναι. Σκεφτείτε το αυτό. Γιατί οι συνέπειες των πραγμάτων που λέμε μπορεί να είναι πολύ σοβαρές σε αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε ως διασφάλιση. Σκεφτείτε το τι μπορεί να, να γίνει. Το ίδιο και η Σουηδία όλε. Α, μπράβο. Οπότε σκεφτείτε το λίγο αυτό. Caps and ceilings. Για τις οροφές, τα πλαφόν, Αστρίντ, εσύ πρέπει να είσαι πιο εξαιρετική εδώ μέσα, οπότε ε, καλύτερα να μην σου πω όχι γιατί είναι και ο συντονιστής σου εδώ πέρα. Θα το σκεφτούμε αυτό. Ε, μη με κοιτάς έτσι, σε παρακαλώ. Θα δούμε τι μπορούμε να, να κάνουμε. Αλλά νομίζω πως αν έχουμε έτσι μια συνολική προσέγγιση και του τι έχουμε κάνει και σε άλλες εκθέσεις, νομίζω πως θα μπορέσουμε να απαντήσουμε παρκώς στην Κομισιόν. Για την υπόθεση εξάντε Ex-post. post. Εδώ πέρα νομίζω θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποια συμβαστική λύση. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ του εξάντε και όταν είσαι σε μια χώρα που έχει ε, ούτως ή άλλως ε, αρκετές ε, τέτοιες επιχειρήσεις και απειλείται ο φορολογούμενος και τελικά δεν θα υπάρχει ο κλάδος για να πληρώσει τελική ανάλυση και έχουμε δει πολλά τέτοιες περιπτώσεις τώρα πρόσφατα θα πρέπει να πούμε πως η εξάντα χρηματοδότηση είναι ο μόνος τρόπος αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να πούμε εκεί όπου υπάρχει λιγότερος ε, κίνδυνος μπορούμε να πούμε πως ε, μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα με περισσότερες έτσι, αποχρώσεις. Δεν είναι ανάγκη όμω να περνάει όλο το κόστος συνεχώς στον ε, καταναλωτή. Αν είμαστε λοιπόν έξυπνοι νομίζω θα βρούμε την, ε, τη λύση που βρήκαμε. Δεν σα θύμωσα εγώ και φεύγετε ελπίζω. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ενδελεχή συζήτηση από αυτού. Και εις βάθος απαντήσει του συγητή. 24 Μαΐου ψηφίζουμε. Και θα πάμε στην Ολομέλεια ενδεχομένω στη δεύτερη σύνοδο του Ιουνίου. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε καθυστερημένα να προβεί σε κάποια σχόλια όσον αφορά τα σχήματα εγγύσεως καταθέσεων. Ξέρω ότι συζήτησε κάποια τα θέματα με τον συγγετή, τον κύριο Σάιμον. Δεν θα σας στερήσω τη δυνατότητα να προβείτε σε σύντομο σχόλιο, πρέπει να είναι σύντομο, διότι έχουμε μείνει κάπως πίσω. Κυρίως αν θα υποστηρίξετε την θέση της Επιτροπής και το έργο του εισηγητού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε επιτρέψω να σχολιάσω και τα δύο θέματα. Ασφάλειες ε, και το σύστημα για την κάλυψη των καταθέσεων. Ασφαλίσεις και Σκίνερ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Εκτιμώ αυτά που είπατε για το βασικό ρόλο της ασφάλειας για να εξασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση των ατόμων. Το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το λαμβάνουμε υπόψη στη φιλοσοφία Φία μας. Το πνεύμα της Λευκής Βίβλου ήταν ακριβώς αυτό να υποστηρίξει όλους εμπλεκόμενους και να ζητήσουμε την αντίδραση των εμπλεκομένων φορέων. Θα σας διαβεβαιώσω ότι θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά αυτά που προτείνετε. Σαφώς η αναλογικότητα είναι η βασική λέξη εδώ, είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα εξετάσουμε το θέμα της ζωής μη ζωής και θα εξετάσουμε και τις διαφορές μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζών. Κάποια σημεία έχω τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν θέλουμε να κάνουμε καλή δουλειά. Το, άλλο, το ένα είναι εκ των προτέρων, το Α μην ξεγελιόμαστε εκ των υστέρων, είναι προκυκλικό. Ε, μπορούμε να έχουμε κάποια ευελιξία εκ των προτέρων όσον αφορά τι λεπτομέρειε. Αλλά να αμφισβητεί κανεί την αρχή του εξάντε, το εκ των προτέρων, είναι κάτι το οποίο ίσω να θεωρηθεί από αρκετού σαν μη επίλυση του θέματος. Δεν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε το σύστημα, που Αντιθέτως, να το κάνουμε όσο πιο ισχυρό γίνεται και καλωσορίζω αυτά που είπατε και σίγουρα θα εργαστούμε επί των θεμάτων αναλογικότητας. Για το DGS, ναι κυρία Πρόεδρε, ε, στερνίζομαι την έκθεση όσον αφορά τις εγγύσεις των καταθέσεων. Το είπα προηγουμένω Έχω έξι σύντομε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα άκουσα διαφόρου οι οποίοι συσχέτισαν το σύστημα αυτό των καταθέσεων, την Βασιλεία και τη διαχείριση των κρίσεων. Βεβαίω πρόκειται σχέσει, πρέπει να γίνει σχέση. Έχουμε περισσότερα κεφάλαια στι τράπεζε, άρα η τράπεζα αυτή καθεαυτή γίνεται ασφαλέστερη. Με τον Καρσία Μαγκάιο και την κυρία Φεραίρα επεξεργόμαστε ένα πλαίσιο διαχειρίσεω των κρίσεων. Ελπίζουμε να αποφύγουμε επηρεασμό τη οικονομία. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και γι' αυτό μπορούμε να έχουμε μόνο 1,5% καταθέσεων κάλυψης. Α μην κάνουμε διπλά λογιστικά επειδή είναι ασφαλής και 1,5% αρκεί διαφορετικά θα χρειαζόμασταν πολλά περισσότερα. Δεύτερον, άκουσα επανειλημμένα κάτι που, ε, για το οποίο λυπάμαι. Πολλοί είπαν ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέταζε μόνο την αρχή του συστήματος Paybox. Κάνουμε, είναι σφαλμένο. Εμείς είχαμε περισσότερα από το Paybox αναφέραμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ξεπεράσουν το paybox. Παρ' όλα αυτά, δοθέντως ότι πολλοί κατάλαβαν κάτι διαφορετικό, εκδώσαμε και διευκρινιστικό έγγραφο ε, πριν από ένα μήνα περίπου, όπου εκεί καταστέσαμε σαφέστατο ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ξεπεράσουν και να λάβουν τις προ, ε, προληπτικές δράσεις που απαιτούνται. Εδώ όμως με την έκθεση. Όσον αφορά εκ των υστέρων και των προτέρων, ε, το είπα και στην περίπτωση των ασφαλιστικών, δεν νομίζω ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τίποτα υπερκυκλικής ακολουθώντας τον κύκλο και θα πρέπει να έχουμε τακτικές εκθέσεις όσον αφορά την κυκλική, ε, τον κυκλικό επηρεασμό των κανόνων. Μετά το χρόνο πληρωμής υποστηρίζουμε πλήρως ε, αυτό που λέμε ένα σχήμα το οποίο να δίνει κίνητρα διότι δίνοντας την επιλογή 5 μέρες ή 20 μέρες ε, δίνει τη σωστή έμφαση. Δεν θα πιστεύετε πόσε τράπεζε ήρθαν και μου είπαν πέντε μέρε κανένα πρόβλημα και δεν ήταν οι μεγαλύτερε. Οπότε, αν κάποιε τράπεζε μπορούν να το κάνουν σε πέντε μέρε, πολύ καλά. Όσον αφορά το κίνδυνο, πολύ καλό να διευρυνθεί το πλαίσιο. Μπορούμε να βάλουμε επιδιώμηση, διαφοροποίηση, μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Ίσως θέλετε να προχωρήσουμε παραπέρα, να θυμόμαστε όμως ότι αυτό δεν είναι καθημερινή εποπτική προσέγγιση, εποπτικό εργαλείο. Αφορά ένα μέτρο μία, μία φορά την, το χρόνο εφαρμόζεται. Δεν έχει σαν στόχο ε, το κίνδυνο να το μειώνει. Διότι είναι επικίνδυνη συμπεριφορά του χρόνου πάει η τράπεζα. Θα μπορούσαμε να το διευρύνουμε, αλλά μην θεωρούμε ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Τέλος, ε, νόμισμα αποζημίωσης πληρωμών ε, προσμετίζεται τις δύο εναλλακτικέ. Το είπατε, Πρόεδρε. Καταναλωτέ διαλέγουμε. Ο καταναλωτέ ε, χρησιμοποιεί ένα νόμισμα για τι καταθέσει. Ο... Αν πάρει άλλο νόμισμα, παίρνει τον κίνδυνο ο καταναλωτή. Μετά αναφέρθηκε από τον κύριο Σίμων χρόνο, πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει η αλλαγή του νομίσματο. Ίσως σε πέντε λεπτά αλλάζουν κάποια νομίσματα και να πληρώσει, άλλα όχι. Άρα πρέπει να μετρήσει κανεί τα δύο αυτά πράγματα και βεβαίω είναι ένα σήμα αυτό, μήνυμα που στέλνει προ εκείνον που θε να προστατεύσει, να τι προστατεύσει του καταναλωτέ είτε όχι. Και τέλο, χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει υποστήριξη για ένα νέο σχήμα. Ε, είδα κάποιες δηλώσεις επί των αρχών που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Πολύ καλό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλωσορίζει αυτό. Λυπούμε που η πρόταση για τη δανειοδότηση από τα μηδέα που ήταν η πρώτη πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση δεν υποστηρίχθηκε ούτε εδώ ε, ούτε σε άλλα βήματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα σχόλια. Είμαι σίγουρη ότι θα ληφθούν υπόψη. Θέλω να προχωρήσουμε γρήγορα και να πάμε στι δύο τελευταίε συζητήσει, τα δύο τελευταία θέματα τη ημέρα. Ναι, συμφωνείτε λοιπόν συνάδελφοι, αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερο χρόνο στους ε, εισηγητές ε, και λίγο λιγότερο στους σκιώδεις. Γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στις τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα δώσω λόγο στον κύριο Χέκμαρκ για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έχω υποβάλει την έκθεσή μου, το σχέδιο έκθεσης και έτσι έχω ήδη λάβει διαφορετικές απόψεις ε, και προτάσεις ε, για αυτό. Θα έλεγα μια από αυτές τις μέρες ε, όταν θα έχουμε σε σχέση με την αξιολόγηση του βάρους ε, είναι πολύ σημαντικό πόσο είναι μεγάλη η εξάρτηση, αλληλεξάρτηση των οικονομιών μας μεταξύ τους, διότι ό,τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ θα είχε επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική εξέλιξη των πραγμάτων σίγουρα και το πώς αντιμετωπίζεται το έλλειμμα ή η νομισματική πολιτική είναι εξίσου σημαντικό όπως είναι σημαντικό πόσο, ε, πώς αντιμετωπίζουν οι Κινέζοι το νόμισμά τους. Η ανάγκη λοιπόν για την παγκόσμια διακυβέρνηση είναι ανάγκη να στοχεύουμε σε ρεαλιστικούς στόχους και αλλαγές που είναι εφικτές. Ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε μια συζήτηση για όλα αυτά είναι η ανάγκη να υπάρξει κάτι που θα είναι καινούριο και θα αναζωογονήσει τις δομές που έχουμε και που δημιουργήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα τρία τελευταία χρόνια είδαμε αυτή την ανάγκη που υπάρχει για μεταρρύθμιση των παγκόσμιων αυτών θεσμικών δομών. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι καμιά φορά υπάρχουν και πολλές ελπίδες ότι μια νέα παγκόσμια διακυβέρνηση αν υπάρξει θα επιλύσει όλα τα προβλήματα. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο βέβαια. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι αποτέλεσμα τεράστιων οικονομικών αλλαγών που γενικά καλωσορίζουμε. Τα τελευταία 25 χρόνια η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε υπερβολικά, ιδιαίτερα γρήγορα και έχοντας ένα δισεκατομμύριο παλιότερα που ζούσαν σε σχετική ευημερία, τώρα έχουμε τέσσερα δις που ζουν σε σχετική ευημερία και για τις ε, παγκόσμιες ανισότητες ε, για τις οποίες γίνεται λόγος είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων και αλλαγών και ελλείψεις και ελληματικές καταστάσεις των παλαιών οικονομιών, μεγάλων οικονομιών να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και γι' αυτό πολλά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εξαρτώνται από τις δομές, ε, της ελλείψεις και προβλήματα που υπάρχουν ε, λόγω της παλαιάς τάξης των πραγμάτων, οικονομικής τάξης πραγμάτων, που ήταν εκείνη που επικρατούσε παγκόσμια οικονομικά. Αυτά που βλέπουμε φυσικά είναι η ανάγκη να συζητηθούν τα ελλείμματα υπό παγκόσμια προοπτική, αλλά επίσης και οι, εποπτείες, οι πολιτικές επιτήρησης και εποπτείες. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στις συζητήσεις για νομίσματα είναι ότι κάποιες οικονομίες, κυρίως η ΕΠΑ, έχουν μια πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική με σημαντικές επιπτώσεις για τις αναδιόμενες ε, οικονομίες των αναδυόμενων χωρών και διαφορετικά μέτρα για τα νομίσματα και τον έλεγχο αλλά επίσης ε, και προστατευτικές ε, ρυθμίσεις και διατάξεις. Γι' αυτό η λέσχη των 20 G20 ιδιαίτερα κατά την έναρξη της κρίσης διαδραμάτισε κέριο ρόλο διότι αυτό που έκανε ήταν έκανε, έδωσε τη δυνατότητα στην παγκόσμια κοινότητα εθνών να επικεντρωθεί σε σημαντικά προβλήματα για την ανάγκη υιοθέτησης ταχείας δράσης, αλλά επίσης και για συμφωνίες ε, που θα έπρεπε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ώστε να μην υπαναχωρήσουν σε προστατευτικά αιτήματα και δράσεις οι κυριότερες οικονομίες. Ε, και καταδείχθηκε ότι υπήρξαν αποτελεσματικές δράσεις διότι πολλές αποφάσεις που ελήφθησαν είχαν τη σημασία τους, τη σπουδαιότητά τους. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές από αυτές τις αποφάσεις δεν εφαρμόζονται, δεν υλοποιούνται πρακτικά στην καθημερινή πρακτική και υπάρχει έλλειψη σταθερότητας όσον αφορά τις παγκόσμιες δομές ε, στη διάρθρωσή τους. Γι' αυτό η έκθεσή μου υπογραμμίζει τη σημασία το, της λέσχης των 20 ως ενός παγκοσμίου βήματος, φόρουμ για τέτοια παγκόσμια διαβούλευση. Τίνω περισσότερο να πω ότι τα ε, θεσμικά όργανα, Παγκόσμιο ε, ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να είναι ο πυρήνας ε, της παγκόσμιας διαχείρισης και διακυβέρνησης και η λέσχη των 20, G20 πρέπει να συνδέεται πολύ περισσότερο με τη σταθερότητα και διαθεσμική θεσμική δομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όταν προσπαθούμε να προχωρήσουμε και να περιγράψουμε πώς αυτή η παγκόσμια διακυβέρνηση θα πρέπει να λειτουργεί και να αποφασίζεται, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της εποπτείας και της παρακολούθησης νομισματικών πολιτικών, συναλλαγματικών πολιτικών, την ανάγκη να συζητούμε τα διαθροτικά ελλείμματα και τις επιπτώσεις του στις άλλες οικονομίες και για το πώς θα επιτύχουμε μια κοινή επαγκοσμιοποιημένη ε, σταθερότητα. Για όλα αυτά τα προβλήματα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να είναι διότι είναι περισσότερο, λογοδοτεί περισσότερο και είναι περισσότερο παγκοσμιοποιημένο από θεσμικής πλευράς από ότι η λέσχη των 20. Και βλέπουμε εδώ σε σχέση με την ε, παγκόσμια προσέγγιση για την παγκόσμια διαχείριση πρέπει υπό αυτό το πρίσμα να αντιμετωπιστεί. Συνολικά θα έλεγα ότι θα έπρεπε όλο και περισσότερο να συζητούμε πώς θα μπορέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι η καρδιά, ο πυρήνας της λειτουργίας της παγκόσμιας διακυβέρνησης οικονομικά. Επαρκούμε σε αυτά για να κερδίσουμε χρόνο. Ευχαριστώ. Ε, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ο κύριος εδώ πέρα νομίζω πως έχουμε ένα αρκετά καλό έγγραφο και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χόκμαρ πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Αλλά νομίζω πως οι βασικοί στόχοι υπάρχουν. Εάν αναρωτηθούμε τι θέλουμε πραγματικά από αυτό το έγγραφο ιδίας πρωτοβουλίας, πρώτα απ' όλα πρέπει να ενισχύσουμε την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε οικονομικά ζητήματα, γιατί πρέπει να μιλάμε με μία φωνή. Στο παρελθόν, όπως ξέρουμε, κάποια κρατημέλη είχαν πολύ ισχυρή φωνή και συμφέροντα στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, ιστορικά μιλώντας, αλλά τώρα πρέπει να έχουμε μία φωνή και για να γίνει αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την εξωτερική εκπροσώπηση στα ζητήματα αυτά. Μετά, αν γίνει αυτό, προφανώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ηγητικό ρόλο, η Ένωση συνολικά, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, στις παγκόσμιες μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να αξιολογήσουμε επίσης ξανά τη σύνθεση των G20. Δεν ε, είμαι επικριτικός για τους G20 τελευταία, ε, πάνε αρκετά καλά, αλλά επειδή ε, εξαρτάται η σύνθεση, νομίζω πως πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση του εάν εκπροσωπεί τους μικρούς και τους μεγάλους, ισχυρούς και τους ανισχυρούς. Να δούμε εάν ε, εκπροσωπούνται αρκετές χώρες. Πρέπει να θυμόμαστε πως έχει αλλάξει το οικονομικό τομείο, αυτό είναι προφανές με την Κίνα και την Ινδία κτλ. Οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο ήταν. Αν θυμάστε το, το Μπέρτον Γουτζ, οι ισχυρέ χώρε ήταν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΠΑ και ότι έλεγαν και συμφώνησαν. Ε, ήταν απλό, αποτελούσε και τη συνένεση το 1945, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα, αυτού, τα θεσμικά όργανα. Μιλάω τώρα για το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το Δούνο του. Να παραμείνουν ανεξάρτητα, αλλά να ξέρουμε πώς θα αντικατοπτρίζεται εκεί το παγκόσμιο τοπίο για να αντικατοπτρίζει τις σημερινές πολιτικές πραγματικότητες. Τώρα, όταν μιλάμε για θέματα έχουμε πολλά. Διεθνή ρευστότητα, είναι η δεν είναι. Εάν είναι επαρκή ποια είναι η ισορροπία. Όσον αφορά το δολάριο. Το παλαιότερο ερώτημα όλων, εάν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εθνικά νομίσματα ω αποθεματικά. Ε, είδατε η αλλαγή που έκανε σαν αρκεπόρους για τις προοπτικές της αμερικάνικης οικονομίας ε, τράνταξε τα, τα θεμέλια του δολαρίου και μετά έχουμε τις δομικές ε, ανισορροπίες. Και εδώ είναι το σοβαρότερο, γιατί το βλέπουμε και εντός της Ευρωζώνης, που είναι τόσο δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε πως είναι πρόβλημα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και αυτό επαναλαμβάνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, το θέμα της ρύθμισης, καθώς οι εταιρείε είναι παγκόσμιε, αλλά όχι οι ρυθμιστικέ αρχέ. Και συνεργαζόμαστε βεβαίω ε, ε, σε υπερατλαντικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν κάποιε προδιαγραφέ ε, ελέγχου, αλλά νομίζω πως οι G20 θα πρέπει να αναθεωρήσουν παραδείγματο χάρη δημοσιονομικούς κανονισμούς και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και να δούμε αν αυτό δημιουργεί προβλήματα ή όχι αν υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές που έχουν σημασία όταν μιλάμε για την ρύθμιση. Οπότε νομίζω πως ε, έρχεται σε πάρα πολύ καλή στιγμή αυτό το θέμα εδώ πέρα. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό. Αν και πρέπει να τα δεχτώ πως κάποιοι θεωρούν πως είναι ακαδημαϊκό το ζήτημα και σέρνεται εδώ και χρόνια αλλά νομίζω πως έχει φτάσει η στιγμή δεν είναι πλέον κάτι το έτσι, απόκριφο που αφορά λίγους γιατί μπορεί να α, δημιουργήσει προβλήματα α, ίσως στις χώρες μας αλλά ξε, εμείς ξέρουμε πως το οικονομικό αυτό τσουνάμι και η κρίση ξεκίνησε από οικονομικές ε, ανισορροπίες. Ελπίζω λοιπόν η έκθεση αυτή να έχει τη σημασία της και αναμένω βεβαίως να συνεργαστούμε και να προτείνουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Χίμνα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρία σημεία μόνο. Θα έλεγα ότι η κρίση, σαφώς και ο Γκούναρ έκανε λόγο γι' αυτό, αποκάλυψε όλες τις ελλείψεις, ε, όλα τα στοιχεία που απουσίαζαν και την ε, έλλειψη αρμοδιότητας και οδήγησε σε αυτή την κατάσταση όπως ε, την εμπλοκή των G20 και των νέων εμπλεκομένων. Σε σχέση με αυτή την πτυχή η αναφορά είναι πολύ σημαντική, διότι έχουν το προτέρημα να είναι πολύ πραγματιστικοί και ρεαλιστικοί και πολιτικά να λαμβάνονται υπόψη εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα και δεν συμμετείχαν στο παρελθόν. Αλλά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία, ένα κοινό όραμα και δεν συμβαίνει αυτό σήμερα. Θέλω στην πρώτη μου παρατήρηση να τονίσω ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα θεσμικά όργανα και πώς μπορούν να βελτιωθούν, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Δεύτερη παρατήρησή μου. Υπάρχει έντονη επικέντρωση στο γενικό πλαίσιο που πρότεινε ο Κούναρ Χέκμακ να αντιμετωπιστούν οι πτυχές εξάντε και εξπόστο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Διακυβέρνηση που χρειάζεται λόγω των παγκόσμιων ανισοτήτων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης όπως πιστεύω ότι χρειάζεται η παγκόσμια διακυβέρνηση επειδή οι αγορές, οι παγκόσμιες αγορές χρειάζονται κανόνες, κανονισμούς και διατάξεις. Αυτή η θεσμική συστημική πτυχή είναι πάρα πολύ σημαντική όπως πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτή όπως όπως και στο σχεδιασμό της παγκόσμιας διακυβέρνησης αυτού του συστημικού ε, συντελεστή του στοιχείου που χρειάζεται για τις παγκόσμιες αγορές και χρηματοοικονομικές αγορές. Και το άλλο σημείο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι το ότι φαίνεται ότι υπάρχουν έντονοι σημαντικοί παράγοντες αλλαγών που λειτουργούν όσον αφορά το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα και κάποιοι θα βλέπαν και θα έλεγαν ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα που αναδύεται. Εδώ είναι λοιπόν το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρωθούμε και να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις προτιμήσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναδυόμενη αυτή δυνατότητα ενός παγκόσμιου νομισματικού συστήματος. Ευχαριστώ. Σύντομο σχόλιο έχω. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Ικλούν και η Ντανούτα και διάφοροι πριν από αυτό. Οι G20 όταν ξεκίνησαν ξεκίνησαν καλά, ήταν αποτελεσματικοί και είχαμε πολύ μεγάλες ελπίδες. Τώρα αισθάνομαι ότι αυτές οι ελπίδες ε, κάπως ξανεμίζονται διότι μετά την κρίση στα μάτια πολλών έχει μειωθεί η κρίση, είναι λιγότερο οξία και επικρατούν τεχνικά συμφέροντα. Το σημαντικό είναι να βρούμε κάποιους επίσημους τρόπους αναδιοργάνωσης των G20. Χρειάζεται κάποια μορφή, κάποιο σχήμα, επίσημο σχήμα που να αποφασίζει επιδεσμευτικών μέτρων. Αυτό που έχουμε τώρα είναι άτυπε συζητήσει, ομάδε συζητήσεων. Συναντώνται, τα περνάνε καλά, διασκεδάζουν, ανταλλάσσουν απόψει, αλλά δεν δεσμευτικέ οι αποφάσει. Χρειάζεται κάποια δεσμευτική χρειάση στι αποφάσει. Δεύτερον, εφόσον είμαστε Επιτροπή Κρίσης και ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, τώρα που ετοιμάζουμε τελική μας έκθεση, και εμείς ασχολούμαστε με αυτό, θα σου ζητούσα Γκούναρ να συμμετάσχει συζητήσεις όταν θα ετοιμάζουμε τελική μας έκθεση. Στέλνουμε το ίδιο μήνυμα όπως και στη δική σου έκθεση. Δεν θα πρέπει να έχουμε διαφορετικά μηνύματα που βγαίνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ίδιο θέμα και το ίδιο ζήτημα. Ευχαριστώ. Ξανά στον εισηγητή θα δώσω το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κ. Χόκμαρκ. Πολύ σοφά και συγκεκριμένα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μια διαδικασία του ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή φωνή στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Λυσμονούμε και ότι η μεγαλύτερη οικονομία στην, ε, στον κόσμο δεν είναι η ΕΠΑ, η Κίνα, αλλά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πρόβλημα, είναι λάτωμα το ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό στο παγκόσμιο προσκήνιο. Άρα ζητούνται διάφορες ε, μεταρρυθμίσεις που αφορούν και την οικονομία μας. Αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να επηρεάζουμε τα τεκτενόμενα. Δεύτερον, όσο μιλάμε για τον έλεγχο των G20 και να γίνουν πιο υπεύθυνοι και πιο διαφανείς και πιο επίσημο σχήμα όσο, τόσο πλησιάζουν το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο στην πραγματικότητα διότι πρόκειται περί παγκόσμιου οργανισμού εν αυτή τη ενία είναι επίσημος θεσμός καλύπτει όλες τις οικονομίες η G20 έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Αλλά οι τελευταίες συναντήσεις τους δεν κατέληξαν κάπου. Όχι μόνο οι δεποφάσεις τους δεν δεσμευτικές, αλλά και για άλλους λόγους. Μην λησμονούμε ότι οι G20 μπορεί να γίνουν G5 αύριο ή G25. G25 εξαρτάται από τις υγου... κυβερνήσεις που ηγούνται τι θα κάνουν. Και αν δείτε τον κατάλογο των προσκλήσεων που απευθύνουν, είναι τυχαίος και αυθαίρετος κατάλογος. Άρα δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτούς, αν θέλουμε να έχουμε έναν επίσημο διαφανή θεσμό. Συμπεραίνω λοιπόν ότι πρέπει να εστιαστούμε επί των σημαντικότερων στόχων όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση. Χρειάζεται, χρειάζονται κοινοί κανόνες για τις χρηματοπιστωτικέ αγορές. Κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής, διαθωτικών ελλημάτων, νομισμάτων. Θα προσθέσουμε και τα πάντα σε αυτό. Όσο πιο πολλά προσθέτουμε, τόσο πιο πολύ θα υπονομεύουμε τις δυνατότητες να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και φυκτό. Γι' αυτό να υπογραμμίσω στους συναδέλφους ότι πρέπει να είμαστε εστιασμένοι στην προσέγγιση μας. Όλα τα σχόλια που παρέλαβα ευθυγραμμίζονται με αυτό. Είναι σημαντικό να είμαστε πραγματιστές. Οι δεμοί δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, δεν θα επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα. Όσο πιο ελεγχόμενος, δεσμευτικός είναι ο φορέας αυτός διαφανής, ο φορέας G20 τόσο πιο πολύ πλησιάζουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτό να το έχουμε υπόψη μας καθώς προχωρούμε. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Να υπενθυμίσω 10 Μαΐου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Θα ξανασυζητήσουμε στις 14 Ιουνίου τις τροπολογίες. Άρα έχετε χρόνο για να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας. Πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ε, συνεδριάσεώς μας η έκθεση τη κυρία Εσάια, τεχνικέ απαιτήσει για τι μεταφορέ πίστοση και τι άμεσε χρεώσει σε ευρώ και την τροποποίηση του κανονισμού ΕΚ 924-2009. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη στην παρουσίασή μου, διότι έχουμε περιορισμένο χρόνο, Όπω όλοι γνωρίζουμε. ΣΕΠΑ, δηλαδή ενιαίος χώρο πληρωμών στην Ευρώπη, είναι σημαντική πρωτοβουλία πολιτική που συνεχώ υποστηρίχθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εν γέννη το 2008 οι μεταφορές ΕΠΑ, το σύστημα μεταφοράς ξεκίνησε μαζί με το STT για τις χρεώσεις τον Νοέμβριο του 2009. Όμως, ερώτημα έχω. Μάλλον, ε, ήταν αργός ο ρυθμός εφαρμογής των νέων σχημάτων. Τον Οκτώβριο 2010, δύο χρόνια μετά την εκκίνηση του STT το μερίδιο αυτών των συναλλαγών εναντίον των συναλλαγών μέσω διαφόρων μηχανισμών ήταν μόνο 9,3%. Το μερίδιο το STT ήταν περίπου 1%. Προφανέστατο λοιπόν ότι αυτή ε, η αλλαγή ε, χρειάζεται μετακίνηση προς την νέα νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δύο ψηφίσματά του του Μαρτίου του 2009 και τον Μάρτιο του 2010 ζήτησε και παραθέτω σαφή, ενδεδειγμένη και δεσμευτική προθεσμία τελική που δεν θα πρέπει να είναι μετά τις 31 του 2012 για την ε, μεταφορά στα συστήματα ΣΕΠΑ. Εγώ ανταποκρίθηκα σε αυτό το αίτημα προθώντας ταχεία προθεσμία, διαφορετικά θα ήταν άδικο το σύστημα για αυτούς που άλλαζαν γρήγορα. Το πιο επίμοχο θέμα ποιο είναι τα καταληκτική προθεσμία, μία ή δύο από αυτές, κατ' εξουσιοδότηση πράξης, μυφς, και πληρωμέ σε μεγάλα ποσά. Θα τα αναφέρω αυτά τα θέματα. Αναφερόμενοι σε αυτά τα ζητήματα. Καταληκτικέ προθεσμίες. Προτείνω. Μία να είναι αυτή. Έτσι θα είναι πιο εύκολη η μετανάστευση στο νέο σύστημα και πιο φθηνή. Δύο χρόνια μετά τη θέση ισχύ του κανονισμού έτσι θα υπάρξει χρόνος και για τα κράτη-μέλη εκείνα που η διαδικασία μετακίνηση ήταν πολύ αργή να γίνει μετακίνηση. Μία προθεσμία καταληκτική θα προστεύσει την ενημέρωση του κοινού και να, να γίνουν πιο αποτελεσματικέ εκστατείε ενημέρωση. Τώρα, κατά εξουσιοδότηση πράξη, είναι ενδεδειγμένο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κατά εξουσιοδότηση πράξη για να αλλάξει τεχνικέ προδιαγραφέ. Αλλά μόνο αυτέ. αφαίρεσα διάφορες απαιτήσει από το παράρτημα τον κανονισμό και περίεργα το πεδίο εφαρμογής των κατεξοδότηση πράξεων. Στις κατεξοδότηση πράξεις θα πρέπει να συνομιλεί με το Συμβούλιο ΣΕΠΑ και του ΣΕΠΑ εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτές είναι βασικές απαιτήσει που πήγαν από το παράρτημα προς το κείμενο. Τις μετακίνησα. Αφορούν κυρίως την προστασία των καταναλωτών είναι ρήτρε γι' αυτό. Αφορούν τι άμεσε χρεώσει και απορρέουν από την επιλογή του βασικού μοντέλου. Ότι οι τράπεζε πληρωμών και πιστώσεων έχουν την εντολή και όχι οι τράπεζε των οφειλετών. Λάθος η επιλογή. Έγινε όμω, και πρέπει να αισθανθούν ότι προστατεύονται οι καταναλωτέ όταν πηγαίνουν από την πεδίο εντολή του. αν το πεδίο αυτό τα MIFS. Πολυμερή τέλη συναλλαγών είναι τα αρχικά. Το θέμα των MIFS είναι περίπλοκο. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει το κόστος όσον αφορά τις συναλλαγές. Όταν απορριφθεί, αντιστραφεί, επιστραφεί η πληρωμή. Και εκ των προτέρων καταβολή μυφ ανασυναλλαγή προσπάθησα να βρω συνενετική λύση. Να είναι συνεχή τα μύφια για μεταβατική περίοδο μακρά. Ούτως ώστε μην πληρωμένα μύφ να είναι τα τέλη που καταβάλλονται να είναι ομοιόμορφα στα κράτη-μέλη και να μειώνται σταδιακά. Αν βασίζονται στο κόστος τα μύφ, θα πρέπει να τροποποιηθούν για να είναι τα ίδια στα κράτη-μέλη και να είναι ισότιμη ε, ισότιμοι, για όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στο σύστημα. Εξαιρέσεις. Χρειάζεται μεταβατική περίοδος. Όσο πιο σύντομη γίνεται. Το γερμανικό ELV είναι άμεση πληρωμή που γεννάται από τη χρήση λογαριασμού για τη χορήγηση βασικών πληροφοριών για, την εντολή, για το ένταλμα. Πολλοί καταναλωτές μπορεί να μην γνωρίζουν ότι χρησιμοποιώντα την κάρτα του σε ένα κατάστημα δημιουργούν άμεση ε, άμεσο χρέος, άμεση πληρωμή. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί όσο αφορά το με των πληρωμών μέσω του κανονισμού. Άρα θα μειωθεί το κόστος πληρωμών. Άρα σε τρία χρόνια θα συμμορφωθούν διάφορε πληρωμέ με το σύστημα ΣΕΠΑ ή δε μη θα πρέπει να βρεθεί υποκατάστατο ΣΕΠΑ. Τέλος. Πληρωμές μεγάλες, μεγάλα ποσά. Πληρωμές μεγάλων ποσών. Πρέπει να εξαιρεθούν από τον κανονισμό. Εξ ολοκλήρου. Και να μην υπάρχει κατάχρηση, κακή χρήση αυτού του μέσου. Αυτού του μέτρου μάλλον. Και άλλα θα ήθελα να τονίσω. Αλλά αυτά ήταν τα βασικά. Ευχαριστώ το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του κοιόδη συναδέλφου για την καλή συνεργασία και προσβλέπω σε καρποφόρα, καρποφόρα μελλοντική συνεργασία και ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Θα ακούσω τους φαρόντες ε, συζητητές. Η Σόφη Νετφέλντ για του φιλελεύθερου πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά τη και για το ότι μας ε, ενέπλεξε και μας ευθύς εξ αρχής. Ξανόματος της ομάδας μου. Υποστηρίζω την προσέγγιση που έχει εδώ πέρα όσον αφορά την ενιαία ημερομηνία και τα δύο χρόνια. Μία ημερομηνία οπωσδήποτε. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η ημερομηνία, αλλά πρέπει να είναι ε, το στομότερο δυνατόν. Γιατί προφανώς ναι, αυτό δεν ε, μας ξημέρωσε ξαφνικά σήμερα. Δέκα χρόνια το κοιτάμε. Συμφωνώ επίσης με την προσέγγισή σας ε, να περιοριστούν όσο το δυνατόν ε, οι τεχνικές προδιαγραφές και να μπουν στον κανονισμό και όχι στο παράρτημα. Πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, να μην υπάρχουν τεχνικές απαιτήσει που δεν είναι απολύτως απαραίτητες. Όσον αφορά τα τέλη, τα πολυμερή, Εκεί μπορούμε να έχουμε μόνο κάποια ερωτηματικά για τη μεταβατική περίοδο. Γιατί ούτως ή άλλως θα λήξουν οι ισχύουσες ρυθμίσεις σε κάνα δύο χρόνια και η μεταβατική περίοδος που προτείνεται πηγαίνει πέρα από την ημερομηνία λήξης θα πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ πέρα νομίζω με την Κομισιόν και να το καταργήσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα γιατί προφανώς η ύπαρξη τέτοιων τελών σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ανταγωνισμό και τη δυνατότητα κάποιων να μπουν στην αγορά. Οι παρατηρήσεις σας για το να υπάρξουν ε, κάποιες εξαιρέσεις, ναι, και να είναι όσο δυνατόν πιο σύντομες οι ε, μεταβατικές περίοδοι. Επίσης, δύο παρατηρήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών. Εμένα μου λένε χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο γιατί δεν το ξέρουν οι καταναλωτές. Εγώ θα, θα απαντήσω ε, τι σας εμποδίζει. Αρχίστε να ενημερώνετε τώρα, από τώρα. Μην περιμένετε μέχρι να έρθει η προθεσμία και να περάσει η προθεσμία. Μια φορά ξεχνάμε πως η προθεσμία είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχει γίνει κάτι, όχι ε, εκείνη τη μέρα. Μπορεί να γίνει και από πριν. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι επαναστατικά αυτά που λέω. Και τελευταία παρατήρηση. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το κείμενο για τυχόν εμπόδια σε νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα ε, ή νέους παρόχους που δεν είναι τράπεζες. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε μια αγορά πληρωμών, ένα χώρο πληρωμών που θα προσφέρει όσο δυνατόν περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες ε, και τους παρόχους να μην ε, ενσωματώσουμε εμπόδια που θα κάνουν δύσκολο, θα καταστήσουν δύσκολες κάποιους να μπουν στην αγορά. Το αντίθετο πρέπει να τους διευκολύνουμε. Αλλά νομίζω πως και η συγγήτρια συμφωνεί εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Κύριος Γκίγκολτ, στους πράσινους. Ναι, καταρχήν και από δική μου πλευράς ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές και την, σκιώδη και την εισηγήτρια για τη συνεργασία τους. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα θέμα όπου πολλοί θα προσέξουν προσεκτικά τι γίνεται και τι προτείνεται, τι συμβαίνει. Είναι στο μέσο που οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βρίσκονται πολύ κοντά στους πολίτες και τους αφορούν άμεσα. Ένα πράγμα να πω, τα προβλήματα κάποιων χωρών μελών, επίσης και στη δική μου χώρα, να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση σε μια ενιαία εσωτερική αγορά, να έχουμε έναν ενιαίο χώρο πληρωμών, αυτό ε, έχει ξεπεράσει ήδη το πλαίσιο του εφικτού. Γι' αυτό είναι σωστό να υπάρξει μια καταληκτική ημερομηνία όπου πραγματικά θα καταλήξουμε σε πλήρη αποδοχή, πλήρη ε, ολοκλήρωση. Δεν έχει κανένα νόημα να παρατείνουμε ακόμα περαιτέρω αυτή την καταληκτική ημερομηνία. Δημιουργεί πρόσθετο κόστος ε, και για τα στοιχεία που είναι ξεχωριστά για διαφορετικούς τομείς όλα αυτά δημιουργούν επιπλέον γραφειοκρατική επιβάρυνση που στο τέλος τέλος οι μικροί εμπλεκόμενοι ε, θα πληγούν περισσότερο από τους μεγάλους. Είμαι υπέρ του ότι σε 24 μήνες πρέπει να καταλήξουμε σε μια τελική κατάσταση. Από την άλλη πλευρά τις ανησυχίε πολλών πολιτών πρέπει να τις πάρουμε στα σοβαρά θα έλεγα. Αυτό αφορά και το θέμα το ότι οι πολίτες αναμένουν συνδρομή υποστήριξη στη μετάθεση αυτή και στην εξοικείωση με τα νέα νούμερα, τους νέους αριθμούς. Αυτό με βοήθεια στο διαδίκτυο απλή μορφή μπορεί να γίνει και τα νέα IBANs τραπεζικών κωδικών και τα λοιπά και των ε, πιστοτικών καρτών, ε, των άλλων ε, ειδών καρτών, όλα αυτά να τυπωθούν και πολλές τράπεζες το κάνουν υποδειγματικά αυτό. Δεν κατανοώ γιατί δεν το καταφέρνουν όλοι να το κάνουν τέλεια και υπό το πρίσμα της επικοινωνίας για αυτό το θέμα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα και στα ίσια. Όλες οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να βοηθήσουν τους πελάτες τους σε αυτή την μετάθεση και να τους συνδράμουν. Αυτό το οποίο δεν γίνεται είναι μετά τον εξευρωπαϊσμό, μετά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που θα θέλουμε να πετύχουμε, οι τιμέ να ανέβουν, να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, τα τέλη και οι τιμέ. Ξέρουμε ότι δεν λειτουργούν τέλεια οι αγορέ. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε στου πολίτε μα ότι για τι συναλλαγέ αυτέ το κόστος συναλλαγών μετά τη μεταρρύθμιση δεν θα είναι υψηλότερο από ό,τι πριν από τη μεταρρύθμιση. Αυτό δεν είναι ε, κατάχρηση παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά όταν διασφαλίζουμε ότι σε αυτόν τον τομέα με εξευρωπαϊσμό θα καταλήξουμε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τότε σε αυτόν τον τομέα δεν θα πρέπει οι τιμές να αυξηθούν περαιτέρω μετά τον εξευρωπαϊσμό. Μία άλλη υπόθεση είναι ο επιμερισμός των τελών και δαπανών. Έχουμε ένα ε, αποτελεσματικό σύστημα με την ηλεκτρονική λειτουργία. Αυτό το σύστημα θέλουν τουλάχιστον στη Γερμανία οι πολίτες να το διατηρήσουν. Έχουμε και παρόμοια άλλα συστήματα. Πρέπει όμως να καταλήξουμε σε επίλυση του προβλήματος. Λύση που θα υιοθετεί τις εξής προϋποθέσεις. Συναλλαγές ε, σε σχέση με την οικονομία πρέπει να είναι το δυνατόν χαμηλότερες. Πρέπει να διασφαλίζονται τα εμβάσματα αλλά σε προσιτές ε, τιμές. Αυτό που δεν είναι αποδεκτό είναι στη συνέχεια να έχουμε ένα πρότυπο που θα επιβαρύνει το εμπόριο και τους πελάτες και τους μικρομεσαίους με υψηλότερα τέλη συναλλαγών από ό,τι γίνεται σήμερα. Από ότι ε, επιβάλλονται σήμερα. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Το γερμανικό πρότυπο με την ηλεκτρονική επιβάρυνση, η ηλεκτρονική ε, ίσπραξη τελών μπορεί να λειτουργήσει ίσως. Αναμένω μια λύση που θα είναι τουλάχιστον εξίσου καλή όπως αυτή που έχουμε εμεί ήδη σήμερα στη διάθεσή μας. Ένα τέτοιο σύστημα που θα εξευρωπαϊστεί, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο όπως το γερμανικό αυτό το εξευρωπαϊσμένο σύστημα, αλλά πρέπει να έχει τα ίδια πλεονεκτήματα για τους πολίτες μας. Ένα άλλο σημείο το οποίο θεωρώ σημαντικό για την, ε, ε, ε, τον συμψηφισμό, τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ανάκλησης πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα ανάκλησης ή παναχώρησης. Όταν γίνεται κάποιος λογαριασμός ο οποίος οδηγεί σε αφαίρεση ποσών από τον λογαριασμό πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα ε, συμφωνεί πάντα ο πελάτης και ότι θα μπορεί να διατυπώσει ενστάσεις. Ε, αυτές οι αφαιρέσεις, οι, ας το πω έτσι, ε, αντλήσεις ποσών ε, οδηγούν πολλές φορές στο να έχουμε την παρέμβαση από πλευράς πελάτη. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης διότι έτσι τα τέλη θα μπορούν με πιο δημοκρατικό τρόπο να επιμερίζονται. Έχω και ένα άλλο ερώτημα το οποίο θέλω να δούμε. Ο τρόπος με τον οποίο στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα ρυθμίζουμε τα πράγματα στην Ευρώπη. Ένα δημοκρατικά αμφισβητήσιμο πλαίσιο. Δεν είναι δυνατόν το European Payment την ε, βιομηχανία να την οδηγεί σε αυτορύθμιση. Οι υπέρμαχοι της προστασίας ε, των καταναλωτών να βρίσκονται με άλλους σε ένα διοικητικό συμβούλιο αλλά στο τέλος να αποφασίζουν οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες ε, τις αποφάσεις αυτές. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο εκδημοκρατισμός αυτού του πλαισίου. Φυσικά οι αρμόδιοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να έχουν λόγο να αρθρώσουν. Φυσικά οι πιο υπεύθυνοι θα πρέπει να μπορούν να δράσουν από πλευρά του τους. Όμως θα πρέπει αυτές οι συναλλαγές δημοκρατικά να διαμορφώνονται και όχι με έναν τρόπο αυτορυθμίσεων που από πλευρά ε, εκείνων που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες θα ρυθμίζονται τα πράγματα αφ' αυτών σε ένα στεγανό πλαίσιο. Αυτό δεν είναι δημοκρατική ρύθμιση. Θα πρέπει να υπάρχουν δημοκρατικές δυνατότητες συνδιαμόρφωσης. Θα ευχόμουν από πλευράς εισήγηση ε, και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υψώσουμε τα λάβαρα της δημοκρατικής διαμόρφωσης των πραγμάτων ώστε σε αυτές τις συναλλαγές με δημοκρατικό τρόπο να διαμορφώνονται τα πράγματα φυσικά με εμπλοκή και συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αλλά δεν βλέπω γιατί σε αυτόν τον τομέα δεν θα μπορούσαμε μέσω εντεταλμένων ε, ε, πράξεων ή ε, πράξεων που θα εκτελούνται με εντολή δεν θα πρέπει να αρνηθούμε μια τέτοια προοπτική. Αν δώσουμε την δυνατότητα να διασφαλίζονται έτσι τα δικαιώματα των πολιτών, θα είμαστε υπέρ της δημοκρατικής διαμόρφωσης πραγμάτων. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα δεκάλεπτο. Έχουμε τον κύριο, τους δύο ομιλητές επόμενους, θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητή μετά. Λοιπόν, παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι στα σχόλιά σας, διότι θα φύγουν οι δερμοί σε 10 λεπτά. Ο κύριο Χουντής έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη σοβαρή δουλειά που έχει κάνει. Μπαίνω κατευθείαν στις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και δεν το αντιμετωπίζει και η εισηγήτρια ως ένα τεχνικό ζήτημα απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, είναι και τέτοιο και χρειάζονται να γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις για να πάμε στον ενιαίο χώρο, αλλά και από τη συζήτηση φαίνεται, και εγώ θα επιμείνω σε δύο-τρεις πλευρές τέτοιες, ε, ότι έχει και οικονομικές και κοινωνικές πλευρές. Νομίζω ότι το βασικό μας μέλημα θα πρέπει να είναι η προστασία του πολίτη και του καταναλωτή. Αυτό σημαίνει αξιοπιστία των υπηρεσιών και βεβαίως ότι δεν θα αυξηθεί το κόστος. Πιο συγκεκριμένα ε, θα πρέπει να προασπίσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, τα συμφέροντα των πελατών και ότι αυτό το κόστος αυτής της μετάβασης δεν θα το μετακυλήσουν στους πολίτες και στους καταναλωτές διαμορφώνοντας ένα ακριβότερο σύστημα πληρωμών. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αυτές οι αδιαφανείς και ιδιαίτερα ψηλές διατραπεζικές προμήθειες πρέπει να καταργηθούν αφού πάμε σε ενίο χώρο. Και επομένως προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Η δεύτερη παρατήρηση είναι πρέπει να προστατεύσουμε και να διασφαλίζονται οι καταναλωτές από τον κίνδυνο της απάτης. Οι έρευνες λένε ότι τα ποσοστά είναι ψηλά και τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης είναι χιλιάδες. Με αυτή την έννοια, το σύστημα που επιλέγεται από την Επιτροπή, CMF, δεν ξέρω αν είναι το καταλληλότερο. Το επισήμανε, αν πρόσεξα καλά, και στην προφορική της ε, παρουσίαση η συγγήτρια, διότι τον έλεγχο όλη αυτή τη υπόθεση δεν τον έχει η τράπεζα του καταναλωτή, την έχει η τράπεζα του δικαιούχου. Έτσι δεν είναι. Και εκεί μπορεί να εμφανιστούν εικονικά ποσά, τα οποία να μην μπορεί να τα ελέξει ο καταναλωτή ή η τράπεζά του. Επομένω, δεν ξέρω αν το σύστημα αυτό που επιλέγεται είναι το καταλληλότερο. Τρίτη πλευρά τονίστηκε και από άλλους ε, ομιλητέ δεν θέλω να επιμείνω περισσότερο, το θέμα τη ενημέρωση είναι σοβαρό και δεν είναι και απλό υπογραμμίζω τμήματα της κοινωνίας, αλλού μεγαλύτερα, αλλού περισσότερα, όπως οι ηλικιωμένοι ή οι μη εξοικειωμένοι στο διαδίκτυο, που πρέπει να ενημερωθούν ή που πρέπει να βοηθηθούν καταλήλως για να μπορούν να μιλάμε για ενίο χώρο, να μπορούν να χειριστούν αυτό το και δεν είναι λίγοι και επομένως πρέπει να το πάρουμε υπόψη. Τέταρτη και τελευταία παρατήρηση και τελείωσα κυρία Πρόεδρος, είναι σχετικά με το χρόνο. Συμφωνώ και εγώ πρέπει να μπει ένα χρόνο μια καταληκτική ημερομηνία ενιαίως. Αλλά να πάρουμε υπόψη ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην προσαρμογή από χώρα σε χώρα. Πρέπει να χρειαστούν να γίνουν και άλλες κινήσεις και είμαστε σε διαφορετικές ταχύτητες. Επομένως θα υποστηρίξω μια ημερομηνία και νομίζω ότι η συγγήτρια πρέπει να το λάβει υπόψη που θα έχει πάρει υπόψη της όλες τις προϋποθέσεις προσαρμογής για να πάμε πράγματι σύντομα σε έναν ενιαίο χώρο πληρωμών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε δεν θέλω τίποτα. Με τις τροπολογίες και τη συνέχεια θα κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Padar, if you could also be brief, I appreciate it. Thank you. Αν είναι σύντομος παρακαλώ. First. Πολύ σύντομος θα είμαι. Καταρχάς, ευχαριστώ την εισηγήτρια που ε, προσπάθησε να πει τα σωστά σημεία από την αρχή. Δεν χρειάζεται δικαιολόγηση ο κανονισμός. Εξυπηρετεί σκοπό ολοκλήρωση μια αγοράς. Υποστηρίζω την εισηγήτρια που υπέβαλε μία ημερομηνία. Η ενδήποτε εξαίρεψη πρέπει να είναι σύντομη και τεκμηριωμένη. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην εισηγήτρια το λόγο. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 16 Μαΐου. Θα έχετε δυνατότητα για συζήτηση των τροπολογιών μετά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στις 14 Ιουνίου. Λοιπόν, η συγγήτρια να ανακεφαλαιώσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμφωνούμε όλοι για ένα γρήγορο χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ο κανονισμός αφορά μια καταληκτική ημερομηνία. Και ε, να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Συμφωνώ με την ε, Σόφη Νετφέλτ και τον κύριο Χουντή πως χρειάζεται μια εκστρατεία ενημέρωσης για τους καταναλωτές και το κοινό έτσι ώστε η μετάβαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ήπια και τέλος επίσης όλοι οι σκιώδεις ηγητές ανέφεραν το θέμα των ρητρών προστασίας των καταναλωτών και του πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ρήτρες, πόσο ουσιώδη ρόλο έχουν. Νομίζω μπορούμε να τις δούμε μαζί για να διατυπωθούν ε, σωστά και να έχουμε έτσι την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση των ε, πελατών. Γιατί εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι, γιατί χωρίς ε, να το δεχτεί το κοινό δεν μπορούμε να περάσουμε στην την νομοθεσία. Αυτά νομίζω ήταν τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν για το ELV δεν ξέρω αν υπήρχε ερώτηση ή σχόλιο. Κύριε Κίγκολτ. Ένα σχόλιο. Α, αν θέλετε δείτε το ως ερώτηση. Ποιο, ποιο ήταν κιόλα. Γιατί άκουγα τη διερμηνία από τα γερμανικά στα φιλανδικά και δεν ξέρω τι ήταν διατύπωση. We ή μπορούμε να το δούμε μεταξύ των ε, ε, σκιωδών εισηγητών, αλλά το βασικό για μένα ήταν να φροντίσουμε πως αυτό το οποίο θα έχουμε τελικά θα έχει την ίδια ποιότητα με αυτό το οποίο έχουμε. Δηλαδή περισσότερη Ευρώπη να σημαίνει φθηνότερε ε, λύσεις και υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Αυτό νομίζω μπορούμε να το επιτύχουμε. Αλλά κανείς δεν θα δεχτεί να χάσουμε ένα φτηνό και αποτελεσματικό σύστημα για να έχουμε μετά ψηλότερες τιμές και ψηλότερο, ψηλότερο κόστος συναλλαγής από αυτό το οποίο έχουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι μικρότερο κόστος συναλλαγής σε ένα κοινό σύστημα που θα λειτουργήσει ολόκληρη την Ευρώπη για να συμπληρώσει την εσωτερική αγορά. Και εκεί πέρα δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε ε, συνένεση. Κοιτάξτε, η πρόεδρος, <laughs> δεν έχουμε χρόνο για τη συζήτηση. Νομίζω πω θα τα δείτε αυτά στι τροπολογίε. Ναι, ναι, πράγματι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμό και θα μειωθεί το κόστος με αυτόν τον κανονισμό για του πελάτες. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν απομένει παρά να σα ευχηθώ καλό Πάσχα και να σα υπενθυμίσω 22 Μαου 3 η ώρα το απόγευμα, επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ στην Άλφη για τη συνεργασία σα και που με βοηθήσατε.